Καλημέρα συνάδελφοι. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση που είχε διακοπεί στις 11 Δεκεμβρίου. Τα πρακτικά και τα εγκεκριμένα κείμενα της 11ης Δεκεμβρίου σας έχουν μοιραστεί. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Δεν βλέπω. Οπότε εγκρίνονται. κάποιε ανακοινώσει. Κατόπιν εκλογής ε, του κυρίου Άλιν Σμιθ ε, στην Βουλή του Ηνωμένου Βασιλείου, το Ηνωμένο Βασιλείο σημειώνει ότι σύμφωνα με την ε, σχετική νομοθεσία που αφορά τις ευρωεκλογές, το αξίωμα αυτό είναι ασύμβατο με το αξίωμα του Ευρωβουλευτή και επιβεβαιώνει ότι χειρεύει η από 13 Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τον κανονισμό. Η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών μου ανακοίνωσε κάποιες αποφάσεις που αφορούν αλλαγές στους διορισμούς σε Επιτροπή Αντιπροσωπεία. Οι αποφάσεις αυτές θα περιληφθούν στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης και τίθενται ενισχύ αμέσως. Οι Επιτροπές ΕΝΒ και μας έστειλαν τρία διορθωτικά σε κείμενα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με το άρθρο 241 παράγραφο 4 του κανονισμού θεωρούνται εγκεκριμένες εκτός εάν εντό 24 ωρών μια πολιτική ομάδα ή αριθμός βουλευτών ο ελάχιστος αριθμός βουλευτών έχει κάποια αντίρρηση. Υπάρχουν αυτά διαθέσιμα στο site της Ολομέλειας και θα δημοσιευτούν στα πρακτικά της τρέχουσας συνεδρίασης οι επιτροπές Ήτρα και Τραν αποφάσισαν να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις ε, στην πρώτη ανάγνωση με το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 72 του κανονισμού μας. Η θέση που έχει εγκρίνει το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας και ο τίτλος της θα δημοσιευτεί στα πρακτικά αυτής συνεδρίασης η διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών με ενημέρωσε ότι δεν έλαβε καμία αντίρρηση για την σύσταση της Επιτροπής ΕΚΟΝ για να μην υπάρξει αντίρρηση σε μια εκτελεστική πράξη σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφο 4 του κανονισμού. Η σύσταση αυτή είναι διαθέσιμη στην σελίδα τη Ολομέλεια. Εάν εντό 24 ωρών καμία πολιτική ομάδα ή ο ελάχιστο αριθμό βουλευτών δεν φέρει αντίρρηση, η σύσταση αυτή θεωρείται εγκεκριμένη. Στην αντίθετη περίπτωση θα τεθεί σε ψηφοφορία. Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 2 του κανονισμού έχω λάβει από την Επιτροπή Απασχόλησης ένα αίτημα για διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για τον αξιοπρεπή ελάχιστο μισθό στην Ευρώπη. Εάν εντό 24 ώρων δεν υπάρξει αντίρρηση από πολιτική ομάδα των ελάχιστων αριθμών βουλευτών, εγκρίνεται σε αντίθετη περίπτωση θα τεθεί σε ψηφοφορία. Οι υπογραφέ νομοθετικών πράξεων που εγκρίθηκαν με την τακτική νομοθετική διαδικασία θέλω να ενημερώσω ότι η αίθουσα πω την Τετάρτη θα υπογράψω σύμφωνα με το άρθρο του 79 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου τρία νομοθετήματα που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο τη τακτική νομοθετική διαδικασία. Οι τίτλοι του ε, θα δημοσιευτούν στα πρακτικά τη σημερινή συνεδρίαση. Και τώρα περνάμε στην ημερήσια διάταξη. Έχετε την ημερήσια διάταξη που εγκρίθηκε στις 11 Δεκεμβρίου και η οποία σας έχει ήδη μοιραστεί. Ας δούμε τώρα κάποια αιτήματα που υπάρχουν για αλλαγές. Σύμφωνα με τις διαβουλεύσεις με τις πολιτικές ομάδες, θα ήθελα να προτείνω τις εξής αλλαγές ε, στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης στην Ολομέλεια όσον αφορά την Πέμπτη η ψηφοφορία για την δήλωση της Κομισιόν για το κράτος δικαίου στην Μάλτα μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις ε, που αφορούν τη δολοφονία της Δάφνης Γαρουάνα Γαλίτσια πάει στην Τετάρτη. Συνεπώς, οι προθεσμίες αλλάζουν ως εξή. Προτάσει για ψηφίσματα Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου, 7 η ώρα το απόγευμα. Τροπολογίες ε, σε αυτά και προτάσεις κοινών ψηφισμάτων, Τρίτη 17 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι τροπολογίες ε, στα κοινά ψηφίσματα 17 Δεκεμβρίου, 1 η ώρα το μεσημέρι. Χωριστές ε, ψηφοφορίες 3η ε, 17 Δεκεμβρίου, 7 η ώρα το απόγευμα. Υπάρχουν αντιρρήσεις? Όχι. Ωραία, εγκρίνεται. Όσον αφορά την Τρίτη, η ομάδα των Πρασίνων ζήτησε η συζήτηση για τη δήλωση Κομισιόν για την στρατηγική της Ένωσης για την αναπηρία μετά το 2020 να ολοκληρωθεί με ψήφισμα, το οποίο θα ψηφιστεί σε μια επόμενη συνεδρίαση. τον, δίνω τον λόγο, με συγχωρείτε, στην κυρία Κάτριν Λάγκενζίπεν για να παρουσιάσει την θέση της ομάδας των Πρασίνων. Έχετε τον λόγο. Καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε. Αύριο θα συζητήσουμε στην Ολομέλεια για την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα άτομα με αναπηρίες μετά το 2020. Θα ήθελα να προτείνω να υπάρξει ένα σχέδιο ψηφίσματος το οποίο θα ψηφιστεί τον Φεβρουάριο. λόγος είναι ότι η τρέχουσα στρατηγική για την αναπηρία εκπνέει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει ακόμα συνεισφέρει τίποτα για την μελλοντική στρατηγική. Επειδή λοιπόν οι άνθρωποι με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να υφίστανται διάφορε διακρίσει, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής ενωση να είναι πιο φιλόδοξη και χωρίς αποκλεισμού. Γι' αυτό θα θέλαμε η συνεισφορά μας να είναι υπομορφή ενός ψηφίσματος το οποίο θα απευθύνεται προς την Κομισιόν πριν προταθεί η νέα αυτή στρατηγική. Θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι αναπηρία στην Ευρώπη βασίζονται στην στήριξή μας. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω αγαπητοί συνάδελφοι να στηρίξετε το ψήφισμα αυτό το οποίο θα ψηφιστεί τον Φεβρουάριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Λάγκεντζίπεν, δίνω τον λόγο. Για ε, όποιον θέλει να μιλήσει κατά το αιτήματο, ε, θέλει κάποιος, όχι. Οπότε, τίθεται σε ψηφοφορία το αίτημα. Ποιο συμφωνεί με την πρόταση της κυρίας Λάγκεν Ζήπεν. Σηκώστε το χέρι. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οπότε, η συζήτηση για τη δήλωση της Κομισιόν για τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναπηρία. Μετά το 2020 θα ολοκληρωθεί με ψήφισμα το οποίο θα ψηφιστεί σε μια επόμενη ολομέλεια. Όσον αφορά την τρίτη, οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες ζήτησαν η δήλωση του Συμβουλίου και της Κομισιόν για τα αποτελέσματα τη COP25 να προσθεθούν το πρωί ως δεύτερο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Δίνω λόγο στην κυρία Μποναφέ. Σας ευχαριστώ. Χτες ε, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ε, της COP25 ε, με ελάχιστα θετικά αποτελέσματα από την πλευρά των χωρών και βεβαίως νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για έλλειμμα όσον αφορά τις πρωτοβουλίες και τις πράξεις για να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή. Λοιπόν, οι συνάδελφοι θα θυμάστε ότι την προηγούμενη Τετάρτη είχαμε μια έκτακτη σύνοδο Ολομέλειας για τον Green New Deal ακριβώς για αυτά τα θέματα και ψηφίσαμε στην προηγούμενη Ολομέλεια του Στρασβούργου ακριβώς ε, ένα ψήφισμα για την επίγουσα κλιματική αλλαγή. Γι' αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα αυτό για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μποναφέ. Ε, κάποιος κατά του αιτήματο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με το γεγονό ότι όντω θα πρέπει να γίνει η συζήτηση για τη διάσκεψη των μερών στη Μαδρίτη, η οποία ήταν πολύ απογοτευτική πράγματι. Όμω να προσθεθεί στην Τρίτη πρωί, την Τρίτη πρωί αγαπητοί φίλοι σοσιαλιστές. Αυτό το κάνετε για να αντιστρέψετε την προσοχή από την κατάσταση στη Μάλτα. Για να μπορέσουμε να συζητήσουμε τα τεκτενόμενα στη Μάλτα χρειαζόμαστε αρκετό χρόνο και δεν θα πρέπει να βιαζόμαστε. Συμφωνώ λοιπόν με την πρόθεση, προτείνω όμως το Προεδρείο ε, η συζήτηση αυτή να μπει την Τρίτη το απόγευμα για παράδειγμα και όχι την Τρίτη πρωί. Εμάς τρίτη το απόγευμα μας βολεύει και θα έχετε την ολόθερμη στήριξή μας. Αλλά αφήστε μας να μπορέσουμε να συζητήσουμε με το χρόνο που χρειάζεται την κατάσταση στη Μάλτα. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, σαφέστατο. Δεν είναι αντίθετη η συνάδελφος, αλλά ας σας ακούσουμε κυρία Μποναφέ. Κοιτάξτε, εδώ πέρα το ΕΛΚ ε, κάνει λάθος. Εμείς ε, ζητήσαμε να γίνει αυτή η συζήτηση τρίτη πρωί, γιατί τρίτη πρωί υπάρχει αρκετός χρόνος να συζητηθεί. Τρίτη απόγευμα έχουμε πάρα πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη, αλλά για μας δεν είναι πρόβλημα. Δεν, το δεχόμαστε, δεχόμαστε και το απόγευμα. Το βασικό είναι να συζητήσουμε τα αποτελέσματα αυτής της αποτυχημένης συνόδου. Οπότε, αν, ναι. αν συμφωνείτε να το θέσουμε σε ψηφοφορία, να συζητηθεί την Τρίτη το απόγευμα. Ποιος συμφωνεί λοιπόν. Αυτή η συζήτηση να λάβει χώρα την Τρίτη το απόγευμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δήλωση Συμβουλίου και Επιτροπής λοιπόν για τα αποτελέσματα της ΚΟΠΑ θα προσθεθεί την Τρίτη το απόγευμα. Λοιπόν. Τετάρτη. Η ομάδα ECR ζήτησε να υπάρξει μια δήλωση διτίου είπα του εκπροσώπου για την βίαιη καταστολή των πρόσφατων διαμαρτυριών στο Ιράν το απόγευμα ως πέμπτο σημείο. Και θα ολοκληρωθεί με ένα ψήφισμα το οποίο θα ψηφιστεί την πέμπτη. Τον λόγο έχει η κυρία Φωτίγκα για να παρουσιάσει το αίτημα. Σας παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφοι, θα ήθελα να ζητήσω τη συγκατάθεσή σας να προσθεθεί το σημείο αυτό στην ημερησία μας διάταξη. Γνωρίζω ότι είναι μια ιδιαίτερη περίοδος αυτή, διότι τα Χριστούγεννα πλησιάζουν. Δυστυχώς όμως, ήδη γνωρίζουμε, όλοι γνωρίζουμε, ότι περίπου ήδη 1500 άνθρωποι έχουν βρει το θάνατο στο Ιράν, λόγω του πρόσφατου κύματος καταστολής και παρά τις δυσκολίες που βιώνουν, τα μέλη της αντιπολίτευσης, οι διαδηλωτέ και οι ανήλικοι μάλιστα, προσπαθούν με επιμελή τρόπο να βρουν τα ονόματα όλων αυτών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων και των διαμαρτυριών, έτσι ώστε να μην ξεχαστούν. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ, είναι πολύ κρίσιμη αυτή η χρονική συγκυρία να ενώσουμε και εμείς τις φωνές μας με τις δικές τους. Διότι είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για πολλούς από τους ανθρώπους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε συνθήκες κράτησης και βιώνουν συνθήκες ανασφάλειας. Ζητώ λοιπόν τη συγκατάθεσή σας για την προσθήκη αυτού του σημείου στην ημερήσια διάταξη. Σας ευχαριστώ κύριε Φωτίγκα. Δίνω τον λόγο ε, σε όποιον θέλει να μιλήσει κατά του αιτήματος. Αν υπάρχει, Μποναφέ. Παρακαλώ κύριε Μποναφέ. Ευχαριστώ. Μα ε, στην πραγματικότητα δεν ε, είμαστε εναντίον. Έχω μια πρόταση γιατί και η δική μας η ομάδα βεβαίω καταδικάζει στεναρά την καταστολή των διαδηλωτών. Προτείνουμε όμως να γίνει μια συζήτηση με ψήφισμα στην επόμενη Ολομέλεια του Ιανουαρίου γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να γίνει μια συζήτηση γενικά για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιράν που αφορά και θέματα που σχετίζονται με την πυρηνική συμφωνία και την καταστολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικώ. Κυρία Φωτίγκα, συμφωνείτε με αυτό το οποίο προτείνει η κυρία Μποναφέ να αναβληθεί συζήτηση και ψήφισμα για τον Ιανουάριο. Κοιτάξτε, προσωπικά διότι έχω προσωπικά βιώματα ε, της ε, μακροχρόνιας διαμαρτυρίας εναντίον του κομμουνισμού. Ξέρω πόσο στοιχίζει αυτό, πόσο κάθε στιγμή που μετράει, κάθε στιγμή που περνάει είναι πολύ σημαντική για τα θύματα. Βεβαίως στάσομαι με την πλειοψηφία. Εγώ δεν θα ήθελα, αλλά αν η πλειοψηφία αποφασίσει ότι είναι καλό να μετατεθεί η συζήτηση χρονικά για τον Ιανουάριο, έστω. Όμως, θα ήθελα τουλάχιστον, εάν εγκριθεί για τον Ιανουάριο τελικά, να εκδώσουμε μια δήλωση. Είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί η φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε θα ε, ψηφίσουμε διανατάσεις χειρός. είναι υπέρ της πρότασης της κυρίας Φωτίγκας. Κώστε το χέρι. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οπότε... Ορίστε. Θέλετε να το επαληθεύσουμε. Μα εμένα μου φάνηκε σαφές. Καλώς. Να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Οπότε, η δήλωση του Αντιπροέδρου είπα του εκπροσώπου για την η καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν προστίθεται το απόγευμα ως πέμπτο σημείο. Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί με ψήφισμα το οποίο θα ψηφιστεί την πέμπτη προσημείες, είναι η εξής προτάσεις ε, ψηφίσματος 3 17 Δεκεμβρίου 12 η ώρα, τροπολογίες στις προτάσεις αυτές ε, ή κοινά ψηφίσματα 4 18 Δεκεμβρίου 12 η ώρα, τροπολογίες στις προτάσεις κοινών ψηφισμάτων ψηφισμάτων στις 1 η ώρα, χωριστές ε, ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματα Τετάρτη 18 του 7 η ώρα το απόγευμα. Ωραία. Και τελειώσαμε με αυτό το κομμάτι. Φεστ, ζητήσατε τον λόγο. Ναι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω έναν βουλευτό εδώ πέρα. Αγαπητέ κύριε Φαράτζ, είστε ο πατέρας του Brexit και έτσι δείξατε ότι ακόμα και ένα αντιδημοκρατικό θεσμικό όργανο όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μεταρρυθμιστεί. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητέ κύριε Φαράτζ. Νομίζω ότι οποιοδήποτε θέλει να μιλήσει αρκεί να το ζητήσει. Αλλά δεν μπορεί να ζητάτε το λόγο επί διαδικαστικού και να ξεκινάτε μετά συζήτηση όμως. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, άρα έχει εγκριθεί η ημερήσια διάταξη. Και τώρα να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει ιδιαίτερο ζήλος για αυτές τις ε, παρεμβάσεις μόνο όταν προέρχονται από εδώ. Πολλές φορές ακούμε συναδέλφους να εκτροχιάζουν μια συζήτηση ή να παρεμβαίνουν σε άσχετο θέμα. Απλά να ζητήσω λίγη ισορροπία να υπάρχει. Κύριε Τσάνη. Σας υπενθυμίζω πως διάφοροι βουλευτές από διάφορες ομάδες ε, έχουν ε, υποστεί επίπληξη. Δεν ζητάμε τον λόγο επί του διαδικαστικού για να μιλάμε για άλλα ζητήματα. Ευχαριστώ. Dear Θέμα της σημερινής διάταξη. Δήλωση της Κομισιόν περί του εορτασμού της 30ης επαιτίου της Ρουμανικής Επανάστασης του Δεκεμβρίου 1989. Δήλωση της Επιτροπής. Σας υπενθυμίζω ότι έχετε το δικαίωμα να μιλήσετε κατά τη διάρκεια του Catch καθώς και να καταθέσετε μπλε κάρτες. Οι σχετικέ ε, οδηγίες ε, βρίσκονται στην είσοδο της αίθουσα. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ. Η συνεδρία συνεχίζεται με συζήτηση. Να δώσω τον λόγο στην Επίτροπο Βαλέαν. Παρακαλώ, κυρία Επίτροπε. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. κυρίες και κύριοι βουλευτές. Έχω την τιμή να γύρω ενώπιόν σας για να ρωτάσουμε μαζί αυτή τη σημαντική επέτειο για τη Ρουμανία και την Ευρώπη γενικότερα. Revoluția română a început la Timișoara. Acesta a fost primul pas spre reîntoarcerea României și a românilor în Europa. Την εποχή εκείνη συνέβησαν ε, γεγονότα τα οποία άλλαξαν άρδιν την κατάσταση στην Ρουμανία. Η Ρουμανική Επανάσταση ήταν το τελευταίο βήμα, η τελευταία εξέλιξη μετά από τις εξεγέρσεις κατά του κομμουνισμού έχασαν τη ζωή τους χίλιοι άνθρωποι κατά τη διάρκεια αιματηρών ταραχών που έγιναν για την ελευθερία τα θεμελιώδη δικαιώματα, το δίκαιο και η δημοκρατία. Αυτές οι αξίες είναι το θεμέλιο της Ευρώπης μας όπως την γνωρίζουμε σήμερα πέρα από τις διαφορές γλώσσες φυλής ή παραδόσεων. Οπότε είμαστε ενωμένοι σε Βορρά, Νότο, Ανατολή και Δύση για να προωθήσουμε αυτές τις αξίες, τα θεμελιώδη δικαιώματα και θα πρέπει ακριβώς να συνεχίσουν να αποτελούν κινητήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κομμουνιστικό καθεστώς προσπάθησε να καταστήλει τις επιθυμίες των Ρουμάνων για ελευθερία και δημοκρατία. Και βεβαίως οι δυσκολίες της μεταβατικής περίοδου μοιάζουν σήμερα να απέχουν έτη φωτός από την ε, Ρουμανία την σημερινή η οποία βεβαίω ε, είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ ήμουν 20 χρονών τότε στο Πανεπιστήμιο και θα θυμάμαι για πάντα μέσα μου αλλά είναι και κάτι το οποίο θα παραμείνει στη συλλογική μνήμη του ρουμανικού λαού αυτή η μετάβαση προς την ε, δημοκρατία μετάβαση η οποία κορυφώθηκε με την ένταξη της χώρας μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε ότι βεβαίω τίποτα δεν είναι μόνιμο. Πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν κανείς να μην ξαναζήσει σε τέτοια καθεστώτα υπ' αυτές συνθήκες και με απομόνωση. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να τήρουμε πάντα αυτές τις αρχές, ειδικά και σε σχέση με τις χώρες της ε, γειτονιάς μας. Υπάρχει πολλής δρόμος ε, ακόμα για την ε, πλήρη σύγκλησή μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και παρακολουθούμε πάντα την κατάσταση του κράτους δικαίου αλλά η Ρουμανία έχει πολλούς πόρους στην διάθεσή της είναι μια χώρα η οποία αναπτύσσεται, υπάρχουν νέες δεξιότητες, υπάρχει η ψηφιακή οικονομία και είμαι σίγουρη πως θα συνεχίσουμε έτσι τα επόμενα χρόνια. Το Green Deal ε, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα σημαίνει ότι θα έχουμε νέες φιλοδοξίες. Η καθημερινή ζωή πρέπει να προσφέρει ευκαιρίες σε όλους, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Ρουμανία η αποδοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 72%, υψηλότερη από ποτέ. Οι περισσότεροι Ρουμάνοι κατανοούν ότι έχουν ωφεληθεί από τη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό αποτυπώθηκε και στις τελευταίες ευρωεκλογές. Ο μεσόρος προσέλευσης ήταν υψηλότερος από το μεσόρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μέρες του 89 είναι μέρες αξέχαστες. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει καλύτερος τόπος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εορτάσουμε την επέτειο αυτή. Την επάνωδο δηλαδή της Ρουμανίας στην καρδιά της ευρωπαϊκής οικογένειας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Εκ μέρους των πολιτικών ομάδων, δύο λεπτά. Ο κύριος Μπασέσκου πρώτα από το ΕΛΚ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους της πολιτικής μου ομάδας αλλά και τις άλλες πολιτικές ομάδες για το ότι συζητάμε το θέμα σήμερα. Είμαστε στον, στο σπίτι της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Έχουν περάσει ήδη 30 χρόνια από τότε, από το 1989 τότε που όλα ξεκίνησαν με κοινωνική αναταραχή που οδήγησε σε ιστορικές εξελίξεις. Στις 17 Δεκεμβρίου του 1989 ο στρατός πυροβόλησε κατά διαδηλωτών στο Βουκουρέστι, στην Τιμισοάρα και αλλού. Εκατομμύρια Ρουμάνων βγήκαν στους δρόμους. Πρόκειται για βίαιη καταστολή από ένα βίαιο καθεστώς. Τα γεγονότα εν τέλει κόστησαν τη ζωή σε 800 Ρουμάνους, 3.000 τραυματίες. Παρά τους αριθμούς αυτούς όμως, παρά τα θύματα, η Ρουμανία επέστρεψε στην καρδιά της ευρωπαϊκής οικογένειας. Σε μια κοινότητα αξιών από την οποία είχε βία αποσπαστεί Εξαιτήσει ενός καθεστώτος καταστολής. Οι Ρουμανοί είπαν όχι. Οι Ρουμανοί είπαν ότι θέλουμε να κάνουμε τη ζωή μας, θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας τον κομμουνισμό και έτσι έγιναν εν τέλει και πάλι για άλλη μια φορά μέλη της Ευρωπαϊκής Οικογένειας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα εγχείρημα μόνο υπέρ της ειρήνης. Είναι μια φωνή κατά της καταστολής και της καταπίεσης. Εκ μέρους των ε, σοσιαλιστών για 1,5 λεπτό, κύριε Στεράχης. Κύριε Πρόεδρε, η παράσταση του Δεκεμβρίου του 1989 σήμαινε το τέλος ενός βίαιου καθεστώτος καταστολής στην Ρουμανία. Σε διαστολή με άλλα κομμουνιστικά καθεστώτα, πέρασαμε μια αιματοχυσία. Εκατοντάδες ήταν τα θύματα. Πληρώσαμε λοιπόν βαρύ φόρο αίματος για να απαλλαγούμε από μια δικτατορία. Εκατοντάδες χιλιάδες Ρουμάνοι από κάθε γωνιά της Ρουμανίας είχαν υποφέρει από το 1946 μέχρι τότε. Δεν είχαμε ελευθερία, δεν είχαμε σεβασμό για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Δώσαμε μακρόχρονο αγώνα, οι παρτιζάνοι στα βουνά και βρεθήκαμε μετά στις φυλακές όπου πολλοί έχασαν την ζωή τους. Κάποιοι εκτελέστηκαν προσπαθώντας να διασχίσουν τα σύνορα προς τη Δύση. Η Ρουμανία είχε γίνει μια μεγάλη φυλακή. Η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία κηρύχθηκε εκτός νόμου το 1948. Οι κληρικοί ρίχθηκαν στις φυλακές, το δύο και οι προτεστάντες κληρικοί. Μόνο και μόνο επειδή δεν δέχθηκαν να υπογράψουν ε, δηλώσεις ε, απόδεχόμενη την κομμουνιστική ιδεολογία. Αυτή ήταν η καταστολή του κομμουνιστικού καθεστώτος. Η γη κατασχέθηκε, έκλεψαν τη γη μας. Όλα αυτά οδήγησαν στον αγώνα στην Επανάσταση του 1989, όταν πια δεν μπορούσαμε άλλο. Η δημοκρατία επιτέλους επέστρεψε το Δεκέμβριο του 1989 και χαίρομαστε που είμαστε εδώ όλοι οι Ρουμάνοι γιατί κάναμε κι εμείς ε, αγώνα για την δημοκρατία. Η Πρόεδρος παρακαλώ να τηρείτε τον χρόνο που σας έχουμε δώσει για την Renew Europe ο κ. Τσιόλος. Σας ευχαριστώ. Πριν από 30 χρόνια, 16 Δεκεμβρίου 1989, στην ε, Τιμισοάρα ξεκίνησε η Ρουμανική Επανάσταση. Κάποιες εκατοντάδες άτομα ε, ξεκίνησαν και επιχείρησαν να ρίξουν ένα ολοκληρωτικό καθιστώς. Στις επόμενες ημέρες ε, προσθέθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες άτομα στο πλευρό τους και η Επανάσταση διαδόθηκε στο Βουκουρέστι, στο Κλούζ, σε ολόκληρη τη χώρα. Ξεκίνησαν οι συγκρούσει κανεί δεν ήξερε τι θα γίνει. Γνώριζαν ότι κινδυνεύει η ζωή τους. Κατέβηκαν στις ε, πλατείες, ε, κατήγγυλαν τη δημοκρατία, την δικτατορία, την καταστολή, την έλλειψη ελευθερίας, ε, την οικονομική αθλειότητα. Σήμερα λοιπόν εμείς τιμούμε αυτά τα άτομα ακριβώς για να τιμήσουμε την επιστροφή της Ρουμανίας στις αρχές δημοκρατίας, του πλουραλισμού, του δικαίου, της ελευθερίας και για το ότι επανήλθε στην ελεύθερη και δημοκρατική Ευρώπη. Τις ε, μέρες αυτές λοιπόν ε, αρκετοί από αυτούς ε, έπεσαν, δεν γύρισαν ποτέ στο σπίτι τους. ενός γνωστού μάλιστα ο Γιο γύρισε με ένα ματωμένο που κάμισε στο σπίτι γιατί ένας φίλος του είχε πεθάνει στα χέρια του. 22 του μηνό ε, πήγε ε, στην δουλειά του και μετά ε, κατέληξε στις 26 του μηνός. Ε, παιδιά έχασαν τους γονείς τους κτλ. Πέρσι τα ονόματα τους τιμήθηκαν στην πλατεία της Ελευθερίας. Ε, το μικρό αυτό παιδάκι πλέον έχει μεγαλώσει και θυμάται την θυσία των γονιών του. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν πρέπει εμείς να παλέψουμε έτσι ώστε ποτέ ξανά να μην κατεβαίνουν οι πολίτες ε, στις πλατείες για να πεθαίνουν για την ελευθερία τους. Ε, ούτε τώρα ούτε για τις ε, μελλοντικές γενιές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα για τους πράσινους, ε, για δύο λεπτά, ο κύριος Μπιουτικόφερ. Κύρια Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, για αυτούς που θυσίασαν τη ζωή τους στην Ρουμανική Επανάσταση ή τραυματίστηκαν. Για τις οικογένειες που θρύνησαν θύματα βεβαίω δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε την θλίψη μας. Θεωρώ ότι είναι η πιο πολύτιμη κληρονομιά που μοιραζόμαστε στην Ευρώπη, ότι έχουμε τόσο πολλά παραδείγματα για το πώς ε, στις ε, χώρες μας θαραλέοι, γενναίοι, άντρες και γυναίκες παλεύουν για την ελευθερία και την δημοκρατία και με υψηλό προσωπικό τίμημα. Θεωρώ ότι το κοινοβούλιο αυτό εδώ πέρα έχει αρκετά μεγάλη συνένεση. Καμία συνένεση όμως δεν υπάρχει από τη δική μου την ομάδα για την προσπάθεια που γίνεται τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εισαχθεί μια νέα πρακτική η οποία σταδιακά συντάσσει διάφορα ψηφίσματα για την ιστορία της Ευρώπης και ε, διαπιστώνει και ορίζει μετά ποια είναι η αλήθεια για την ε, ιστορία της Ευρώπης. Όποιος αναζητεί την αλήθεια πρέπει να αναζητήσει την ποικινομορφία και να δεχτεί την αντιπαράθεση και θα πρέπει να πάει στον οίκο της ιστορίας. Αλλά δεν είναι αποστολή του Κοινοβουλίου να αποφασίζει κατά πλειοψηφία ποια είναι η αλήθεια για ιστορικά γεγονότα. Και θεωρώ ότι ε, δεν βοηθάει αυτό, ανεξαρτήτως του από ποια πλευρά έρχεται, από κέντρο, αριστερά, δεξιά θεωρώ ότι είναι λάθος αυτός ο δρόμος. Γι' αυτό θέλω και η ομάδα μου παρακαλά τις άλλες ομάδες να ξανασκεφτούν αν θέλουν να ακολουθήσουν αυτήν την πορεία. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να δείξουμε σεβασμό χωρίς να μπούμε σε αυτό το αδιέξοδο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τους ε, συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ. για 1,5 λεπτό ο κύριο Προκατσίνη. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα τιμούμε την ε, τελευταία πράξη αυτής της εκπληκτικής εποχής των λαών και της ελευθερίας που ζήσαμε στην Ευρώπη το 1989. Τιμούμε το θάρρος χιλιάδων ανθρώπων, ανδρών και γυναικών που θυσίασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία έτσι ώστε τα παιδιά τους να μπορέσουν να ζήσουν σε ε, μια χώρα ελεύθερη επιτέλους από την κομμουνιστική καταπίεση. Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρω τα λόγια ενός μεγάλου διανοούμενου, ε, χριστιανού, Ρουμάνου, του Καμίλα Δεμετρέσκου, που έλεγε ότι θέλαμε πάντα να ζήσουμε σε αυτήν την ε, χώρα μας ε, σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν ήθελε να καταλάβει ότι ήδη η κομμουνιστική οτοπία είχε καταδικαστεί από την ιστορία. Όλη η χώρα λοιπόν έβγαινε στα παράθυρα. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα ένα φόρο αιματος τον οποίο πρέπει να τιμήσουμε αν και έχουν περάσει τόσα χρόνια. Να πω και κάτι άλλο. Οι αρχές αυτή τη ρουμανικής Επανάστασης συνεχίζουν να ανθούν ανά τον ε, κόσμο. Παραδείγματο χάρη έχουμε τους νέους στο Χονγκ Κόνγκ που διώκονται σήμερα από το κινέζικο κομμουνιστικό καστός με πλήρη αδιαφορία από τον υπόλοιπο κόσμο. Πάλι νέοι, πολύ γενναίοι, εξίσου γενναίοι με τους ε, νέους ε, της Τιμισοάρας, του Βουκουρεστίου και της πλατείας Τιέναν Μέν. Thank you very much now for... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για δύο λεπτά ο κύριος Μουρεσάν. doamnă președintă, stimați colegi, pe 16 decembrie 1989, în urmă cu exact 30 de ani. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακριβώς πριν από 30 χρόνια κατέβηκαν για πρώτη φορά οι Ρουμάνοι στις ε, πλατείες και τους ακολούθησαν τις επόμενες ημέρες εκατοντάδες χιλιάδες ε, Ρουμάνοι. Όλα αυτά οδήγησαν στην κατάρρευση του κομμουνισμού στην ε, Ρουμανία και επανήλθε βεβαίως η Ρουμανία στα χέρια του λαού της ε, και στην Ευρώπη. Εκατομμύρια λοιπόν Ρουμάνοι βγήκαν στους δρόμους για να μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα, για να συγκεντρώνονται ελεύθερα, για να ταξιδέψουν στο εξωτερικό ο ρουμανικός λαός ε, κατάκτησε με μεγάλες ε, θυσίες ε, την θέση του στην Ευρώπη. Η λέξη κλειδί εδώ πέρα, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συναδελφοί, πρέπει να είναι η μνήμη. Σήμερα πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο από ποτέ τους 1142 Ρουμάνους που έχασαν την ζωή τους στην επανάσταση αυτή, ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ε, έπεσε ειρηνικά το καθεστώς. Σε εμάς στην Ρουμανία θυσιάστηκαν 1.142 άνθρωποι. Πολλοί από αυτούς νέοι πολέμησαν ε, για την δημοκρατία, για την ελευθερία, για την ελευθερία έκφρασης ε, και πρέπει να τους ε, σκεφτόμαστε σήμερα. Τα τελευταία 30 χρόνια οι Ρουμάνοι συνέχισαν αυτόν τον αγώνα, έναν αγώνα για τις ευρωπαϊκές αξίες και για να κατακτήσουμε τη θέση της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Πρόεδρε, εμείς όλοι οι ευρωβουλευτές από τις 28 ε, χώρες έχουμε το καθήκον να υπερασπιστούμε τις αξίες για τις οποίες έδωσαν τη ζωή τους οι Ρουμάνοι το 1989. Την δημοκρατία, την ελευθερία, την ελευθερία έκφρασης, τη δικαιοσύνη και πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την ειρηνική ένταξη των χωρών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μπενέα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Ξέρετε τότε υπήρχε ένας άνθρωπος που λεγόταν Νικήτας και ζούσε μια απολύτως φυσιολογική ζωή. Ήθελε, σκόπευε να παντρευτεί την επόμενη χρονιά, τότε το 1989, αλλά στις 22 Δεκεμβρίου δυστυχώς πέθανε. Μία σφαίρα του αφαίρεσε τη, ζωή κατά τη διάρκεια της Ρουμανικής Επανάστασης. Ήταν ερευνητής στο επιστημονικό πεδίο της φυσικής. Η οικογένειά του τον ονόμαζε Γεώργιος ο Θαραλέος και δεν κατάφερε ποτέ να ε, ζήσει τη ζωή που ονειρευόταν. Έχασε τη ζωή του, σκοτώθηκε και βρίσκεται σήμερα στο νεκροταφείο του Μπακάου. και κάθε, χρόνο, κάθε χρόνο στις 22 Δεκεμβρίου έρχεται η μητέρα του και θέτει το ίδιο ερώτημα επιτακτικά. Ποιος είναι αυτός που σκότωσε το γιο μου. Είναι χιλιάδες τα θύματα κατά τη διάρκεια της Ρουμανικής Επανάστασης και θα πρέπει να χυθεί άπλετο φως σε αυτή την κατάσταση ε, και θα πρέπει να επικρατήσει εκ νέου ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γι' αυτό θέλουμε να διαλευκάνουμε όλα αυτά τα περιστατικά και να ε, να δώσουν λόγο οι ένοχοι ενώπιον της δικαιοσύνης. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Madam Επόμενος ο ομιλητής από το Ρηνιού, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Εορτάζουμε φέτος ε, την 30η επέτειο από την Ρουμανική Επανάσταση. Είναι η μόνη χώρα στην οποία το κομμουνιστικό καθεστώς αγωνίστηκε για να παραμείνει στην εξουσία παρά τη στεναρή αντίδραση του ρουμανικού λαού. Πάνω από χίλια άνθρωποι βρήκαν το θάνατο, 3.000 και παραπάνω ήταν οι τραυματίες κατά τη διάρκεια των ε, δράσεων καταστολής από τις αστυνομικές αρχές προς το λαό της Ρουμανίας. Ε, τα περισσότερα θύματα ήταν στην Τιμισοάρα και το θάρρος που έδειξαν ήταν κάτι το απίστευτο να υψώσουν τη φωνή τους, να προτάξουν τα στήθη τους ενάντια του κομμουνιστικού καθεστώτος, ενώ ήταν απολύτως μόνοι τους. Δεν φαντάζονταν ποτέ ότι οι αρχές καταστολής θα τολμούσαν να πυροβολήσουν άοπλους άντρες, γυναίκες και παιδιά. Και παρά τους πυροβολισμούς αυτούς, ο λαός της Τιμισοάρα παρέμεινε στο δρόμο εκεί να αντιστέκεται υπό τον καταιγισμό των ρηπών και των πυροβολισμών. Αυτή είναι η πιο ζωντανή ανάμνηση που έχουμε από το 1989. Έβλεπαν εκεί στην πλατεία τους διπλανούς τους, τους φίλους τους, τους συγγενείς τους να πέφτουν από τις ε, σφαίρες των δυνάμεων καταστολής. Θα μπορούσαν να είχαν ε, φύγει τρέχοντας, αλλά δεν το έπραξαν. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό αποτείουμε φόρο, φόρο σε αυτά τα θύματα διότι ακριβώς το αξίζουν. Η Ρουμανική Επανάσταση του 1989 είναι η στιγμή της ιστορίας μας η οποία αποδεικνύει πόσο μεγάλη ισχύ έχει ο λαός, έχουν οι πολίτες όταν αγωνίζονται από κοινού για να υπερασπιστούν τις αξίες τους. Βγήκαμε όλοι τότε στο δρόμο και το γεγονός ότι ήμασταν όλοι μαζί είναι που μας έδωσε τη δυνατότητα να καταπολεμήσουμε τα πολιταρχικά και αυταρχικά καθεστώτα και οφείλουμε πάντοτε να είμαστε έτοιμοι να το πράξουμε. Οφείλουμε να απαιτήσουμε αλήθεια, αποκατάσταση της αλήθειας και δικαιοσύνη για όσους ε, διακινδύνευσαν τη δική του ζωή κατά τη διάρκεια αυτών των σκοτεινών ημερών. Θα πρέπει λοιπόν να ανοίξει αυτό το σκοτεινό κεφάλαιο, να χυθεί άπλετο φως στην ιστορία της Ρουμανικής Επανάστασης. Θα πρέπει να πούμε την αλήθεια, να μάθουμε ποιοι είναι οι ένοχοι αυτής ε, της τραγωδίας του 1989 ε, για να μπορέσουν να ξεκουραστούν ευχαριστούν εν ειρήνη οι ήρωές μας. Ευχαριστώ για το ΕΛΚ. Η κυρία Γκάλ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν από 30 χρόνια ξεκίνησε η επανάσταση στην ε, Ρουμανία. Ρουμάνοι, Σέρβοι, Ούγγροι ξεσηκώθηκαν κατά της πρότασης ε, του Επισκόπου Τέκες γιατί πλέον δεν άντεχαν ε, την ε, καταστολή του κομμουνιστικού καθεστώτος. Διαμαρτυρήθηκαν για την καταστροφή χώριων από τον Τσαουσέσκου, διαμαρτυρήθηκαν υπέρ των οικογενειών τους κατά του καθεστώτος. Αυτές οι αξίες ακριβώ μας καθοδηγούν στην Ρουμανία και στην Ουγγαρία. Και πρέπει να αναφέρουμε και τα όσα έκανε ο Επισκοπός Τέκιος. Ναι, είχαμε λοιπόν ε, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ε, τα οποία πρέπει να θυμόμαστε. Είναι μια στιγμή στην ιστορία της Ευρώπης όπου πάλεψαν διάφοροι λαοί ο ένας στο πλευρό του άλλου και είχαμε την επανάσταση στην Τιμισοάρα, στη Ρουμανία. Ε, μια κοινή ευρωπαϊκή αξία την οποία πρέπει να θυμόμαστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκάλ. Δέχεστε μια μπλε κάρτα τον κύριο Γιουρτάνοφ. Ναι. Κύριε Γιουρτάνοφ, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, λαμβάνω το λόγο. Γιατί άκουσα αυτά που άκουσα. Θέλω να ευχαριστήσω τη συναδελφό. Όμως να προσθέσω ότι πρέπει να αποτείνουμε φοροτιμής σε αυτούς που έχασαν τη ζωή τους. Αυτό κάνουμε σήμερα, να αποτείνουμε φοροτιμή στους νεκρούς. Όσα βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τη Βουλγαρία. Θέλω να θυμίσω ότι στις 14 Δεκεμβρίου της χρονιάς εκείνης, οι πολίτες της Σόφιας είχαν αποκλείσει το Βουλγαρικό Κοινοβούλιο και απαιτούσαν την κατάργηση του άρθρου 1 του Βουλγαρικού Συντάγματος, στο οποίο λεγόταν ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι... Α, με συγχωρείτε, λέει η πρόεδρος Διακόπτη, ε, Ερώτηση περιμένουμε από εσά. Αν δεν έχετε ερώτηση, έχετε ερώτηση για την κυρία Γκάλ ή όχι. Αλλιώ πρέπει να σα αφαιρέσω το λόγο. Έχετε ερώτηση, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, το ερώτημά μου είναι το εξή. Κύριε Γκάλ, είστε πεπισμένοι ότι σήμερα που ακόμη έχουμε δικτατορίες ότι πρέπει να συνεχίσουμε ή όχι στην προσπάθεια να προλάβουμε περαιτέρω μετοχυσίες. Είστε πεπισμένοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να, συνεχίσει να κάνει ό,τι μπορεί κατά των δεκτοριών. Ευχαριστώ. Κύριε Γκάλ. Κύριε Πρόεδρε, όπως ε, μόλις είπα, η ελευθερία αυτή είναι κομμάτι της ευρωπαϊκής μας ε, ταυτότητας και η επανάσταση αυτή πριν από 30 χρόνια στην Ρουμανία είναι επίσης μια κοινή ευρωπαϊκή αξία, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα σήμερα. Ε, γιατί ακριβώς το σεβόμαστε και το τιμούμε. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για ένα μισή λεπτό, ο κύριος Λιμπεράτσικη. Παρακαλώ, από τους σοσιαλιστές. Κύριε Πρόεδρε, είμαι Πολωνός, δεν είμαι Ρουμάνος. Εξαίρεση σε αυτήν την συζήτηση. Και στην Πολωνία πριν από 40 χρόνια, το 1980, το σύστημα άρχισε να κλειδονίζεται. Τον Ιούνιο ξεκίνησε η πτώση του παλαιού καθεστώτος. Τον Νοέμβριο του 89, θυμάστε, το τείχος του Βερολίνου δεν υπήρχε πια. Η Ρουμανία, η Βόρειος Κορέα και η Κούβα ήταν τα μόνο απομεινάρια, τα τελευταία καταφύγια του παλαιού καθεστώτος και γι' αυτόν τον λόγο υποστηρίζω το σχετικό ψήφισμα το οποίο καταδικάζει τον εγκληματικό χαρακτήρα του συστήματος. Βεβαίως από την εποχή εκείνη η Ρουμανία δίνει σε δρόμο μακρύ. Είναι καιρός να αποτείνουμε φόρο τιμή στα θύματα σε όσους έδωσαν τη μάχη και που, συνεχίζουμε, και που συνεχίζουν τον αγώνα για την επιτυχία της Ρουμανίας. Χαιρετίζουμε λοιπόν με ικανοποίηση την προσχώρηση μεταξύ άλλων της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εύχομαι κάθε καλό στην Ρουμανία και να γίνει σύντομα μέλος και της ζώνης Σέγγεν. Πρόεδρος, δύο λεπτά ο κύριος Μοντρεάν, παρακαλώ, από το ΕΛΚ. Κυρία Πρόεδρε, φέτος εορτάζουμε τα 30 χρόνια από την ε, Ρουμανική Επανάσταση του Δεκεμβρίου του 1989. Οι βιότητε είναι ακόμη στο μυαλό των ε, ανθρώπων που έδωσαν τη μάχη κατά του αιματοβαμένου καθεστώτος. Η επανάσταση αυτή του Δεκεμβρίου του 1989 δεν αφορούσε όμω μόνο τους Ρουμάνους. Αφορούσε όλους τους Ευρωπαίους οι οποίοι την εποχή εκείνη διαδήλωναν υπέρ του ρουμανικού λαού. Και άλλοι λαοί, εκτός από τους Ρουμάνους, τα τελευταία 30 χρόνια προσπαθούν να βρουν απαντήσεις. Τι έγινε εκείνο τον Δεκέμβριο του 1989 στη Ρουμανία. Ακόμη περιμένουμε απαντήσεις. Θέλουμε όλοι υπεύθυνοι επιτέλους να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και να καταδικαστούν. Αυτό απαιτούν τα θύματα. Στην ρουμανική κοινωνία, ξέρετε, υπάρχει ακόμη ο φόβος ότι η ελπίδα αυτή ότι κάτι θα γίνει, ότι η υπόθεση θα διαλευκανθεί, δεν θα ευοδοθεί, δεν θα ποτέ. Οι Ρουμάνοι ακόμη αναζητούν την αλήθεια. Πρέπει να μιλήσουμε με τους πρωταγωνιστές και με τα θύματα για να καταλήξουμε κάπου. Αλλά όπως είπα, πολλοί φοβούνται ότι δεν πρόκειται ποτέ να έχει φως άπλετο στην υπόθεση αυτή. Πρέπει να καταλάβουμε, πρέπει να μάθουμε ποιος εξεγέρθηκε, κατά ποιου, ποιος ήταν ε, επικεφαλής των δυνάμεων που είναι υπεύθυνε για τα θύματα. Πρέπει κάποτε να μάθουμε την αλήθεια. Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για, την, για τις βιότητες της εποχής εκείνης. Πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή η αλήθεια να λάμψει. Ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε πολύ άλλωστε. Αυτό είναι και ο στόχος αυτού του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλουμε ο Δεκέμβρης του 1989 να μην ξεχαστεί. Να γίνει φάρος ελευθερίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μοντριάνου. Δέχεστε μπλε κάρτα από τον κύριο Σοκόλ. Ναι. Κύριε Σοκόλ, παρακαλώ. 30 δευτερόλεπτα για ερώτηση. Ευχαριστώ. Θέσατε το ερώτημα ποιος είναι υπεύθυνος, ποιος φταίει για τους νεκρούς στην Επανάσταση. Να επέκταθω λοιπόν. Γνωρίζουμε τι συνέβη με τον ε, Τσαουσέσκου. Σημαίνει αυτό ότι η πτώση του Τσαουσέσκου ήταν και η πτώση του καθεστώτος. Οι κομμουνιστές ε, παρέμειναν ε, στις θέσεις τους, στα πανεπιστήμια, στις αρχές, στην διοίκηση. Ήταν υπεύθυνοι για αυτό το έγκλημα, αλλά δεν καταδικάστηκαν. Ε, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι ακόμα και εξακολουθούν να αποτελούν πρόβλημα για την ε, Ρουμανία. Παρακαλώ, έχετε λόγο. 30 δευτερόλεπτα. Κοιτάξτε, στην Ρουμανία η αλήθεια ποτέ δεν έλαμψε. Το δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξέδωσε σχετική απόφαση και κάλεσε να γίνουν προσπάθειες για να λάμψει αλήθεια. Εγώ στην παρέμβασή μου είπα ότι η Ρουμανία είχε υποφέρει πολύ. Και το ακόμα χειρότερο είναι ακριβώς αυτό, ότι από το 89 δεν βρέθηκαν ποτέ οι υπεύθυνοι. Το αίτημα λοιπόν εκείνη τη επανάσταση παραμένει ακόμα και σήμερα ζωντανό. Ευχαριστώ. Λέει πρόεδρο, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ως γυναίκα που ζήτησε τη μισή τη ζωή σε καταπίεση, πρέπει να πω ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο ταπεινωτικό από το να ζει κανείς σε δικτατορία. Η μετάβαση από τη μία κατάσταση στην άλλη, από τη δημοκρατία στη δικτατορία και τον Μπαλίν, πολλές φορές μπορεί να είναι θέμα πολύ μικρού χρόνου. Λοιπόν, το Δεκέμβριο του 89 πολλοί βρήκαν το θάνατο από σφαίρε από αυτούς, από τα χέρια αυτών που συνεργάστηκαν με το καθεστώς, που ήταν συνυπεύθυνοι με το καθεστώς. Να μην ξεχάσουμε λοιπόν ποτέ το 89. Είναι χρέος μας Γι' αυτό και σήμερα εορτάζουμε την 30η επέτειο. Θυμόμαστε τους νεκρούς που πολέμησαν την δικτατορία. Πολλοί κινδύνευσαν μόνο και μόνο εξαιτίας αυτών που πίστευαν. Αυτό είναι δικτατορία. Τώρα δεν μπορεί κανείς να δηλώσει καν αυτά τα οποία σκέφτεται. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε ξανά τη μάχη μέχρι την πτώση κάθε δικτατορίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά, ο κύριος Βίντσε. Κυρία Πρόεδρε, πριν από 30 χρόνια, τα κομμουνιστικά καθεστώτα κατέπεφταν το ένα μετά από το άλλο στην Ευρώπη. Το φως έλεμψε πάνω από την Ανατολική Ευρώπη. Όμως το καθεστώς Τσαουσέσκου φαινόταν να είναι εγκιστρωμένο στην εξουσία περισσότερο από άλλα. Ξέσπασε όμως ε, η Επανάσταση, η Ελπίδα στις πόλεις και στα χωριά της Ρουμανίας. Από την εποχή εκείνη όμως πολλά ερωτήματα επικρέμανται χωρί να βρίσκουν απάντηση. Έγινε μια μεγάλη αδικία, η οποία παραμένει και σήμερα. Οι Ρουμάνοι διερωτώνται τι έγινε. Ο αγώνας έγινε για την δημοκρατία και ο αγώνας αυτός δεν έχει ολοκληρωθεί. αναζητούμε όλοι μας την αλήθεια. Τι έγινε την εποχή εκείνη στη Ρουμανία. Αυτό αναζητούμε όλοι μας. Θέλουμε να επιστραφούν οι περιουσίες και η γη που έκλεψε το κομμουνιστικό καθεστώς. Γιατί δεν είναι μόνο οι νεκροί, αυτοί που έχασαν τη ζωή τους τένα χρόνια πριν. Και δεν υπάρχει χρόνος. Ήρθε η στιγμή να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, και να καταβληθούν και αποζημιώσει σε αυτού στα θύματα του κομμουνισμού για να βασιλέψει το δίκαιο στην κοινωνία μα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Ο κύριο Τσιοντάρου. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα Μιλάμε για το θάρρος ε, του ρουμανικού λαού απέναντι σε ένα δικτατορικό καστός, ε, στο ότι πολέμησε κόντρα στο κρύο, στην πείνα. Τις 14 ε, Δεκεμβρίου στο Ιάσιο άνοιξε ο δρόμος της Επανάστασης, παρά το ότι είχαμε παρέμβαση της Σεκουριτάτε ε, χωρίς την οποία η κατάσταση θα ήταν ε, τελείως ε, διαφορετική. Εγώ τα έχω πει αυτά στην κόρη μου και βεβαίω μεγάλωσε πιστεύοντας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί θα πρέπει να πέσουν και οι άλλοι τύχοι. Πρέπει να αναγνωρίσουμε το θάρρος των πρωταγωνιστών της Επανάστασης και να κάνουμε κάτι το πάρα πολύ σημαντικό σήμερα μετά από 30 χρόνια σας υπενθυμίζω ότι πληρούμε τους όρους για να μπούμε στην ζώνη Σέγγεν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Γραπίνη για 1,5 λεπτό έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, εγώ είμαι από την, ε, τη Μισοάρα. Πριν από 30 χρόνια ήμουν στους ε, δρόμους στο πλευρό των άλλων πολιτών της πόλης αυτής και σας παρακαλώ να αντιληφθείτε ότι η Επανάσταση δεν ανήκει σε ένα άτομο ή σε μια ομάδα. Είναι η Επανάσταση των Ρουμάνων, των κατοίκων της τη που άναψε το φυτίλι και μετά διαδόθηκε σε ολόκληρη την χώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ήταν μια επανάσταση παλαϊκοί βγήκαν οι άνθρωποι από τα εργοστάσια από όλε τι γωνιέ τη ε, Τιμισοάρα και στι άλλε πόλει κατέβηκε ο κόσμο στι πλατείε. Σήμερα λοιπόν τιμούμε αυτό το γεγονό. Και ε, θα ήθελα εδώ να υπενθυμίσω τους νεκρούς κατοίκους της ε, Τιμισοάρας που βγήκαν άοπλοι στου δρόμους απέναντι ε, σε αυτούς που τους ε, πυροβολούσαν. Λοιπόν, έχουμε την υποχρέωση απέναντι σε αυτούς να σεβαστούμε τον λαό της Ρουμανίας που είναι φιλοευρωπαϊκός. Ο ρουμανικός λαός είναι υπέρ της Ευρώπης και η θέση μας είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ζητάω από Συμβούλιο Κοινοβουλίου και Κομισιόν να σεβαστούν τα δικαιώματα των Ρουμάνων να αναγνωριστεί η αξιοπιστία μας γιατί έχει αλλάξει πολύ η Ρουμανία τα τελευταία 30 χρόνια. Ίσως να μην το ξέρετε, αλλά είστε πάντα ευπρόσδεκτοι σε μας. Αυτά λοιπόν και το μήνυμα βεβαίω είναι ενότητα και αγάπη προς την πατρίδα μας. Ευχαριστώ για τη διαδικασία ΚΑΤΣΤΙΑΙ. Θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους που δεν έχουν πάρει το λόγο. Για ένα λεπτό ο κύριος Τόματς, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πριν από 30 χρόνια, ξέρετε, ακριβώς σαν σήμερα, χιλιάδες ήταν οι Ρουμάνοι που νίκησαν το φόβο τους, που βγήκαν στο δρόμο, που απέτησαν να πέσει επιτέλους αυτό το εγκληματικό και δικτατορικό καθεστώς. Πάνω από 12 εκατομμύρια πυροβολισμοί σημειώθηκαν εναντίον αυτών που φώναζαν «Ελευθερία σ' αγαπώ, για σένα είμαι έτοιμος να πεθάνω». Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πλημμύρισαν τους δρόμους πριν από 30 χρόνια εξέφρασαν αυτή τη βαθιά τους επιθυμία, τη σφοδρή επιθυμία για ελευθερία. Και αυτοί είναι που έφεραν τη Ρουμανία στο δρόμο που την οδήγησε στη δημοκρατία και στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Από εκείνη τη μέρα η Ρουμανία γύρισε οριστικά την πλάτη στα κομμουνιστικά καθεστώτα κατά τη διάρκεια των οποίων πάρα πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κλεισμένοι σε μπουντρούμια. Θα ήθελα αγαπητοί συνάδελφοι σήμερα να είμαστε σε θέση να αποτίσουμε φόρο τιμής σε αυτούς τους ήρωες που πέθαναν για την ελευθερία μας. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, ξέρετε, πράγματι είναι αληθές ότι πριν από 30 χρόνια, τη στιγμή που συνέβαιναν αυτές οι δραματικές εξελίξεις στη Ρουμανία, είδαμε παράλληλα ε, και την κατάληξη του καθεστώτος Τσαουσέσκου. Δεν ήταν καθόλου εύκολο να τους πολεμήσει κανείς. Παρεμφερή ήταν τα κινήματα και οι δράσεις στη Τσεχοσλοβακία, ξέρετε. Το επίπεδο ζωής ήταν παρόμοιο, ήταν παρεμφερές. Η δημοκρατία είναι ένα καθεστώς που σίγουρα έχει ελλείψεις και πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να καλύψουμε αυτό το δημοκρατικό έλλειμμα που σημειώνεται. Θέλουμε να εξαντληθούν τα νομοθετικά και τα νομοπαρασκευαστικά μέσα για να εξεταστεί εκ του σύνεγγυς η κατάσταση που έχει να κάνει με το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί παντού υπάρχουν ε, αδύναμοι κρίκοι. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό η επόμενη ομιλήτρια, παρακαλώ, κυρία Ντέιλι. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, ξέρετε, εγώ πριν από 30 χρόνια ήμουν φοιτήτρια στην Ιρλανδία και εμπνεύστηκα από τον ηρωισμό των φοιτητών των Ρουμάνων και γι' αυτό πήρα, ταξίδεψα αμέσω και πήγα στην ε, Μισοάρα και πέρασαν ένα μήνα ανάμεσα σε αυτού ε, κατά τη διάρκεια αυτή τη επαναστατική εποχή. Και ήταν ε, ένα από τα συμβάντα τη νιώτη μου που πραγματικά με σημάδεψαν στη συνέχεια. Είδαμε την πτώση του καθεστώτος Τσαουσέσκου, ήταν μια ελίτ η οποία πλούτιζε σε βάρος του πληθυσμού η οποία είχε αναπτύξει ένα κρατικό μηχανισμό για να μπορεί να συνεχίσει να διαβιεί παρασιτικά σε βάρος του υπολείπου λαού. Είδαμε τις ελπίδες του λαού για μια πιο ασφαλή ζωή, για ελευθερία, για δημοκρατία, για οικονομική ανάπτυξη και αυτά είναι βιώματα τα οποία μας θύμισαν το πόσο ταπεινό είναι το ανθρώπινο όν και πόσο μεγαλειώδης ε, η κοινωνία και η μάχη αυτών των λαών. Θα πρέπει ε, αυτές τις ελίτες να τις κατα να, να αντιστεκόμαστε σε αυτές. Σήμερα έχουμε νεοφιλελεύθερες ελίτ. Γιατί η Ρουμανία έχει το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό προσφύγων. 5 εκατομμύρια Ρουμάνοι ζουν εκτό τη χώρα, το δεύτερο μεγαλύτερο μετά τη Συρία. Υπάρχει τεράστια διαφθορά. Η επανάσταση μπορεί να ξεκίνησε, αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, ο κύριος Γουίνκλερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πράγματι, η Επανάσταση ξέσπασε στην Τιμισοάρα πριν από 30 χρόνια. Όταν ε, οι Ρουμάνοι και οι Ούγγροι συγκεντρώθηκαν μπροστά σε μία εκκλησία για να προστατεύσουν έναν κληρικό. Αυτό ήταν το ένασμα, η αφορμή. Και ε, επέδειξαν τέτοια ελληνική ώστε να φτάσουν σε ένα ε, απόγειο αντίστασης που ήταν πρωτόγνωρο ε, για το ρουμανικό λαό. ο αγώνας μετατράπηκε σε κοινό στόχο του λαού για να μπορούν να έχουν όλοι αυτού του είδους την προστασία. Η πολιτική μας ομάδα, όλοι εμείς αγωνιζόμαστε έτσι ώστε οι αξίες που υπερασπιστήκαμε πριν από 30 χρόνια να παραμείνουν ε, ε, προστατευμένες, να παραμείνουν ενισχύ. Αυτόν τον αγώνα το δίνουμε εδώ στην Ευρώπη και κυρίω στο Στρασβούργο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρεθούν οι υπέτειοι όλων αυτών των βιοπραγιών και ε, δολοφόνιων. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό η κυρία Ward παρακαλώ. Συγγνώμη κυρία Πρόεδρε, Βλέπω ότι μία συνάδελφος εδώ ε, θέλει να δείξει μία μπλε κάρτα και έχει ερώτημα στην προηγούμενη ομιλήτρια. Θέλετε αυτό το θέμα το ρυθμίσετε πριν ε, πάρω το λόγο. Όχι, δεν επιτρέπεται η διαδικασία της μπλε κάρτας κατά τη διάρκεια του ΚΑΤΣΔΙΑ. Έχετε το λόγο κυρία Ward. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εκπροσωπώ την ε, βορειοδυτική Αγγλία και εκεί έχουμε μεγάλο, μεγάλο ποσοστό ρουμανικού πληθυσμού με τους οποίους συνεργάζομαι στενά. Πολλοί είναι στενοί μου φίλοι, είναι γιατροί, νοσοκόμοι, νοσηλευτέ, καλλιτέχνες, επιχειρηματίες, δάσκαλοι. Πολλοί από αυτούς θυμούνται τη Ρουμανική Επανάσταση και την ε, ε, σκληρή δικτατορία που προηγήθηκε της ε, Ρουμανικής Επανάστασης. Σήμερα είναι οι Ρουμάνοι ελεύθεροι στη δική τους χώρα και από το 2007 έχουν προσχωρήσει και στην Ευρωπαϊκή. Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, το Brexit αποτελεί μια επίφοβη προοπτική για τη ρουμανική διασπορά, για τους Ρουμάνους ομογενείς εκτός ε, των ε, συνόρων της χώρας τους, οι οποίοι βιώνουν ε, περιστατικά ρατσιστικά τακτικού ε, μίσου. Μία ομάδα παιδιών από τη Ρουμανία που τακτικά παίζει στο δρόμο στο Μάντσεστερ αναγκάστηκαν να μπουν μέσα, τα φώναξαν οι γονεί του, ε, γιατί ανησυχούσαν για την ασφάλειά του σε ένα περιβάλλον ε, όλο ένα και πιο εχθρικό. Δεν έχουν ελευθερία να βγαίνουν στον δρόμο να παίζουν έξω με άλλα παιδιά και αυτό είναι μια θλιβερή επίπτωση του Brexit και τη Βρετανία του Brexit ότι οι άνθρωποι που έχουν βιώσει την απολυταρχία σε αυταρχικά καθεστώτα τώρα νιώθουν ότι δεν είναι ευπρόσδεκτοι ε, ε, στη χώρα που τους υιοθέτησε. Και αυτό είναι πολύ δυστυχέ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Επίτροπε, έχετε το λόγο. Κυρία Βαλέαν. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν έχω και πολλά να προσθέσω σε αυτό το στάδιο. Σα άκουσα όλου πολύ προσεκτικά και θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά, διότι φέρατε αυτό το θέμα προ συζήτηση. Ε, διότι στηρίξατε την προσθήκη αυτού του θέματος στην ημερήσια διάταξη. Σας εύχομαι καλή επιτυχία με το ψήφισμα της Πέμπτης και ε, θεωρώ ότι για τους Ρουμάνους, για εμάς, το γεγονός ότι ζούμε στην Ευρώπη, ότι είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι μπορούμε να δουλέψουμε για το καλό όλων, είναι κάτι το οποίο μας ε, ε, κάνει να αναλογιζόμαστε το ύψος της ευθύνης που φέρουμε, γιατί ουσιαστικά ε, κομίζουμε μαζί μας τις ελπίδες όλων αυτών των ανθρώπων που επαναστάτησαν το 1989 γιατί ζήτησαν μια καλύτερη ζωή για όλους και μια καλύτερη Ευρώπη. Και αυτή, αυτή η σκέψη θα μας συνοδεύει πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Λίγη συζήτηση για αυτό το θέμα. Η σχετική ψηφοφορία θα λάβει χώρα την Πέμπτη. Προχωρούμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Κοινή συζήτηση για την απάτη στο τομέα του ΦΠΑ και πάροχη υπηρεσιών πληρωμών. Θα παρακολουθήσουμε την παρουσίαση της κυρίας Λίδια Περέιρα που έχει συντάξει την έκθεση απαιτήσει για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών αλλά θα μιλήσουμε και για την έκθεση επίσης της κυρίας Λίδια Περέιρα για, με αντικείμενο τα μέτρα ενίσχυσης διοικητικής συνεργασία για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Είναι δυνατόν κανείς να ζητήσει να συμμετάσχει στη διαδικασία Catch the Eye αλλά και στη διαδικασία της Black κάρτα και έχετε οδηγίες σχετικά και για την ηλεκτρονική ψηφοφορία και για τον ηλεκτρονικό τρόπο ε, παρέμβασης στην είσοδο. Ε, η κυρία Περέιρα έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, οι κοινωνίες μας ψηφιοποιούνται όλο και περισσότερο και οι οικονομίες μας ψηφιοποιούνται όλο και περισσότερο και αυτό δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τους περισσότερους πολίτες. Έχουμε νέα προϊόντα, νέα παροχή υπηρεσιών, ε, νέα ε, παροχή επίσης αγαθών Έχουμε πρόσβαση δηλαδή σε νέους τρόπους απόκτησης και λήψης υπηρεσιών και αγαθών, όμως αυτά τα φαινόμενα οδηγούν στην αύξηση των περιστατικών απάτης. Η ψηφιοποίηση της οικονομίας απαιτεί την παρέμβαση των επισήμων αρχών διότι διαφεύγουν έσοδα πολύ σημαντικά για τις ελεγκτικές και φορολογικές αρχές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οφείλουμε να προστατεύσουμε την ακαιρεότητα της ενίας αγοράς και την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών. Να καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή και φόρο αποφυγή και ε, να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη του Ευρωπαίου πολίτη στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στις επίσημες αρχές των κρατών μελών. Μιλούμε λοιπόν για την ανακοίνωση των προμηθευτών, των παρόχων της υπηρεσίας και την, ε, ε, μιλούμε για την επικοινωνία μεταξύ τους. Μιλούμε για τον εντοπισμό του κατά πόσο είναι αυτοί νομικές οντότητες στους οποίους μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη. Υπάρχει λοιπόν ένα κενό στην ε, ίσπραξη του ΦΠΑ, η οποία ανέρχεται σε, το οποίο ανέρχεται σε 130 εκατομμύρια ευρώ και πάνω ετησίως. Στο ηλεκτρονικό εμπόριο το ΦΠΑ ε, αντιστοιχεί σε 5 ε, δις ευρώ ετησίως. Τα νούμερα είναι πολύ ψηλά και στην Πορτογαλία και αλλού και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι και να καταπολεμήσουμε αυτή την απάτη η οποία Μα φέρνει σε δύσκολη θέση. Πρέπει να έχουμε δημιουργία ενό ηλεκτρονικού συστήματο για να μπορούμε να συγκεντρώνουμε στοιχεία για τι πληρωμέ και να εντοπίζουμε την ευθύνη των παρόχων και των προμηθευτών, ε, αυτών που προβλέπουν ε, αυτό το σύστημα ηλεκτρονική πληρωμή. Δηλαδή, θέλουμε να καταπολεμήσουμε με πιο φιλόδοξο τρόπο την ε, φόρο διαφυγή και φόρο αποφυγή σε επίπεδο ΦΠΑ. Βασικά στοιχεία της πρότασής μας είναι τα εξής. Διατήρηση στοιχείων και δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να μπορούν να δράσουν πιο αποτελεσματικά οι ελεγκτικές φορολογικές αρχές, να μειώσουμε το ανώτατο όριο την οροφή για την ελάχιστη αξία, για την καταχώρηση στο ηλεκτρονικό σύστημα, έτσι ώστε να μην μπορεί να διαφύγει κανείς και μιλούμε και για την προστασία των δεδομένων η προστασία των δεδομένων πρέπει να υπάρχει, αλλά ε, θα πρέπει να υπάρχει και σωστή εποπτεία. Ε, το σημαντικό είναι όλα αυτά να εναρμονιστούν. Να εναρμονιστούν και τα διάφορα ηλεκτρονικά πρωτόκολλα ώστε να διευκολυνθεί η ζωή των πολιτών και των επιχειρήσεων. Αξιότιμοι συνάδελφοι, ουσιαστικά αυτό το θέμα έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη. Έτσι ώστε όλοι με τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν να αναλαμβάνουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί. Αλλάζει η ψηφιακή τεχνολογία, μας φέρνει πολλά καλά, αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε αγαθά και ε, λαμβάνουμε υπηρεσίες. Οφείλουμε να προσαρμοστούμε ε, στο, στη νέα ψηφιακή εποχή. Η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή σε θέματα ΦΠΑ δεν γνωρίζουν σύνορα και γι' αυτό πρέπει οι φορολογικές και φοροελεγκτικές αρχές να ενισχύσουν τη συνεργασία τους, έτσι ώστε να ε, είναι πρωτοπόροι στην επίτευξη των στόχων μας. Πρέπει να έχουμε μια πιο δίκαιη φορολογική απεικόνηση για να μην ε, διαφεύγει κανείς από τη φορολογική του ευθύνη. Ε, το σημαντικό είναι να επιλέξουμε την πιο ισορροπημένη λύση. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε και κύριοι βουλευτές, είμαι υπερήφανος που στεκόμαι σήμερα εδώ για πρώτη φορά ως Επιτροπός Οικονομικών. Προσβλέπω στο πολύ σημαντικό έργο το οποίο έχουμε να επιτελέσουμε στο οποίο προτεραιότητα κατέχει η καταπολέμηση της απάτης. Ευχαριστώ την κυρία Περέιρα και τα μέλη της Επιτροπής ΕΚΟΝ για την πρόταση που συζητάμε. Η απάτη στον ΦΠΑ απασχολεί όλα τα κράτη-μέλη και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επιτακτική ανάγκη να συζητήσουμε το θέμα με τρόπο δημοκρατικό και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να εξετάσουμε την σημερινή πρόταση σε συνάφη με το πακέτο που συζητά το Συμβούλιο και θα ψηφιστεί στις αρχές του 2020. Πρέπει να αποκτήσουμε ένα ισχυρό, ένα πανίσχυρο εργαλείο για να εντοπίζουμε την απάτη και να την καταπολεμούμε. Απαιτείται δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο λοιπόν. Το 2015, όπως επενθυμίζει η εισηγήτρια, χάθηκαν δισεκατομμύρια μόνο και μόνο επί των εισαγωγών αγαθών. Αντίστοιχα νούμερα αφορούν τις εισαγωγές υπηρεσιών. Φοβούμαι ότι τα μεγέθη αυτά θα συνεχίζουν να αυξάνονται λόγω και της αύξησης του όγκου του εμπορίου. Προτείνουμε λοιπόν να θεσπίσουμε υποχρέωση για τους παρόχους υπηρεσιών να καταθέτουν πληροφορίε των δικαιούχων των υπηρεσιών. Η υποχρέωση αυτή αποσκοπεί στην μείωση του διοικητικού φόρτου, γιατί οι πληροφορίε αυτές ούτω ή άλλω υπάρχουν και χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση αυτών καθ' αυτών των συναλλαγών. Η πρότασή μα λοιπόν αποτελεί πολύ σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση τη απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, αλλά όπω καταλαβαίνετε έχουμε πολλά να κάνουμε μπροστά μα. Η μελέτη της Κομισιόν για το χάσμα του ΦΠΑ δείχνει ακριβώς ότι χάνουμε 137 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Αυτό είναι το νούμερο του 2017. Το νούμερο αυτό είναι απαράδεκτο. Λόγω της κατάστασης κηρύσουμε τον πόλεμο και θεωρούμε προτεραιότητα την καταπολέμηση θα πάρει στον ΦΠΑ κατά τη διάρκεια της θητείας μας. Εννοείται ότι η φορολογική απάτη είναι το αντίθετο της φορολογικής συμμόρφωσης. Πρέπει να δώσουμε μάχη και στα δύο μέτωπα. Αυτό είναι και το σχέδιο δράσης, το οποίο θα παρουσιάσω σε λίγους μήνες. Οι επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να μπορούν να δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην εσωτερική αγορά, επί ίσης με τους παραγωγούς των τρίτων χωρών. Όπως αντίστοιχα οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πρέπει να έχουν πρόσβαση ελεύθερη και στην υπόλοιπη, την παγκόσμια αγορά και πάλι επίσης Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ο Αντιπρόεδρος ο κύριος Κάρας έχει τον λόγο. Κύρια Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Εισηγήτρια, κάθε χρόνο καταγγέλουμε την, το κενό των φορολογικών εισπράξεων κατά 137 δισεκατομμύρια ευρώ στον τομέα του ΦΠΑ ε, για διασυνοριακή απάτη άνω των 50 δισεκατομμυρίων και φορολογική απάντη στο διαδίκτυο που αφορά 90% ε, σχεδόν των ε, συναλλαγών. Γι' αυτό Χαίρομαι ιδιαίτερως για αυτά τα οποία ανακοινώσατε κύριε Επίτροπε για το σχέδιο δράσης αλλά και για, τις ε, εκθέσεις, ε, για την έκθεση της ε, συναδέλφου Φερέρα η οποία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την δημιουργία ενός ενιαίου χώρου ΦΥΠΙΑ και βεβαίω αφορά και τι συναλλαγέ από το διαδίκτυο και θα τεθεί ενισχύ τον Ιανουάριο του 2021. Χρειαζόμαστε λοιπόν αντί για ένα σύστημα με εξαιρέσει και παραθυράκια, ένα σύστημα με κοινού κανόνε. Πρέπει να εμποδίσουμε αυτούς που κάνουν απάτη με ΦΠΑ και να περιορίσουμε το πεδίο δράσης τους και αυτό το λέω και προς την κατεύθυνση του Συμβουλίου παρά τις θετικές ε, αποφάσεις ε, απαιτείται περισσότερη ευρωπαϊκή φορολογική πολιτική και όποιος την μπλοκάρει στηρίζει τους ε, απατεώνες. Πρέπει λοιπόν να καταπολεμήσουμε τη φορολογική απάτη. Χρειάζεται περισσότερη συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών και των υπηρεσιών πληρωμών. και εναρμόνιση όσον αφορά τις διασυνοριακές ε, πληρωμές, ε, πρόσβαση στις πληροφορίες ε, από τις φορολογικές αρχές. Είναι κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα για την αποθήκευση πληροφοριών πληρωμών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Για δύο λεπτά ο Μόλνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια από τις σημαντικότερες αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η κοινωνική δικαιοσύνη την οποία πρέπει να εγγυηθούμε για κάθε πολίτη. Ένα στοιχείο αυτής είναι η δίκαιη φορολογία. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εμείς ως Ευρωβουλευτές πρέπει κάτι να κάνουμε. Δεν πρέπει να αφήσουμε να υπάρχουν παραθυράκια λόγω ελλειπούς ε, συνεργασίας για να γλιτώνουν έτσι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις ε, φόρους ε, στη χώρα μου ο συντελεστής ΦΠΑ είναι ο υψηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιθανώς στον κόσμο με 27% και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, απλά παρακολουθεί το ότι δεν καταλήγουν εκεί που θα έπρεπε τα φορολογικά έσοδα. Μιλάμε για πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ ζημιές και γνωρίζουμε ότι εδώ πέρα υπάρχει και ένας κίνδυνος που συνδέεται με αυτό το ζήτημα, το οποίο αφορά τις συντάξεις, την εκπαίδευση, υπονομεύεται η κοινωνική δικαιοσύνη, η κοινή Ευρώπη και τελικά η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Έχουμε λοιπόν τα έγγραφα, τα έχετε υπόψη σας, έχουμε εργαστεί από κοινού έτσι ώστε να μην πληρώνουν φόρους μόνο αυτοί που έχουν μια οικογενειακή επιχείρηση ή είναι μισθωτοί ο καθένα πρέπει να πληρώνει αυτό το οποίο του αναλογεί και δεν θα πρέπει να υπάρχει κατάχρηση του συστήματος. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των αρχών, ανταλλαγή των δεδομένων έτσι ώστε να μπορέσουμε να πολεμήσουμε την και απάτη του ΦΠΑ. Νομίζω ότι είναι σωστό να εγκριθεί το σχετικό νομοθέτημα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ομάδα Renew για 4 λεπτά. Κόβαρικ. Κύριε Διπρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, χαιρετίζω την δέσμευσή σας, όπως την διατυπώσατε, να καταστήσετε την μάχη κατά της απάτης των ΦΠΑ προτεραιότητα του έργου σας. Έχετε την υποστήριξή μας. Αναφέρετε και κάποια νούμερα όσον αφορά δηλαδή το χάσμα του ΦΠΑ όπως το ονομάζουμε το οποίο τίνει να μειωθεί. Παρ' όλα αυτά μιλάμε ακόμη και σήμερα για περίπου 130 δισεκατομμύρια ευρώ το 18. Θα είναι νούμερο του 18. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, έχουμε και τις α, κυκλικές απάτες που απειλούν το εμπόριο και εκεί έχουμε απώλεια 50 δισεκατομμυρίων σε φόρους. Το νομοθέτημα που συζητούμε θα βοηθήσει τα μάλα στην ανάκτηση απολεσθέντων φορολογικών εσόδων. Η απώλεια αυτή δεν είναι ζημία μόνο για τις κυβερνήσεις, για τα φορολογικά έσοδα. Αυτά πλήττουν ολόκληρη την κοινωνία μας, τις επιχειρήσεις μας και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε πώς υποστηρίζω 100% τον αγώνα κατά της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Από την οπτική γωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουμε θεσπίσει νομοθεσία για την μοντέρνα εποχή μας. Θα συνεχίσουμε το πράγμα αυτό για να διασφαλίσουμε ότι οι κανόνες μας είναι προσαρμοσμένοι στις ανάγκες και με στόχο εν τέλει να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού εισπράξης του ΦΠΑ. Δεν θέλω να ξεχνάτε ότι η κοινοποίηση των πληροφοριών για τον ΦΠΑ, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι εξαιρετικά επιπονή. Έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν οι νέοι κανόνες να μην επιφέρουν ε, αδικαιολόγητα υψηλό φόρτο εργασία, ειδικά στι μικρομεσαίες επιχειρήσει και ειδικά στις διασυνοριακέ συναλλαγέ στην ενιαία αγορά. Αγαπητοί συνάδελφοι, η νομοθεσία που θα θεσπίσουμε πρέπει να βλέπει το μέλλον. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα σύγχρονα επιχειρηματικά μοντέλα, τα οποία συνεχίζουν μάλιστα να εξελίσσονται. Χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφέρει και την ψηφιακή οικονομία, γιατί προς τα εκεί πορευόμαστε. Καλό επίση τι αρχέ, τι φορολογικέ αρχέ που ασχολούνται με τον ΦΠΑ, να υιοθετήσουν προηγμένε μεθόδου τεχνητή νοημοσύνη για να αντιμετωπίσουν την απάτη. Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που θα διαπιστώνει ή θα εντοπίζει με κάποιο τρόπο την πιθανότητα απάτης. Έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και την κυκλική απάτη με τρόπο πιο αποτελεσματικό. Καταλήγοντας, να ευχαριστήσω την συγκητρία και τους συναδέλφους για τη συνεργασία επί των δύο αυτών φακέλων. Έχουμε δύο εκθέσεις που αποτυπώνουν τι προτεραιότητε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά κατά κύριο λόγο την διοικητική συνεργασία στον τομέα των υπηρεσιών. Πιστεύω ότι τα βήματα που ακριβώ χρειαζόμαστε για να ενισχύσουμε τα φορολογικά έσοδα, να ενισχύσουμε την διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ διοικήσεων και εν τέλει να καταπολεμήσουμε την απάτη. Ευχαριστώ πολύ. εκ μέρους των Πρασίνων, ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. E Γιατί στοιχίζει ετησίως 5 δις ευρώ η φυγεί σε θέματα ΦΠΑ για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως όλο και περισσότεροι κάνουν αγορές διαδικτυακές και για αυτό θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ φορολογικών αρχών. Εξαιρετικά σημαντικό για μια ενιαία αγορά όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση όπου οι διασυνοριακές συναλλαγές είναι πάρα πολλέ. Θα πρέπει να είναι σωστά επανδρομένες οι ε, φορολογικές αρχές και σωστά καταρτισμένες και δεν συμβαίνει αυτό συχνά να αυτή η μεταρρύθμιση είναι μέρο σειρά μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση των κανόνων για το ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο δεν καλύπτεται από τη μεταρρύθμιση, αλλά θα πρέπει να το εξετάσει επισταμένω και επιγόντω η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η απαλλαγή ΦΠΑ στον τομέα τη αεροπλοεία. Δεν είναι λογικό να υπάρχει αυτή η απαλλαγή όταν να υφίστανται αυτή την υποχρέωση άλλη κλάδη τη οικονομία, πόσο μάλλον σήμερα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει πράσινη συμφωνία και πρέπει να τηρήσει τι δεσμεύσει που έχει αναλάβει για τη διάσκεψη των μερών για την καταπολέμηση πολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ εκ μέρους του ID. Για δύο λεπτά ο κύριος Μπέκ παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η απάτη ΦΠΑ είναι πράγματι ένα πρόβλημα, αλλά η Κομισιόν εδώ πέρα προτείνει μόνο ψεύτικες λύσεις και μια συνταγή για περαιτέρω μεγιστοποίηση των φορών και παρακολούθηση. Έχουμε λοιπόν υστέρηση των προσδοκόμενων φορολογικών εσόδων. Γιατί λέει από κάθε πολίτη θα πρέπει η Κομισιόν να παίρνει 262 ευρώ κάθε χρόνο. Είναι δικαιολογημένο αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τον υψηλότερο φόρο κατανάλωσης στον κόσμο. Κατά μέσο όρο οι Ευρωπαίοι πολίτες πληρώνουν πάνω από το διπλό από πολίτες άλλων χωρών. Σε σύγκριση με την Ιαπωνία ή με τον Καναδά πληρώνουμε τριπλάσιο και τετραπλάσιο και στη φορολογία εισοδήματος και στις κοινωνικές δαπάνες είμαστε κορυφή. Πουθενά αλλού δεν έχει το κράτος το χέρι του τόσο βαθιά σε τόσες πολλές τσέπες όσο στην Ευρώπη. Άρα θα περιμέναμε να περνάνε πολυτελώς οι πολίτες από τον υπεργογείο μέχρι τον τάφο με όλα τα ενδιάμεσα και τις υψηλότερες συντάξεις. Στην πράξη όμως μειώνονται οι συντάξεις, έχουν παγώσει οι πραγματικοί μισθοί, αυξάνεται η χρέωση και η οικονομία έχει πέσει σε τέλμα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις πρέπει να είναι ειλικρινείς επιτέλους. Χρειάζονται όλο και περισσότερα λεφτά για να χρηματοδοτήσουν την τις φαντασίες τους περί πολυπολιτισμού, ΛΟΑΤΚΙ και κοσμοδιορθωτισμού. Και συνεχώς υπονομεύουν την οικονομία με νέους φόρους και ζητούν όλο και περισσότερη επιτήρηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει περισσότερους φόρους και λιγότερη δημοκρατία. Οι πολίτες όμως θέλουν το αντίθετο. Τώρα, για τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές για 1,5 λεπτό ο κύριος Γιουριζίτσα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή, η ΦΠΑ, είναι από τα χειρότερα ε, από τις χειρότερες μορφές 137 εκατομμύρια ευρώ χάνονται κάθε χρόνο. Είναι τεράστια τα νούμερα αυτά, είναι τρομακτικά. Και θα έλεγα ότι αυτό βλάπτει την ευρωπαϊκή οικονομία αλλά βλάπτει και τους Ευρωπαίους πολίτες. Οι πιο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες είναι αυτές που υφίστανται και το μεγαλύτερο κόστος από λόγω αυτής της φοροδιαφυγής. Μπορεί να δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν δούμε τη γραφική παράσταση που έχω φέρει εδώ για να σας δείξω, βλέπουμε το χάσμα που υπάρχει σε σχέση με το πόσο πολλοί ΦΠΑ καταφέρνουν να εισπράξουν οι χώρες μέλη. Οι χώρες που έχουν τις καλύτερες επιδόσεις είναι το Λουξεμβούργο και η Κύπρος. Βλέπουμε όμως ότι το ποσοστό είναι 1%. Όμως αυτός που είναι πολύ μακριά είναι στο 30%, πέντε φορές πιο μακριά από τη δυνατότητα ίσπραξης. Βλέπετε λοιπόν τα διαφορετικά ε, ποσοστά. Θα πρέπει να γίνει μια ανάλυση ποιότητας και να είμαστε σε θέση στη συνέχεια να υιοθετήσουμε τις σωστές αποφάσεις με βάση τα περιστατικά και όχι με βάση τις εικασίες και τις γνώμες ή ε, το πώς διάκειται συναισθηματικά, αν θέλετε, ο καθένας εναντί αυτού και να εφαρμοστούν οι βέλτιστες πρακτικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ εκ μέρους της ε, ΓΚΟΕ της Ευρωπαϊκής Ενωμένης Αριστεράς. Για δύο λεπτά το λόγο έχει ο Αντιπρόεδρος κ. Παπαδημούλης. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Τζεντιλόνη, σας καλωσορίζουμε στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο είναι η πρώτη σας παρουσία εδώ αλλά επειδή μιλάμε για μια μεγάλης έκτασης φορολογική απάτη και φοροδιαφυγή αυτό που ζητά το ευρωκοινοβούλιο από την κομισιόν είναι να ανεβάσετε ταχύτητα στην αποτελεσματικότητα για τον περιορισμό αυτής της εκτεταμένης φορολογικής απάτης. Τα μεγέθη είναι τρομακτικά πολύ μεγάλα 137 δισεκατομμύρια το χρόνο τα υπολογίζετε εσείς στην Κομισιόν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή η φορολογική απάτη φορτώνεται στην πλάτη των συνεπών και των έντιμων φορολογούμενων, οδηγεί σε περικοπές του κοινωνικού κράτους και παραβιάζει και τον δίκαιο ανταγωνισμό ανάμεσα στις επιχειρήσεις γιατί ευνοούνται οι απατεώνες και τιμωρούνται οι συνεπείς. Για να αντιμετωπιστεί αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συνεργασία, αποτελεσματικότερη ελεγκτική μηχανισμοί, βαρύτερες κυρώσεις προς τους παραβάτες. Χρειάζεται περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη. Και για να γίνει αυτό χρειάζονται και νόμοι και κανονισμοί αλλά και χρήματα και θα ήθελα να καυτηριάσω την απουσία του συμβουλίου γιατί το κοινοβούλιο ζητάει πράγματα η κομισιόν τα υπόσχεται αλλά το συμβούλιο είναι απόν και επιπλέον η φιλανδική προεδρία στην πρόσφατη πρότασή της για το νέο πολιετή προϋπολογισμό προτείνει περικοπή των κονδυλίων για το πρόγραμμα συνεργασίας για την αντιμετώπιση της φορολογικής απάτης κατά 40% αυτού που προτείνει το Κοινοβούλιο και κατά 20% αυτό που είχαμε στο προηγούμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Επομένως κοροϊδευόμαστε. Δεν αρκούν τα λόγια, χρειάζονται έργα και αποτελέσματα. Thank you very much uh, ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τους μη εγγεγραμμένους για 1,5 λεπτό ο κύριος Overhart στην συζήτηση αυτή οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση για το ΦΠΑ θα επηρεάσει την εμπορική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Την Πέμπτη ο λαό του Ηνωμένου Βασιλείου ψήφισε συντριπτικά υπέρ του Brexit και μια συμφωνία τύπου Καναδά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης καταψήφισε την Τελωνιακή Ένωση, καταψήφισε την ενιαία αγορά και καταψήφισε οποιαδήποτε αρμοδιότητα του ΔΕΚ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όλοι συμφώνησαν ότι οι εκλογές αυτές αφορούσαν το Brexit. Οπότε για δεύτερη φορά μίλησε ο λαός για το θέμα αυτό. Και πάλι λοιπόν μας είπε ο λαός ότι ήξερε τι ψήφισε το 2016. Οι εκλογές αυτές έχει αποδείξει ότι όταν δοθεί η επιλογή, οι Βρετανοί επιλέγουν το ελεύθερο εμπόριο και τη συνεργασία και όχι ένα πολιτικό υπερκράτος οι υπόλοιποι πολίτες τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν ποτέ αυτή την επιλογή ή θα συνεχίσουν να πορεύονται προ τι Ηνωμένε Πολιτείε τη Ευρώπη. Οι πολίτε τη Ευρώπη θα πρέπει να έχουν την επιλογή. Και αν επιλέξουν, όπω οι Βρετανοί, που σταμάτησαν τον φεντεραλισμό να συνεχίσουν να συνεργάζονται ω εθνοκρατή. Λέγεται δημοκρατία, μπορεί να σας φαίνεται περίεργο, αλλά δεν συμφωνούν όλοι με την συγκεντρωτική μονολυθική πολιτική σας. Κάποιοι από εμά πιστεύουμε στη δημοκρατία. Όπως είπε και ο Ραβίνος Σάξ, ο κάθε ένα μετράει. Ο κάθε ένας μας έχει φωνή. Αν το χάσει αυτό, χάνει τα πάντα. Γιατί τότε γίνεται παιχνίδι των πλούσιων και ισχυρών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για δύο λεπτά ο κύριος Αρία Σετσεβερία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κυρία Εισηγήτρια, όλα τα κράτη-μέλη βιώνουν αυτό το πρόβλημα της φοροαποφυγής κατά τη διάρκεια των συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, χάνονται εις πράξεις ΦΠΑ 5 δις ευρώ σε ό,τι έχει να κάνει με τις διασυνοριακές συναλλαγές και υπάρχει φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή κατά την παροχή υπηρεσιών και η ποσοτικοποίηση ε, του ύψους αυτής της φοροδιαφυγής είναι πολύ πιο δύσκολη. Οι φορολογικές αρχές δεν έχουν απαραίτητα στοιχεία, ε, τις απαραίτητες πληροφορίες για να εφαρμόσουν σωστά τους κανόνες ΦΠΑ. Η ανταλλαγή των στοιχείων και δεδομένων δεν είναι πάντοτε εφικτή και για λόγους ε, νομικούς. Υπάρχουν νομικοί περιορισμοί και γι' αυτό η διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατικών αρχών κρίνεται ανεπαρκή αυτόν τον αγώνα καταπολέμησης της διαφυγή στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Χρειαζόμαστε νέα εργαλεία για να μπορέσουμε να σταθούμε στο ύψο των περιστάσεων. Χρειαζόμαστε περισσότερη ανταλλαγή πληροφοριών, μεγαλύτερη ευελιξία κατά τη λήψη των αποφάσεων και απλούστευση των κανόνων. Αυτά είναι ζωτική σημασία για να καταπολεμήσουμε την φόρο διαφυγή και φόρο αποφυγή με αποτελεσματικό τρόπο. Στηρίζουμε την πρόταση δημιουργία κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματο αποθήκευση ε, στοιχείων για τι συγκεκριμένε πληρωμέ δομές και υποχρέωση ε, των ε, Ιδρυμάτων των Χρηματοπιστωτικών να παρέχουν αυτές τις πληροφορίες στις φορολογικές αρχές. Είναι απαραίτητη η απλούστευση ε, και η εναρμόνιση της διαδικασίας συγκέντρωσης των δεδομένων και απλούστευση της μορφής με την οποία θα τηρούνται όλα αυτά τα στοιχεία και δεδομένα. Και έτσι θα πρέπει οι αρμόδιοι να μην παρουσιάζουν πια την ίδια πληροφόρηση με διαφορετική μορφή σε κάθε κράτος μέλος, αλλά να υπάρχει ομοιομορφία. Θα είναι πιο εύκολη η αναζήτηση των ε, στοιχείων και θα είναι πιο αποτελεσματική η δράση. Θα εξοικονομήσουν όλοι ε, και χρόνο και πόρους και θα ε, καταπέσουν ακόμα περισσότερα εμπόδια ε, που ε, δεν μας έχουν επιτρέψει ακόμα να φτάσουμε σε μια πραγματική ενιαία ψηφιακή αγορά. Αυτό είναι το πνεύμα που θα πρέπει να διέπει την εργασία μας και σας καλώ όλους να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Μπέλκα παρακαλώ. Από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Κύριε Πρόεδρε, Μιλούμε για ένα φόρο που αποτελεί πολύ σημαντική πηγή εσόδων για τα κράτη-μέλη. Η καταπολέμηση των απολειών ΦΠΑ είναι προσπάθεια να μειωθεί ο αντίκτυπο στον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι ένας αγώνας που δίνουν οι κυβερνήσεις για να χρηματοδοτήσουν τα νοσοκομεία, τα σχολεία ε, και για τις επενδύσει σε έργα υποδομών. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, η απόκληση αυτή ε, ανέρχεται σε 137 δις ευρώ 260 ευρώ ανά Ευρωπαίο πολίτη χάθηκαν. Απόκληση μεταξύ του ΦΠΑ που εισπράχθηκε και αυτού που θα έπρεπε να είχε εισπραχθεί δηλαδή. Ε, νομίζω ότι ο αγώνας πρέπει να είναι ενιαίος και ολομέτωπος. Ε, μια κοινή σειρά δράσεων θα καταφέρει να επιλύσει το πρόβλημα ή τουλάχιστον να το ελαχιστοποιήσει. Να μην ε, δίνει κάθε χώρα το δικό της αγώνα ξεχωριστά. Χαίρομαι με τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις και προαπαιτούμενα για όσους παρέχουν αυτά τα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών και διάφορα άλλα μέτρα. Επιτρέψτε μου όμως να θίξω δύο ζητήματα σημαντικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει και τις πλατφόρμες ψηφιακών νομισμάτων και το κατά πόσο θα πρέπει και αυτές να καλύπτονται και να υπάγονται στη σχετική νομοθεσία για να έχουμε πιο ακριβή στοιχεία για την απόκληση μεταξύ εισπραχθέντος και ε, ΦΠΑ και αυτού που θα έπρεπε να είχε εισπραχθεί ε, καλό να υιοθετήσουμε μια πιο στατιστική προσέγγιση για να μπορέσουμε να ποσοτικοποιήσουμε με ακρίβεια το φαινόμενο αυτό. Ευχαριστώ ο κύριος Ρονίτσα για 1,5 λεπτό από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, η κλίμακα της εν είναι τεράστια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανείς δεν ξέρει τις πραγματικές της διαστάσεις. Χρειάζεται συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Εμείς υποστηρίζουμε την Κομισιόν και το Συμβούλιο στον αγώνα αυτών, στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και φοροποφυγής στον χώρο του ΦΠΑ και δι στις ψηφιακές συναλλαγές. Φαίνεται ότι πρέπει να εφεύρουμε νέα εργαλεία, νέους τρόπους αντιμετώπισης για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο χωρίς φυσικά να θέσουμε σε κίνδυνο την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πρέπει να πάρουμε πληροφορίες για τις συναλλαγές των παραβατικών επιχειρήσεων όπου και αν βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε τρίτες χώρες. Η Πολωνία, πρέπει να σας πω, τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ αποτελεσματική στην προσπάθεια αυτή, καταπολεμώντας την φορολογική απάτη. Μπορούμε λοιπόν να είμαστε αποτελεσματικοί με τη συνεργασία όλων των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ένα λεπτό, ο κ. Μορέλ από την ΚΟΕ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είναι αληθές ότι η παγκοσμιοποίηση και η αποϊλοποίηση των αγορών οδήγησαν στην ανάδυση διαφόρων ειδών απαταιώνων που κάνουν μαζικές απάτες ε, σε επίπεδο ΦΠΑ, όπου η απόκληση αυτού που θα έπρεπε να εισπράττουμε και αυτό που εισπράττουμε ανέρχεται σε 137 δις ευρώ. 12 δις ευρώ είναι το, ε, αυτό που μας αναλογεί στη Γαλλία. Τρεις φορές το έλλειμμα δηλαδή στο συνταξιδοτικό καθεστώς στη Γαλλία. Μιλούμε για κολοσσία νούμερα για αστρονομικά ποσά. Ο συντονισμός είναι ανεπαρκής μεταξύ των κρατικών αρχών και οι φορολογικές αρχές δεν είναι ε, πολύ προσεκτικές. Όλα αυτά είναι αληθινά. Όμως υπάρχουν και αληθινοί ένοχοι. Μιλούμε για συστήματα διαδικτυακής πληρωμής, αλλά πρέπει να τονίσουμε όλες αυτές τις πλατφόρμες πωλήσεων, το Alibaba, το Amazon. Όλοι αυτοί είναι εκτός του δικού μας προβληματισμού, κανείς δεν τους ενοχλεί, μπορούν να κάθεκτη να εμπορεύονται προϊόντα τα οποία δεν υπόκειται σε ΦΠΑ. Στη Γαλλία 98% των αγαθών που περνάνε από το Amazon δεν ε, υπάρχει επιβολή ΦΠΑ. Πρέπει λοιπόν ε, να ε, τους δώσουμε την απάντηση που τους αξίζει και τους αναλογεί. Δεν πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέπει σε αυτές τις να μην πληρώνουν φόρο ενώ το οφείλουν. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής για 1,5 λεπτό, ο κύριος Σίντσετς. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλάμε για την ε, φορολογική απάτη και όταν μιλάμε για αυτά τα θέματα στην Κροατία πρέπει να αναφέρουμε την Algocor, μια μεγάλη επιχείρηση η οποία χρεοκόπησε πριν από δύο χρόνια. Η μεγαλύτερη επιχείρηση στην περιοχή αυτή της Ευρώπης με περίπου 60.000 εργαζόμενους. Και το παράδειγμα αυτό μας έδειξε πως έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην ε, Κροατία, ούτε κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό τα λέω από όταν μπήκα στην πολιτική. Δηλαδή άμα ξέρει κάποιο ε, κάποιο, ε, κάνει ό,τι θέλει και δεν τον αγγίζει κανείς. Έχουμε ε, περί τους 600 μεγάλους φορολογούμενους στην Κροατία. Και σε 146 από αυτές τις 600 μεγαλύτερες επιχειρήσεις δεν έχει πατήσει ποτέ η εφορία μεταξύ των οποίων και η Αλγκοκόρ. Ποτέ δεν έχει γίνει έλεγχος ε, σε σχέση με διάφορες ε, φορολογικές ε, παραδιάσεις και σε 170 από αυτές τις επιχειρήσεις δεν έχουν ελέγξει ποτέ το ΦΠΑ. Δηλαδή θεωρητικά στους νόμους υπάρχει ΦΠΑ, αλλά στην πράξη ποτέ δεν έχει εφαρμοστεί. Οι ιδιοκτήτες της Αλγκοκόρ έκαναν ό,τι ήθελαν, το αφεντικό συγκεκριμένα χρησιμοποιούσε διάφορα χρηματοπιστωτικά μέσα εμφανιζόταν να έχει λεφτά που, κεφάλαια που δεν ε, έχει και τελικά αποδείχθηκε η Κροατία Ελντοράντο και άγρια δύση της ε, φοροδιαφυγής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για δύο λεπτά κύριο Στεφανέτς. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι πεπισμένος ότι η αντιμετώπιση τη απάτης πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για όλους μας. Η αγορά παγκοσμιοποιείται, ψηφιοποιείται, κάτι το οποίο φέρει οικονομίες, όμως ε, είναι πεδίο δόξης λαμπρών για τους εγκληματίες τα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διαθεσή μας είναι όλο και λιγότερα για να αντιμετωπίσουμε την απάτη. Και όλα αυτά ισχύουν και για τον ε, τομέα του ΦΠΑ που κάθε χρόνο χάνουμε 137 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία θα έπρεπε να περιέλθουν στις τσέπες της εφορίας και ανταυτού περιέχονται στις τσέπες της μαφίας. Ποιοι είναι οι χαμένοι? Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αυτά είναι τα πραγματικά περιστατικά. Εξού και οι δολοφονίες δημοσιογράφων που διερεύνησαν το φαινόμενο στη Μάλτα και στην Σλοβακία. Έχει λοιπόν τεράστια σημασία οι αρχές των κρατών μελών να ανταλλάσσουν πληροφορίε στο μέγιστο δυνατό βαθμό, να τις αξιοποιούν και να τις χρησιμοποιούν και για την προσαγωγή των υπευθύνων ενώπιον της δικαιοσύνης. Μην ξεχνάτε επίση ότι τα κρυπτονομίσματα διευκολύνουν ε, την την φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Και εδώ πρέπει τα κράτη-μέλη να ασχοληθούν σοβαρά με αυτές τις νέες ελλαγέ, ενημερώνοντας την νομοθεσία και ενδύνοντας τη συνεργασία τους. Μπορούμε λοιπόν να τα πάμε καλύτερα σε όλους αυτούς τους τομείς. Ελπίζω λοιπόν ότι η νέα Κομισιόν θα εντοπίσει όλε αυτέ τι αδυναμίε και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κατορθώσει να μειώσει τι απώλειε στα φορολογικά έσοδα. Από την πλευρά μα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να πλουστεύσουμε το φορολογικό σύστημα και όπω είπα να δώσουμε τη μάχη μαζί κατά αυτών που καταχρώνται του συστήματο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγο στον κύριο Κούσμιουκ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπέ, 140 δισεκατομμύρια ευρώ το έτος είναι το εισπρακτικό έλλειμμα του ΦΠΑ. Σχεδόν ίσο με τον ετήσιο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς η κατάσταση διαφέρει από κράτος σε κράτος. Η Πολωνία κατάφερε να μειώσει αυτό το εισπρακτικό έλλειμμα από το 24% στο 12% το 2018. Και αυτή τη χρονιά το έλλειμμα θα πέσει στο 10%. Ελπίζω ότι και άλλα κράτη-μέλη θα πάρουν την Πολωνία για μοντέλο. Η οδηγία αυτή προφανώς ανταποκρίνεται στο κέλευσμα των καιρών. Ο ρόλος των ηλεκτρονικών πλατφορμών έχου, έχει αυξηθεί, αυξάνεται το ηλεκτρικό εμπόριο, αλλά αυτό καθιστά ακόμα πιο δύσκολο το έργο των φορολογικών αρχών. γίνεται όλο και πιο δύσκολη η καταπολέμηση τη φορολογική απάτη. Η πρόταση που προβλέπει ανταλλαγή πληροφοριών, προβλέπει την ε, δημιουργία ενός κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος έχει και αποτελεί πλεονέκτημα για όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ο λόγος του κύριο Μάντερς για δύο λεπτά. Δεν είναι εδώ. Μετά ο, ο λόγος του κύριου Μπουξαντέ Βιγιάλβα. Για ένα λεπτό. Ούτε ο ίδιος είναι εδώ. Κυρία Ταλέχ. Για δύο λεπτά. Κυρία, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητό κροακτήριο, στις οθόνες μας μπρά στις οθόνες, μιλώ σαν βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σήμερα ως επιχειρηματίας ε, IT. Ακούσαμε το 2017 ε, το, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο, υπήρξε ένα τεράστιο έλλειμμα του ΦΠΑ, ε, ένα έβδομο του πολιτισμού δημοσιονομικού πλαισίου ή το ίδιο ποσό το οποίο δώσαμε για τον, ε, την ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό. Αυτό καθιστά σαφές το πόσο κατεπηγόντως θα πρέπει να δημιουργηθούν κάποιοι κανόνες ούτως ώστε να αποτρέψουμε αυτές τις απάτες με το ΦΠΑ. Ένας άλλος ε, λόγος αύξησης του ελλείμματος είναι η αύξηση της απάτης στο ηλεκτρονικό εμπόδιο. Αλλά οι, οι χώρες μεμονωμένες δεν έχουν τη δυνατότητα να ε, ανταπεξέλθουν γιατί δεν διαθέτουν τα, τις πληροφορίες. Με την πρόταση αυτή, οι χώρε μέλη έχουν ένα αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια του, ώστε να δημιουργήσουν θεμητού όρου ε, ανταγωνισμού για το ηλεκτρονικό εμπόριο και για τη διεξαγωγή ελέγχων. Με τον τρόπο αυτό θα αποστείλουμε ένα θετικό σήμα προ όλε τι ε, μικρομεσαίε επιχειρήσει που φέρνουν το μεγαλύτερο βάρο στι ε, πλάτε του. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα, ξεκινήσουμε, θα συνεχίσουμε με, το, με τη διαδικασία Catch the Eye για ένα λεπτό. Η κυρία Γραπίνη. ευχαριστώ πολύ κύριε, ε, Επίτρο, κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ε, πραγματικά αισθάνομαι μεγάλη εμπιστοσύνη γιατί ε, συζητήσαμε το θέμα αυτό και στην προηγούμενη θητεία. πρέπει να προσπαθήσουμε μαζί να βρούμε τα εργαλεία τα οποία θα μας δώσουν τη δυνατότητα να καταπολεμήσουμε αυτή την πληγή. Υπάρχει ας πούμε το εργαλείο Eurofisk μέσω του οποίου ανταλλάσσουν πληροφορία στα κράτη-μέλη. Δυστυχώς όμως υπάρχει υπάρχει ακόμα ε, ε, μεγάλη ε, απάτη όσον αφορά το διασυνοριακό ΦΠΑ. Επίσης γίνονται και εικονικές πληρωμές και εικονικά τιμολόγια. Πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε την κατάσταση αυτή. Πρόκειται για μεγάλη πληγή. Και εδώ μιλάμε για οργανωμένο οικονομικό έγκλημα και επομένως θα πρέπει να βρούμε άλλα εργαλεία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Το 2016 250 δις ήταν ε, ε, η φοροδιαφυγή. Πρέπει, μειώθηκε λίγο το ποσό αυτό, αλλά πρέπει να μειωθεί κι άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό κύριος Μποτός. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, συμφωνώ απολύτως ε, μαζί σας. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα κεντρικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών και όλα τα κράτη-μέλη να ενταχθούν στο σύστημα αυτό έτσι ώστε τα δεδομένα να εισάγονται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Υπάρχουν όμως χώρες-μέλη που δεν έχουν την διοικητική και οικονομική <clears throat> τεχνική ικανότητα να βάζουν σε πραγματικό χρόνο ε, αυτά τα στοιχεία στο σύστημα και ούτε έχουν την δυνατότητα ε, να προσαρμόζονται τόσο γρήγορα ε, στις τεχνολογικές εξελίξεις. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές λοιπόν να αποκτήσουν αυτές τις τεχνικές ικανότητες. Επίσης θα πρέπει να βρούμε ένα τρόπο έτσι ώστε το κεντρικό σύστημα να ενημερώνεται πιο γρήγορα και να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ για ένα λεπτό ο κύριος Τσιχοντάρου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Τζεντιλόνι, πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ ανήσυχος. Για πρώτη φορά ε, έρχομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως εκλεγμένος και ε, με ανησυχία ακούω αυτά που ε, λέτε όσον αφορά την, τα χρήματα της Ευρώπης. Πρόκειται για χρήματα τα οποία δεν πρέπει να δαπανώνται με οποιοδήποτε τρόπο. Ναι, φυσικά χρειάζεται ένα κεντρικό κεντρικό ε, σύστημα, αλλά και αυτό δεν είναι εύκολο. Μήπως θα πρέπει αντιθέτως να κάνουμε προληπτική ε, φορολογική ε, πολιτική στις χώρες μέλη. Νομίζω ότι όταν μιλάμε για τόσο μεγάλα ποσά θα πρέπει πραγματικά να κινηθούμε αποτελεσματικά. Ενδεχομένως και η νέα Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να αναλάβει ρόλο, να επιβάλλει κυρώσεις έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η κατάσταση ε, ευχαριστώ κύριε Τζεντιλόνη για όσα μας είπατε και πραγματικά δεν θα ήθελα καθόλου να είμαι στη θέση σας. Σας ευχαριστώ και τώρα θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο ε, Τζεντιλόνη. Παρακαλώ κύριε Τζεντιλόνη έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την ποιότητα της συζήτησης εδώ και επίσης για την βρία ε, υποστήριξη προς τις ε, προτάσεις που συζητούμε εδώ. Έχω δύο μόνο παρατηρήσεις να κάνω. Η πρώτη είναι η εξής. Όπως, είπατε, όπως είπαν πολλοί από εσά, η διοικητική συνεργασία ε, θα διευκολύνει πάρα πολύ αυτή τη διαδικασία. Οι φορολογικές αρχές και χώρες μέλη θα πρέπει να κάνουν πλήρη χρήση των ε, εργαλείων, των νέων εργαλείων που υπάρχουν. Ε, δεύτερον, προφανώς ε, θα πρέπει να γίνουν περισσότερα πιο φιλόδοξα βήματα προς τα μπρος, λόγω ακριβώς ε, της διάστασης του προβλήματος το οποίο αντιμετωπίζουμε εδώ. Θα δουλέψουμε χέρι με χέρι, στενά συνεργαζόμενοι και η Επιτροπή θα διοργανώσει ένα συνέδριο προκειμένου να συζητήσουμε το πώς θα πετύχουμε φορολογική συμβατότητα, φορολογική εναρμόνιση και καταπολέμηση της φορολογικής απάτης. Ελπίζω, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι η δική σας εισφορά στο συνέδριο αυτό θα είναι πολύτιμη γιατί από αυτή την ε, ε, συνδιάσκεψη θα καταλήξουμε σε κάποια μέσα πολέμης της απάτης και ε, τρόπους εξασφάλισης της φορολογικής εναρμόνισης. Είμαι σίγουρος ότι το Κοινοβούλιο θα εισφέρει σε αυτή τη διαδικασία. Μπορείτε να υπολογίσετε στη δική μου δέσμευση να συμβάλλω επίσης στην κατεύθυνση αυτή ε, της χάραξης μιας ε, σωστής φορολογικής ε, πολιτικής. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Και τώρα τελευταία μιλήτρια είναι η κυρία Περέιρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεισφορά σας δείχνει ότι ε, είμαστε προσιλωμένοι στην καταπολέμηση της ε, απάτης σχετικής με τον ΦΠΑ. Νομίζω ότι η φιλοδοξία μας είναι ε, δικαιολογημένη και το πρόβλημα είναι σημαντικό. Αυτή τη στιγμή το νομοθετήν δεν σημαίνει γενικές και αόριστε λύσεις, αλλά συγκεκριμένε λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα όταν υπάρχει επιβάρυνση στους προπολισμού και στον κόσμο. Ε, η ε, απάτη του ΦΠΑ επηρεάζει και τις οικογένειες και τα δημόσια κρατικά οικονομικά. Το ηλεκτρονικό εμπόριο διαρκώ αυξάνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα αυξάνεται και η κίνδυνη η προστασία της εσωτερική αγοράς μερικές φορές σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε και να αφήσουμε την αγορά να λειτουργήσει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως δεν είναι αλήθεια αυτό. Χρειαζόμαστε μια δίκαιη αγορά και η φορολόγηση αποτελεί εργαλείο απονομής δικαιοσύνης. Οι εκθέσει αυτέ αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο και το ΦΠΑ, αλλά θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα μήνυμα για μια πιο ευρεία μεταρρύθμιση του ΦΠΑ σε όλη την Ευρώπη. Έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια φορολόγηση που είναι πιο πολύ προσανατολισμένη στην ψηφιακή εποχή. Θα βοηθήσει αυτό τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συν, ε, την ε, συνοχή ε, και τα νοικοκυριά. Η, το, η πρόκλησή μας είναι να αυτά τα προβλήματα να τα ε, τους δώσουμε να τα, αντιμετωπίσουμε έτσι ώστε να αυξηθεί η απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λίγη η κοινή ψηφοφορία, η, ψηφοφορία θα, η κοινή συζήτηση, η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Περνάμε στην επόμενη κοινή συζήτηση για το διορισμό μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δύο εκθέσεις της κυρίας για το διορισμό δύο μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί και η μπλε κάρτα και να ζητήσετε το λόγο στη διαδικασία του Catch the Eye. Ε, αν θέλετε να δείτε οδηγίες για το πώς να το, τα κάνετε αυτά, υπάρχουν στην είσοδο της αίθουσας. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Τινάλη. Thank Σα Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Με αυτές τις δύο εκθέσεις που θα ψηφιστούν αύριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει μια μη δεσμευτική γνώμη όσον αφορά το διορισμό νέο, δύο νέων μιλών ε, της Εκτελεστικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής ε, ε, Κεντρικής Τράπεζας. Η αφορά τα δύο ονόματα, δηλαδή την Ιζαμπέλ Σναμπέλ, καθώς επίσης και τον Φάμπιο Πανέτα. Είναι γεγονός ότι ο πρόεδρος του Συμβουλίου ε, καταδεικνύει ότι τα δύο αυτά άτομα ε, ε, είναι άτομα εγνωσμένου κύρους όσον αφορά τον τομέα τους και καλύπτουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 283 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Φάβιο Πανέτα έχει λάβει πολλές θέσεις σε ευρωπαϊκό, ιταλικό και διεθνές επίπεδο και έχει υπάρξει και επικεφαλής της ε, ε, ε, Ιταλικής Κεντρικής Τράπεζας. Η κυρία Σνάμπελ για πέντε χρόνια ήταν μέλος του Γερμανικού Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων μεταξύ άλλων. Επίσης έχουν οργανωθεί όσον αφορά τους δύο διορισμούς ε, ακροάσεις ε, επίσης ε, έχουν απαντήσει στις ερωτήσεις που τους είχαν υποβληθεί και με πολύ καλή επίδοση. Ωστόσο και παρά το γεγονός ότι εμείς υποστηρίζουμε τους διορισμούς του Φάβιο Πανέτα και της Ιζαμπέλ Σνάμπελ δεν πρέπει να λησμονούμε τα εξής η ε, διαδικασία για την επιλογή ε, των υποψηφίων θα πρέπει να εμπλέκει πολύ περισσότερο ε, τον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μετά από δική μας επιμονή, ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, μας προώθησε τους φακέλους. Ωστόσο, θα πρέπει να επιμείνουμε ότι το Συμβούλιο πριν από οποιοδήποτε διορισμό θα πρέπει να υποβάλει ε, στο Κοινοβούλιο τουλάχιστον δύο υποψηφίους και τουλάχιστον έναν άντρα και μία γυναίκα για κάθε θέση. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε πραγματικά ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών στην διαδικασία επιλογής ε, και με τον τρόπο αυτό ε, να προωθήσουμε την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε διάφορα όργανα. Ε, πρόσφατα ανανεώθηκε το, το Συμβούλιο της ε, Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας ε, και μόνο δύο είναι γυναίκες. Βεβαίως δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η κυρία Λαγκάρντ έχει διοριστεί ως η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ωστόσο αυτό δεν είναι αρκετό. Το άλλο κυβερνών ε, όργανο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής ε, Τράπεζας άλλωστε έχει ε, ως εκπρόσωπο μονάχα μία γυναίκα, την ίδια την πρόεδρο, την κυρία Λαγκάρντ. Επίσης ε, και τα 19 μέλη ε, του, ε, της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που εκπροσωπούνται από τους διοικητές των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ είναι άνδρες. Θα πρέπει οπωσδήποτε να πιέσουμε το Συμβούλιο για να προωθήσει το μήνυμά μας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να πω ότι έχουμε εδώ δύο εξαιρετικές υποψηφιότητες ε, που οπωσδήποτε θα συμβάλλουν στην καλή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό όμως δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να μειώνει την αποφασιστικότητά μας να αγωνιστούμε για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φίλων στο μέλλον. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Επιτροπή. Κύριε Επίτροπε Τζεντιλόνι, έχετε το λόγο. Ε, thank you, Madam President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριε και κύριοι, κυρία Τινάλη. Γνωρίζουμε τη σημασία του ρόλου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την οικονομία μας η τράπεζα έπαιξε ένα κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση της πρόσφατης κρίσης. Η νομισματική της πολιτική απετέλεσε εργαλείο για την αναθέρμανση της οικονομίας και με αυτόν τον ε, τρόπο καταπολεμήθηκε ο κίνδυνος από πληθωρισμού. Χαίρομαι που συζητάτε αυτούς τους δύο διορισμούς, ιδιαίτερους αυτούς τους δύο διορισμούς, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί χρειάζεται ε, διαφάνεια. Η συνθήκη κατοχυρώνει την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι μια αρχή την οποία η Κομισιόν στηρίζει ολόθερμα. Η ανεξαρτησία και η λογοδοσία είναι όμως δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Δεύτερον, όπως βλέπετε από την σύνθεση του, της Κομισιόν και των πολιτικών γραφείων των Επιτρόπων, εγώ ίδιο μπορώ να σα πω ότι ε, είμαι προσιλωμένος στην ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Είμαι πεπισμένο ότι όργανα όπω η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν ιδιαίτερε ευθύνε σε αυτό. Συνεπώ στηρίζω το έργο, του, την προσπάθεια του Κοινοβουλίου να εξασφαλίσει ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων σε όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το υπογράμμισε και η κυρία Τινάλη. Όπως πολύ σωστά λέτε στην έκθεσή σας, όλοι όσοι εργάζονται στο οικονομικό κλάδο πρέπει να κάνουν κάτι παραπάνω προς αυτήν την κατεύθυνση. Όμως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να διευκολύνουμε την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πολύ δε περισσότερο που η ίδια τράπεζα δεν μπορεί να κατηγορηθεί για λάθη που έκαναν άλλοι στο, στις υποψηφιότητες και τους διορισμούς. Πάντως οι προσπάθειες έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσετε να... Ε, και, είμαι σίγουρος ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συνεχίσει να προσπαθεί να εξασφαλίσει όταν μεταξύ των δύο φίλων υπό την Προεδρία της κυρίας Λαγκάρτ. Μετά τον διοσμό της κυρίας ε, Λαγκάρτ και την εκλογή της Ursula von der Leyen ως Προέδρου της Κομισιόν δείχνει ότι φαίνεται ότι οι γυναίκες ε, έχουν ε, προσφέρει και θα προσφέρουν στις, σε μερικές από τις πιο σημαντικές θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσμένω σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ευχαριστώ. Εκ μέρους των πολιτικών ομάδων ξεκινάμε το ΕΛΚ και τον κύριο Φέρμπερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Εκτελεστική Επιτροπή τη ΕΚΤ ε, ζει μια καμπή. Η Κριστίν Λαγκάρτ μαζί με το Φάμπιο Πανέτα και την Ιζαμπέλ Σνάμπελ ε, είναι νέα πρόσωπα ε, σε αυτό τον οργανισμό. Και σίγουρα αυτή είναι μια ευκαιρία να αναθεωρηθούν κάποιες ε, προτεραιότητες της ε, ΕΚΤ. Για παράδειγμα, της ε, χρηματοπολιτικής στρατηγικής της ΕΚΤ, αλλά κατά την εξέταση αυτή θα πρέπει να μην θέσουμε υπερβολικά φιλόδοξους στόχους, γιατί η εντολή της ΕΚΤ ε, προέρχεται, απορρέει από τις ε, συνθήκες. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι στο περιεχόμενο της εντολής, θα πρέπει να αλλάξουμε τις ίδιες τις συνθήκες. Αυτό όμως το οποίο είναι εφικτό είναι να σκεφτούμε τι σημαίνει η σταθερότητα των τιμών στον 21ο αιώνα. Ο επικεφαλής της ΕΚΤ ανέφερε τους δομικούς παράγοντες, διαρθρωτικούς παράγοντες που επηρεάζουν ε, αυτή την πολιτική. Οι δημογραφικές μεταβολές, η αυξανόμενη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά προϊόντα. Ωστόσο, αν ευσταθεί αυτή η ανάλυση, η ΕΚΤ θα πρέπει να κάνει ένα βήμα παραπέρα. Αυτό σημαίνει όταν ε, ε, υπάρχει ε, μια τέτοια ισορροπία θα πρέπει να προσαρμόζεται εδώ και η ΕΚΤ. Δεν έχει κανένα νόημα να παραμένει προσιλωμένο στο στόχο του ανάπτυξη 2% εάν τα ποσοστά ανάπτυξη σύμφωνα με τις προγνώσεις του ίδιου του οργανισμού είναι χαμηλότερα. Ως ε, ΕΛΚ θα στηρίξουμε τις δύο αυτές ε, υποψηφιότητες και ε, αναμένουμε με ενδιαφέρον μια στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Thank you very much. Next speaker. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για δύο λεπτά, ο κύριος Φερνάντες παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Επιτροπέ. Αύριο θα ψηφίσουμε αυτές τις δύο υποψηφιότητες για να συμπληρώσουμε την Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και οι δύο υποψήφοι πληρούν τις απαιτήσει. Αυτό το ανέφερε και η Αρμόδια Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο διορισμός τους συνοδεύει τον διορισμό και της ε, κυρίας Λαγκάρντ. Ανοίγει μια καινούρια περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας θα πρέπει να ξαναδούμε τη δραστηριότητα της ΕΚΤ. Η εντολή η οποία έχει δοθεί στην ΕΚΤ είναι σαφώς καταχωρημένη στη συνθήκη. Όμως τι γίνεται ε, με την μετάφραση αυτή τη εντολή σε συγκεκριμένα μέτρα, σε συγκεκριμένη νομισματική πολιτική. Και εκεί χρειάζεται συζήτηση η στρατηγική, η νομισματική στρατηγική της Κεντρικής ε, Τράπεζας ε, συμφωνήθηκε το 2003, δηλαδή πριν από 15 περίπου χρόνια. Από τότε όμως έχουν αλλάξει πολλά. Έπεσε, έπεσαν τα επιτόκια ως ε, απάντηση στου, στις δημογραφικές αλλαγές και στην αύξηση της ψηφιοποίησης. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να βρούμε καινούριου στόχους μέσα στην ίδια εντολή. Πρέπει να αναλύσουμε το κατά πόσον μπορούμε να λαμβάνουμε υπόψη την τιμή των μετοχών και να ξαναδούμε επίσης το, τα καινούργια εργαλεία του ψηφιακού κόσμου, ψηφιακής εποχής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Πάντω η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα είναι έτοιμη γιατί και οι πρόεδρο και τα δύο αυτά καινούργια μέλη ε, είναι ικανά να φέρουν σε πέρα στο έργο του. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους του Renew Europe, ο κύριος Γκαρικάνο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήταν ε, το μόνο όργανο το οποίο εξ ονόματος όλων των Ευρωπαίων ανέλαβε να λύσει την κρίση. Δυστυχώς λαμβάνοντας υπόψη και τα νέα τα οποία μας φτάνουν από διάφορες ε, χώρες, ε, ε, δεν πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Άλλοι παραπονιούνται ότι έκανε υπερβολικά πολλά, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάνει πολλά, γιατί άλλωστε η νομισματική πολιτική είναι η μόνη η οποία άντεξε. Η νομισματική πολιτική όμως δεν μπορεί να είναι το μοναδικό εργαλείο καταπολέμησης της οικονομικής κρίσης. Ε, και ε, οπωσδήποτε θα πρέπει να έχουμε μια, ειδικό προϋπολογισμό για την ε, Ευρωζώνη που οπωσδήποτε θα πρέπει να είναι αρκετά, αρκετός και σημαντικός. Θα πρέπει επίσης να λέμε την αλήθεια όσο και αν αυτή δεν αρέσει. Πρέπει να γίνουν λοιπόν, και αυτή είναι η αλήθεια, πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα. Η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων έχει από αποδεχτεί τους διορισμούς των δύο ε, υποψηφίων, αλλά και με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να κάνει περισσότερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, για την Ευρωζώνη. Επίσης, ε, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μονάχα και τόσο πολύ να μιλάμε για την νομισματική πολιτική. Θα πρέπει οπωσδήποτε να καταπολεμηθεί η κακή επικοινωνία και ο νομισματικός λαϊκισμός θα χρειαζόμαστε μια Ευρωπαϊκή ε, Ένωση η οποία θα έχει ένα πολύ ξεκάθαρο αφήγημα και θα εξηγεί στους ε, πολίτες ε, γιατί οι κινήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ήταν απαραίτητες και εξακολουθούν να είναι απαραίτητες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει οπωσδήποτε με μεγάλη ενεργητικότητα να διαψεύσουμε τα λαϊκίστικα ψέματα, τα ψέματα των λαϊκιστών. Θα πρέπει να βασιστούμε στις ιδέες που ε, αποτελούν κίνητρο έτσι ώστε να πάρουμε τις αποφάσεις που παίρνουμε. Ε, και να μην λησμονούμε ότι όλες μας οι πράξεις θα πρέπει να έχουν σαν στόχο την επιβίωση ε, και του κοινού νομίσματος που αποτελεί άλλωστε ένα από τα μεγάλα μας επιτεύγματα. Οι δύο υποψήφοι, η Ζαμπέν Σαμέλ και ε, ο, κύριος Πενέτα, είναι δύο εξαιρετικοί υποψήφοι, τους οποίους η Ρινιού θεωρεί ικανούς υποψηφίους και επομένως θα τους υπερψηφίσει. Όπως ε, είπε προηγουμένως ε, και η συγγήτρια ε, και πρόεδρος της Επιτροπής μας, θα πρέπει οπωσδήποτε να ξαναδούμε τα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας και οπωσδήποτε να δούμε και το θέμα της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων. Δεν είναι δυνατόν στα 24 μέλη μονάχα να υπάρχει μία γυναίκα, ε, αυτό σημαίνει ότι δεν εκπροσωπείται ε, η ισόρροπα ε, ο πληθυσμός, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ έχουμε, ε, όπω είπαμε και προηγουμένω, πρέπει να υπάρχει υποχρέωση να υποβάλλονται ταυτόχρονα δύο υποψηφιότητε ενό άνδρα και μίας ε, γυναίκα. Είναι γεγονό από την άλλη πλευρά ότι ε, και από την πλευρά των κρατών μελών δεν υπάρχει ισόρροπη εκπροσώπηση. Όλοι οι επικεφαλεί των κεντρικών τραπεζών είναι άντρε Εγώ όμω, ω καθηγητή οικονομία, οι διοικητέ των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών είναι όλοι άντρε. Εγώ όμω ως καθηγητή Γνωρίζω πάρα πολλές γυναίκες ε, οι οποίες ασχολούνται με τα οικονομικά και οι οποίες είναι εξαιρετικά άξιες. Ε, αυτά ήθελα να πω. Σας ζητούμε λοιπόν από τα κράτη-μέλη να αλλάξουν τακτική. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρου των ε, Πρασίνων, για δυόμιση λεπτά έχει το λόγο ο κύριος Γκίγκολτ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εμείς οι πράσινοι υποστηρίζουμε την Ιζαμπέλ Σνάμπελ και τον Φάμπιο Πανέτα. Ωστόσο, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία αυτή εδώ για να επισημάνουμε το πώ έγιναν τα πράγματα. Εδώ και τέσσερα χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μάχεται ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των φύλων στι ε, κεντρικέ θέσει ε, των, μεγάλων ε, των μεγάλων οργανισμών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μέχρι στιγμή δεν το έχουμε πετύχει. Αυτό το οποίο εδώ έγινε είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπε ξεκάθαρα ότι μελλοντικά θέλουμε να υπάρχουν ισορροπίε ισορροπημένοι κατάλογοι υποψηφίων, ούτω ώστε να μπορούμε να παίρνουμε τις αποφάσεις ε, βάσει των ε, προσόντων και των δύο φύλων ε, και το Συμβούλιο και πάλι δεν τα κατάφερε γιατί συνεχίζουν οι ψηλές θέσει να δίδονται βάσει άλλων κριτηρίων μια φορά ένας Γερμανός, μια ένας Ιταλός κλπ. Με τον τρόπο αυτό δεν πληρούν τις ε, θέσεις ε, στελέχη με υψηλά προσόντα, ούτε επιτυγχάνεται η ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια ε, διεθνή συμφωνία, ούτω ώστε να μπορέσουμε μελλοντικά, χωρίς να ζημιώνουμε τους υποψηφίου, να μπορούμε να πετύχουμε αυτή την ισορροπία. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να προβεί σε μια τέτοια διοργανική συμφωνία όσον αφορά την επίτευξη ισορροπίας στα όργανα, στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ε εάν ήταν μια γυναίκα πρόεδρος της ε, ΕΚΤ, ε, ο κύριος Ντράγκη ε, καθόρισε για το μέλλον μια πολιτική χαμηλών επιτοκίων. Γι' αυτό θεωρώ ορθό το ότι είπε η νέα διευθύντρια ότι θα, θα αναθεωρήσουμε την, ε, ε, την στρατηγική της χρηματικής πολιτικής. Και θεωρώ ότι αυτή η απόφαση ήταν απολύτως ορθό, γιατί θα πρέπει να δούμε και τις αρνητικές συνέπειες των χαμηλών επιτοκίων γιατί ο κίνδυνος ε, να υπάρχουν μελλοντικά άλλε φούσκες είναι απολύτως ε, ρεαλιστικός. Ε, και όπως είπε η κυρία Λαγκάρντ, μόνο με μια κοινή νομισματική πολιτική, με μια ολοκλήρωση της νομισματικής, χρηματικής και τραπεζικής ένωσης, μπορούμε να αποφύγουμε μελλοντικά τέτοιου είδους φαινόμενα. Um- Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρινάλντι, δύο λεπτά. Ε, ε, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η αντιπροσωπεία μας έχει εκφραστεί ευνοϊκά όσον αφορά ε, το, δύο, το, όσον αφορά τον, το διορισμό του δόκτωρα Φάμπιο Πανέτα την Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καθότι έχει επιδείξει ανεξαρτησία, αμεροληψία ε, και ε, όλα τα στοιχεία τα οποία ε, αποτελούν απόδειξη αξίας όσο ή το διοικητής στην Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας. Θα ήθελα όμως να εκφράσω εδώ την ευχή το νέο, η νέα εκτελεστική επιτροπή ε, στο σύνολό, του, στο σύνολό της ε, να λάβει υπόψη τα πολύ χαμηλά ε, επιτόκια. Πρέπει να υπάρξουν νέα νομισματικά κίνητρα. Είναι γεγονός ότι υπήρξε ανάγκη πριν από μερικά χρόνια να ληφθούν έκτακτα μέτρα. Ωστόσο, αυτά τα μέτρα πλέον έχουν δημιουργήσει σημαντικότατα προβλήματα στο ενεργητικό, ειδικά δε στο επενδυτικό ενεργητικό ε, των ε, τραπεζών. Θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να ληφθεί υπόψη ένα calendar provisioning που θα λαμβάνει η υπόψη όλα τα στοιχεία τα οποία καθορίζονται ως level 2 και level 3 έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η εξυγίανση ε, των χρηματοπιστωτικών ε, ιδρυμάτων όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να λάβει υπόψη ε, και όλα τα στοιχεία τα οποία υποβάλλει η ΕΣΜΑ όσον αφορά την βιωσιμότητα ε, των Ιδρυμάτων στις χώρες μέλη και ε, να λάβει υπόψη και το, τον αντίκτυπο που έχουν τα μηδενικά επιτόκια στην τοποθέτηση των δημοσίων ομολόγων. Ε, ε, και ε, οπωσδήποτε να, ληφθεί υπόψη, να ληφθούν υπόψη όλα αυτά στην εφαρμογή της ποσοτικής μεθόδου. για την ομάδα ECR θα πάρει το λόγο για ένα λεπτό ο κύριος Βαν Οβερτεβέλτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα ήταν πολύ ακριβή στις πολιτικές τα τελευταία δέκα χρόνια. Υπήρχαν λόγοι βέβαια, αλλά σήμερα, ε, παρόλο που η κρίση έχει περάσει, εξακολουθούμε να επιμένουμε στην ίδια πολιτική. Πολιτική που έχει παρενέργειες. Για παράδειγμα, η απειλή των αποταμιεύσεων, η μείωση της ε, παραγωγικότητας γιατί όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ζόμπι κρατούνται ζωντανές και τρίτον γιατί υποσκάπτεται η χρηματοοικονομική σταθερότητα. Και η πρόεδρος και τα μέλη του, της Εκτελεστικής Επιτροπής θα πρέπει να το λάβουν υπόψη αυτό. Τα δύο, ε, οι δύο αυτοί υποψήφοι μας έκαναν πολύ καλή εντύπωση και θα τους υπερψηφίσουμε βέβαια. Να επιστρέψω όμως στο σχόλιο της κυρίας Σνάπελ που κατά τη διάρκεια της ε, ακρόασης είναι ελάχιστοι αυτοί που πραγματικά καταλαβαίνουν τι σημαίνει, είπε. Ε, είπε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε τα ανακοινοθέντα της ε, Κεντρικής Τράπεζας να είναι πιο κολονόητα, ευνόητα από τους πολίτες. Ε, χαίρομαι γι' αυτό, ευχαριστώ. Ε, ωραία. Περνάμε στην ΚΟΕ. Ο λόγος στον κύριο Γκουσμάου. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά τη διάρκεια της θητείας του κύριου Ντράγκη κινητοποιήθηκαν ε, έκτακτα μέτρα νομισματικής πολιτικής όμως ε, η, παρόλα αυτά η ανάπτυξη ήταν πολύ περιορισμένη, ενώ αυτά τα όργανα, τα εργαλεία δημιουργούν κινδύνους και απειλές για το μέλλον, που δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Θα θέλαμε, αν οι υποψήφοι συμφωνούν με την ανάγκη να έχουμε μια, ένα μείγμα πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με πολύ πιο σημαντικά δημοσιονομικά εργαλεία, Θέλουμε να ξέρουμε τι πιστεύουν για το κατά πόσον η ΕΚΤ θα πρέπει να αντιμετωπίσει περισσότερο το θέμα των ανισοτήτων και της α, ε, ε, ανεργίας, ε, ξεχνώντας λίγο το θέμα του πληθωρισμού και πώς μπορεί η ΕΚΤ να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αυτά ρωτήσαμε κατά τη διάρκεια της ακρόασης. Οι απαντήσεις του κυρίου Πανέτα ήταν ικανοποιητικές, γι' αυτό θα στηρίξουμε την υποψηφιότητά του. Οι απαντήσει τη κυρία Σνάμπελ δεν ήταν τόσο πιστικές, αλλά δεν θα θέλαμε να αντιτεθούμε στο διορισμό της ακριβώς για λόγους ισότητας μεταξύ των δύο φύλων. Το σημαντικό είναι τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους σε αυτούς τους στόχους. Είναι στόχοι που θα πρέπει να μας ενώσουν όλους και ο στόχος της ισότητας των δύο φύλων είναι πρωταρχικός. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, από τους μη εγγεγραμμένους ε, ο κύριος Φάμπιο Μάσιμο Καστάλτο 1,5 λεπτό. Δεν τον βλέπω, είναι απόν προφανώς. Επομένως ο κύριος Στεφάν Μπεργκέρ, ε, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Και εγώ θα ήθελα εδώ καταρχήν να συγχαρώ την κυρία Σνάμπελ και τον κύριο Πανέτα και να τους ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή τύχη. Ολόκληρη η Ευρώπη ε, έχει στραμμένη την προσοχή της στο νέο προσωπικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή τη συγκυρία για να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις. Εδώ και χρόνια ζούμε σε μία φάση ε, πολύ χαλαρής νομισματικής πολιτικής ε, και αν δούμε τα αποτελέσματα αυτής της ε, πολιτικής, διαπιστώνουμε ότι η νομισματική πολιτική της ε, ΕΚΤ δημιουργεί τεράστιες ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν είναι όλες οι κοινωνίες κοινωνίες μετόχων. Πολλές κοινωνίες στις χώρες μέλη είναι κοινωνίες αποταμιευτών. Ε, ε, οι οποίοι όμως ε, είναι αναγκασμένοι να συρρυκνωθούν και ε, εδώ παρεμβαίνουν οι τράπεζες οι οποίες ασκούν όλο και περισσότερες πιέσεις σε αποταμιεύσεις. Γι' αυτό θα ήθελα να κάνω μία έκκληση προς τους υποψηφίους, τους οποίους εμείς στο ΕΛΚ στηρίζουμε, ούτε ώστε στο Διευθυντήριο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εξετάσουν αυτά τα επιχειρήματα. Ίσως θα είχε νόημα να γίνει μια σχετική συζήτηση κατά πόσο το, ο στόχο πληθωρισμού το 2% ε, παραμένει επίκαιρο και κατά πόσο θα πρέπει πάση θυσία να επιτυγχάνεται. Ελπίζω λοιπόν οι αλλαγέ στο προσωπικό της ΕΚΤ να συνοδευτούν από μια ουσιαστική συζήτηση για την πολιτική της ΕΚΤ. Και ε, εύχομαι λοιπόν σε όλους τους ενδιαφερόμενους υπό ε, το πνεύμα αυτό καλή επιτυχία. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Πέδρο Μάρκες για δύο λεπτά. Χωρίς μικρόφωνο ο μιλητής δυστυχώς. Yeah, now it's okay. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, ξεκίνησε ήδη ένας νέος πολιτικός κύκλος. Η ατζέντα για το μέλλον της Ευρώπης ε, υφίσταται και θα πρέπει να εφαρμοστεί. Ε, αναμένουμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η εκτελεστική της Επιτροπή να παίξουν το ρόλο που τους πρέπει στα πράγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε καταρχήν στα μικρά αλλά και στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Δεν μπορούμε να αναμένουμε ότι ο οικονομικός αυτός κύκλος θα παραταθεί επαόριστον. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στη νομισματική πολιτική. Είναι σημαντική η νομισματική πολιτική, αλλά όχι επαρκής. Χρειάζεται να επενδύσουμε δραστικά και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον προπολογισμό μας για τη σταθεροποίηση που θα χρειαστούμε κάποια στιγμή. Ξέρουμε ότι θα τη χρειαστούμε. Θα πρέπει να δράσουμε για το κλίμα, για την οικονομία, αλλά και για την κοινωνική συνοχή. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει να παίξει σημαντικό ρόλο και θα πρέπει να αναλύσουμε την εντολή της λαμβάνοντας υπόψη τις ε, σημερινές ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Θα πρέπει επίσης τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής να λογοδοτήσουν ε, για την ε, υπόσχεση και την ανακοίνωση της Προέδρου θα διατηρηθεί η ίδια δημοσιονομική πολιτική. Ε, η ίδια νομισματική πολιτική, συγγνώμη. Ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό ε, για να μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι η νομισματική πολιτική θα παραμείνει όπως έχει και μετά να κάνουμε και όλα τα υπόλοιπα και τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται. Ευχαριστώ πολύ. Ο... Λόγος στον κύριο Ουρτασούν τα μη σημαντικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, ε, έσωσαν την Ευρώπη ε, και αυτό επειδή τα κράτη-μέλη δεν είχαν την αποφασιστικότητα να δράσουν. Δεν είναι σωστό αυτό που λένε κάποιοι ότι ήταν παράνομα τα μέτρα αυτά. Κάποιοι κατέφυγαν, στο Δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον αυτών των μέτρων και το Δικαστήριο δικαίωσε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Βέβαια, θα πρέπει να αναλύσουμε του κινδύνου που μπορεί να δημιουργηθήκαν εξαιτία αυτών των μέτρων, για παράδειγμα τη φούσκα στην αγορά κινήτων ή κάποιου άλλου ε, τύπου παρενέργειες. Επίσης θα πρέπει να ξαναδούμε το σύνολο της νομισματικής πολιτικής έτσι ώστε να προσαρμοστεί αυτή σε πιο επίκαιρα φαινόμενα όπως για παράδειγμα ε, στην καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής πολλά τραπεζικά ιδρύματα και άλλοι φορείς ε, αγοράζουν, έχουν αγοράσει τα προηγούμενα χρόνια πολύ μεγάλο αριθμό ε, μετοχών εταιριών που ε, έχουν σχέση με την οικονομία του άνθρακα. Αυτό πρέπει να το δούμε λοιπόν. Θέλω επίσης να πω ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ε, εγκρίνουμε εκτελεστική επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας χωρίς ε, γυναίκες. Ε, η φωτογραφία της κυρίας Λαγκάρτ μόνο με άντρες είναι προσβλητική πραγματικά. Όπως είπαν και πολλοί άλλοι εδώ, έχουμε στη διάθεσή μας εξαιρετικές γυναίκες. Γυναίκες με εξαιρετικά προσόντα που θα μπορούσαν να αναλάβουν τέτοιου είδους ευθύνες. Οπότε είναι δική μας ευθύνη και μέρημνα να φροντίσουμε έτσι ώστε στο μέλλον να έχουμε ε, υποψήφιους που να μπορούν να είναι αρκετοί σε νούμερο ώστε να καλύπτουμε ε, τις θέσεις με ίσο αριθμό ανδρών και γυναικών. Οπότε για τη σωστή λειτουργία των θεσμών ελπίζουμε ότι τέτοιου είδους κατάλογοι υποψηφίων θα έρθουν στα χέρια μας στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Ερβέ για δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Έλαβα υπόψη μου τα ε, σοβαρά προσόντα και την σταδιαδρομία των δύο υποψηφίων που μας έχουν υποβληθεί ε, και ε, θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να αντιταχθούμε στο διορισμό του στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Απ' την άλλη πλευρά βέβαια έχουμε αυτό το στόχο του 2% ουτοπιστικό ή όχι. Έχουμε τα προβλήματα τα οποία ε, σχετίζονται με το νόμισμα ελικόπτερο το οποίο ενδεχομένως θα δημιουργήσει προβλήματα σε όλες τις χώρες μέλη και άλλα ερωτήματα τα οποία είναι ε, καινούργια ερωτήματα καθότι βρισκόμαστε σε μια ε, νέα κατάσταση όσον αφορά τα νομισματικά. Σε όλη τη χώρα οι νεοκαπιταλιστικές θεωρίες έχουν αποτύχει σε όλο τον κόσμο ε, λειτουργούν καταστάσεις οι οποίες φέρνουν ε, πρώτους στις εκλογές τον κύριο Τραμπ ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή τον Μπόρι Τζόνσον στην Μεγάλη Βρετανία. Νομίζω ότι βρισκόμαστε πλέον στα πρόθυρα ενός νέου νομισματικού κόσμου. Γι' αυτό λοιπόν όταν εγώ αναφέρομαι σε διαφοροποίηση θα ήθελα να ρωτήσω το εξή το σώμα. Δεν θα έπρεπε στο Συμβούλιο της ΕΚΤ να υπάρχουν εκπρόσωποι εκπρόσωποι της ψηφιακής οικονομίας. Δεν θα πρέπει ε, να ε, υπάρχουν εμπειρογνώμονες, ε, πολιτικοί επιστήμονες που να μας θυμίζουν ότι το εργαλείο της της κυριαρχίας ε, ε, ισχύει ακόμα και οπωσδήποτε δεν είναι δυνατόν να ακολουθήσουμε βιώσιμες πολιτικές σε ένα κόσμο που δεν είναι βιώσιμος. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να το λάβει αυτό υπόψη του και το Συμβούλιο έτσι ώστε να μας υποβάλει διαφοροποιημένες λίστες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μακάρθη για ένα λεπτό. ECB η ΕΚΤ ε, θα αναθεωρήσει την ε, πολιτική της. Ε, συμφωνώ με τα όσα είπε ο, ο πρόεδρος ε, εν σχέση με, τα, με την παροχή ε, κινήτρων. Ωστόσο, η ΕΚΤ ήταν υπεύθυνη για την πολιτική λιτότητα στα προηγούμενα χρόνια. Φαίνεται τώρα να αλλάζει η πολιτική η αναθεώρηση ε, της ΕΚΤ θα πρέπει να γίνει στη βάση μια σοβαρής ανάλυση των επιπτώσεων της πολιτικής της ΕΚΤ σε όλη την Ευρωζώνη ε, ε, και να περιλάβει και τα φαινόμενα της φούσκας στις αγορές. Οι πολιτικές της ε, ΕΚΤ ε, συνέβαλαν στην αύξηση της ευημερία ενός πολύ μικρού ποσοστού πολιτών, αλλά όχι του συνόλου των Ευρωπαίων ε, πολιτών. Θα πρέπει να επανεξαταστούν οι πολιτικές πληρονομών στα νοικοκυριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων. Ο κύριος Φάβιο Μάσιμο Καστάλντο ε, ήρθε πλέον. Θα του δώσω το λόγο για 1,5 λεπτό, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να προσθέσω κάποιε σκέψει όσον αφορά το διορισμό του Φάβιο Πανέτα ω ε, μέλο ε, τη Εκτελεστική Επιτροπή Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Οπωσδήποτε πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίο είναι ιδιαίτερα γνώστη του τραπεζικού τομέα. Πρόκειται για επιστήμονα ο οποίο γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα τεκτενόμενα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχοντας συμμετάσχει μαζί με τον διοικητή της ε, Τράπεζας ε, και, μαζί με τον πρόεδρο ε, των προηγούμενων Ευρωπαϊκή Κεντρικής Τράπεζας σε πολλές εργασίες της ιδείας. Έχει αναλύσει αίτια της κρίσης, σενάρια σχετικά με την επίλυση της κρίσης, σενάρια για, την, για το μέλλον και τα συμφέροντα της Ευρώπης. Φτάνει στην Φραγκφούρτη μια πολύ ευαίσθητη στιγμή. Ε, που μια στιγμή που η έκτο θα πρέπει να ασχοληθεί με θέματα ευρύτατα ε, από τα οικονομικά, νομισματικά αλλά και τα κλιματικά. Ε, οπωσδήποτε θα αρθεί στο ύψος των περιστάσεων βάσει αρχών που διείπαν πάντοτε την εξαιρετική του καριέρα και στα διαδρομή. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να δώσω τον ε, λόγο στον επόμενο ομιλητή, ο κύριος Πολ Τάγκ, δύο λεπτά, από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε, κύριε Επιτρόπε. Μερικές φορές ε, μια φωτογραφία είναι όσο καλή και χιλιάς λέξεις. Η φωτογραφία της κυρίας Λαγκάρτ ε, μαζί με τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ήταν πραγματικά πολύ ευγλωτή. κάτω από ένα κλασικό πολυέλαιο και δίπλα σε πίνακες ε, μπαρόκ το χαμόγελο της ε, κυρίας Λαγκάρτ <laughs> φώτιζε όλους τους υπόλοιπους άντρες που είχε γύρω της. Πραγματικά θα πίστευε κανένας ότι ε, η φωτογραφία ερχόταν από την εποχή του άνθρακα, του κάρβουνου, συγγνώμη, του Ζαν Μονέ. αυτή η φωτογραφία θα πρέπει να μας ξυπνήσει. Δείχνει ότι ο αγώνας για την ισότητα των δύο φύλων παραμένει επίκαιρος. Και εγώ προσωπικά, αλλά και οι σοσιαλιστές και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλούν το Συμβούλιο να υποβάλει πάντοτε έναν άντρα και μία γυναίκα για την ίδια θέση. Ε, το Eurogroup <laughs> άλλωστε έχει μόνο μία γυναίκα μεταξύ των 19 μελών του. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι συμβαίνει αυτό. Αν το, κοινοβου... το Συμβούλιο δεν επικαιροποιήσει την πολιτική διορισμό του, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Πώς μπορούν να λαμβάνονται δίκαιες αποφάσεις όταν ο μισός πληθυσμός της γης εξαιρεί, της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιρείται από τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Πώς μπορούμε να, είμαστε, να ζούμε στη σύγχρονη εποχή με διαδικασίες που ανήκουν στον προηγούμενο αιώνα. Ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα κάνει τα λόγια πράξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζωμαν Χάιντερ. Δύο λεπτά. Κύριε Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή η ΕΚΤ ε, με την πρόεδρο Λαγκάρτ ε, αποδεικνύει πόσα, πόσο λέθριες ήταν οι επιπτώσεις της ε, πολιτικής χαμηλών ε, επιτοκίων στο παρελθόν με τη διατήρηση και με την αύξηση τεχνητών τιμών στην αγορά κινητήτων και τη δημιουργία από φούσκες στην αγορά. Ε, με τον τρόπο αυτό ε, ε, τελικά ζημιώνονται οι Ευρωπαίοι πολίτες και όλα αυτά δεν σχετίζονται καθόλου με σταθερότητα τιμών. αυτοί οι οποίοι ευνοούνται είναι μόνο οι κεροσκόποι και οι απατεώνες. Εδώ αυτό το οποίο χρειάζεται είναι πειθαρχία και ε, βλέπουμε ότι εδώ είναι κατάλληλη η κυρία Σνάμπελ. Οι προκάτοχοί τη, τρεις προκάτοχοι τη κυρία Σνάμπελ παρετήθηκαν ακριβώ λόγω των ολέθρων επιπτώσεων των χαμηλών επιτοκίων. Ε, με την εξαγγελία της ότι Ε, η ΕΚΤ ε, θέλει να καταπολεμήσει τις αρνητικές ε, περιβαλλοντικές επιπτώσεις μετατρέπει την ΕΚΤ σε λόμπι καιροσκόπων και απαταιώνων. Η κυρία Σνάμπελ πιστεύω ότι και αυτή θα υποστηρίξει αυτή την ε, νομισματική πολιτική η οποία στρέφεται κατά των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Δύο λεπτά κυρία Μπέκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εμείς οι γυναίκες ε, ε, αποτελούμε το ίμιση του πληθυσμού. Ε, γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε και το ίμιση από το γλυκό. Ε, και αυτό είναι διάφορο κατά πόσο πρόκειται για την ε, ΕΚΤ ή οποιοδήποτε άλλον ε, οργανισμό. Θα πρέπει να εκπροσωπούμε εκπροσωπούμεθα ισόρροπα. Όλοι γνωρίζουν αυτή τη φωτογραφία όπου βλέπουμε μοναχική την κυρία Λαγκάρτ μεταξύ αντρών. Ε, η εικόνα αυτή δεν ανταποκρίνεται στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. Χρειαζόμαστε ευφυεί γυναίκες όπως και νοήμονες άνδρες. Ε, θέλουμε και εμείς να συμβάλλουμε στην διαμόρφωση αυτής της πολιτικής. Ε, έχουμε και εμείς το δικό μας λόγο όσον αφαιρά τι βιώσιμε επενδύσει για την Ευρώπη όσον αφορά μια σωστή νομισματική πολιτική προκειμένου να κάμψει η οικονομία, όσον αφορά τους κοινούς φορολογικούς ε, κανόνες και την ε, ε, πρόθεση μιας πράσινης οικονομίας. Αξιότιμα κύριε Επίτροπε, βλέπετε ότι το εφιστάμενο σύστημα διορισμού ε, είναι παροχημένο. Ε, θα πρέπει να το αναθεωρήσετε και να το διαμορφώσετε εκ νέου. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπέκ. Αξιότιμοι συνάδελφοι, ε, στα μέσα Νοεμβρίου η κυρία Σνάμπελ στο Twitter είπε στους πράσινους ε, οικολόγους να μην ε, κάνουν σαλμένες κριτικές όσον αφορά την ΕΚΤ γιατί με τον τρόπο αυτό ε, απειλείται το ευρώ, η ευρωζώνη. η κυρία Σνάμπελ αναφέρθηκε υποτιμητικά σε οικονομικά αναλφάβητος. Όμως όλοι γνωρίζουμε ότι η ΕΚΤ έχει αποτύχει. Η οικονομική της πολιτική οδήγησε σε μια αύξηση φόρων και μια ζημίωση του περιβάλλοντος. Ε, η ίδια η ΕΚΤ ομολόγησε ότι οι χρηματικές ε, ροές ε, εισραίουν σε υπερχρεωμένες επιχειρήσεις σε χώρες που διανύουν κρίσεις. Και η πολιτική αυτή ε, στήχησε 650 εκατομμύρια διαφυγόντων ε, εσόδων για τους ε, Γερμανούς φορολογουμένους. Εμείς ε, θέλουμε την άμυλα των ιδεών, γιατί μόνο αυτή μπορεί να μας οδηγήσει στην αλήθεια και δεν συμφωνούμε με την οτροπία της κυρίας Σνάμπερ. κύριος Μαξιμίλιαν Κράχ, για ένα μισή λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, ε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα τα όσα υπόθηκαν, ιδιαίτερα τα όσα είπε ο κύριος Μπέργκερ, ο οποίος μας είπε ότι υπάρχουν δύο τύποι κοινωνιών, οι κοινωνίες των μετόχων και οι κοινωνίες αυτών που αποταμιεύουν. Και, και οι κανόνες, ο κ. Πανέτα είπε ότι οι κανόνες του ΕΚΤ δεν στοχεύουν στη διάσωση ε, της ε, Ιταλίας. Ενδεχομένως ε, έχει δίκιο. Ωστόσο βλέπουμε ότι εδώ υπάρχουν διαφορετικές οικονομικές προσεγγίσεις. Και το πώς μπορούμε να επενούμε αυτούς τους διορισμούς. Αυτό είναι μυστικό των ε, Γερμανών ε, συντηρητικών ε, κομμάτων και του ΕΛΚ. Ο κύριος Πανέτα μπορεί να έχει εξαίρετη μόρφωση και γιατί η Γερμανία προτείνει την κυρία Σνάμπελ η οποία ζημιώνει τους ε, Γερμανούς ε, πολίτες που επιθυμούν να αποταμιεύσουν παραμένει μυστικό της γερμανικής κυβέρνησης. Κυρία Ρέγνερ, εδώ δεν πρόκειται για κανένα γλυκό, πρόκειται για χρήματα, πρόκειται για ποιότητα και εξασφάλιση υψηλών ε, προσόντων. θα πρέπει να κάνουμε κάποια σκέψη για την οικονομία, όχι να μιλάμε για γλυκά. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσει τώρα ε, η διαδικασία Catch the Eye. Δεν υπάρχει όμως κάποιος εγγεγραμμένος, άρα ο κύριος Τζεντιλόνι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι πρέπει να συγχαρούμε τον κύριο Κερέ που ήταν μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής ε, τα τελευταία 8 χρόνια, συγχαρητήρια. Επίσης την Σαβίν Λάουτενσλέγκερ για τη συνεισφορά της ως ε, μέλος του, της Εκτελεστικής Επιτροπής επίσης και για, τον, ε, για το συνολικό της ε, έργο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όπως γνωρίζετε η Κομισιόν δεν εμπλέκεται στην διαδικασία διορισμού, όμως Εκτιμούμε ιδιαίτερα τα, τα δύο νέα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, είναι πολύ ικανά και ταυτόχρονα συμμεριζόμαστε και την προσήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επαναλήφθηκε από πολλά στόματα σήμερα προκειμένου να αντιπροσωπευτεί καλύτερα και το άλλο φύλλο ε, ε, στον, σε όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούσαμε επίσης με πολύ προσοχή τα σχόλιά σας για την ε, μακροοικονομική πολιτική της Ευρωζώνης. Και να προσθέσω το εξής μόνο. Πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια το βάρος της αναθέρμανσης της ευρωπαϊκής οικονομίας έπεσε υπερβολικά πολύ στην νομισματική πολιτική στην ζώνη του ευρώ. Χρειάζεται μια, ένα μείγμα πολιτικών πιο αποτελεσματικό και πιο ισορροπημένο και αυτό θα βασιστεί στην φορολογική πολιτική και σε διαστοτικές μεταρρυθμίσεις. Η φορολογική πολιτική ε, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη βιωσιμότητα του χρέους, ιδιαίτερα των υπερχρωμένων κρατών μελών. Αυτή η φορολογική πολιτική μπορεί να αυξήσει την εσωτερική ζήτηση ε, και να αυξήσει τις ε, προσδοκίες για τον πληθωρισμό. Ε, το τόνισε αυτό η κυρία Λαγκάρ στο κοινοβούλιο εδώ πρόσφατα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Ευχαριστώ πολύ κυρίε και κύριοι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να κλείσω αυτή την κοινή συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης. Είναι μια προφορική ερώτηση που αφορά τη δίκαιη φορολόγηση σε μια ψηφιοποιημένη και παγκοσμιοποιημένη οικονομία ε, BPS e 2.0. Για να λάβετε τον ε, λόγο, ε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνήθεια διαδικασία. Επίσης υπάρχει διαδικασία και για την μπλε κάρτα και για την διαδικασία Catch the Eye. Στην είσοδο θα βρείτε οδηγίες. Δίνω το λόγο στην κυρία Τινάλη που για να μας παρουσιάσει την ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, 250 δις δολάρια αυτό είναι το ποσό ε, των ε, διαφυγέντων εσόδων ε, από την φοροδιαφυγή. Ε, μία μελέτη του Πανεπιστημίου της ε, Κοπενχάγης ε, κατέληξε ότι 40% των κερδών των πολλών εταιριών έχει προωθηθεί προς παραδείσους, φορολογικούς παραδείσους, ενώ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά έτσι ώστε να ενισχυθούν οι δημόσιες υπηρεσίες και οι δημόσιες σε παροχές, την εκπαίδευση, την υγεία κλπ. Για να μην αναφέρουμε επενδύσει, οι οποίε θα μπορούσαν να έχουν ε, επενδυτικό ε, ενδιαφέρον και απόδοση. Όλοι πρέπει να συμβάλλουν ε, αλλά ενώ οι πολίτες, οι καταναλωτές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πληρώνουν ό,τι τους αναλογεί, ε, με φορολογικούς συντελεστές που μπορεί να φτάνουν ή και να ξεπερνούν ακόμα το 40% πολλές πολυεθνικές εταιρείες δεν ε, συμβάλλουν με τον ίδιο τρόπο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί προβλήματα κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά προκαλεί ε, και στρέβλωση του ανταγωνισμού. Πολλά συζητούμε και επιμακρών όσον αφορά ε, την δημιουργία ενός ε, ίσου ε, τρόπου όσον αφορά τον ανταγωνισμό και με ίσων προϋποθέσεων. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν εάν να υπάρξει κάτι τέτοιο, εάν δεν υπάρχει ένα ίδιο πλαίσιο ε, για όλους. 135 χώρες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν ε, αυτό το πρόβλημα και τώρα ε, έχουμε όσον αφορά την μεταρρύθμιση και έκθεση και ερώτημα με έτοιμα προφορικής απάντησης προς την Επιτροπή. Θα πρέπει να συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια συμφωνημένη, συνεκτική και ε, φιλόδοξη θέση. Ε, ερωτώ λοιπόν προ την Κομισιόν Πώ προτίθεται η Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμμετέχει με κοινή θέση στι διεθνεί συζητήσει των ΩΣΑ σχετικά με τι φορολογικέ προκλήσει που εγείρει η ψηφιοποίηση τη οικονομία. Επίση, πώ προτίθεται η Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι συνεχιζόμενε συζητήσει στο διεθνέ επίπεδο σχετικά με τον πρώτο και το δεύτερο πυλώνα θα είναι συνεκτικέ και συνεπεί με τι προτάσει Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τρίτη ερώτηση, με ποιο τρόπο προετοιμάζει η Κομισιόν την εφαρμογή αυτή τη πιθανή διεθνή συμφωνία και τι θα γίνει σε περίπτωση που δεν εξευρεθεί λύση σε διεθνέ επίπεδο, τι προτίθεται να πράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πότε, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δράσει συντονισμένα για να προστατέψει την ενιαία αγορά από περαιτέρω κατακαιρματισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει και μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο ε, σε όλα ε, αυτά τα θέματα, με την προϋπόθεση όμως ότι θα έχει συνεκτική και ενωτική θέση. Το Κοινοβούλιο επικεντρώνεται σε δύο στοιχεία. Θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να μεταρρυθμιστεί η ιδέα της φορολόγησης σε σύγκριση, σε σχέση μάλλον με την εδαφική παρουσία, έτσι ώστε να αποσχιστεί από την φυσική παρουσία. Δεύτερον, θα πρέπει οπωσδήποτε να καθοριστεί ε, ένα ε, συγκεκριμένο ελάχιστο ε, εισοδηματικό επίπεδο έτσι ώστε να μην υπάρχει πλέον στρέβλωση του ανταγωνισμού. Επίσης υπάρχουν χώρες στις οποίες ο ενιαίο, το ενιαίο ποσοστό φορολόγησης των επιχειρήσεων είναι 0% ή σχεδόν 0%. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να υπάρξει ένα συμφωνημένο ελάχιστο όριο. Ε, θα πρέπει τα χρήματα από τους φόρους να χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία περαιτέρω ε, αξίας. Ε, θα πρέπει σε αυτήν την νέα ψηφοποιημένη, παγκοσμιοποιημένη οικονομία να μην αφήσουμε περιθώρια στον, στην εφοροϋποφυγή και στην εφοροδιαφυγή. οι χώρες ε, οι οποίες ε, ε, αποφασίζουν να χρηματοδοτήσουν τις κοινέ τους δημόσιες πολιτικές μέσα από την φορολόγηση των επιχειρήσεων θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Δεν είναι σωστό, δεν είναι δίκαιο να μην υπάρχει δικαιοσύνη φορολογική. Την ζητούν οι πολίτες μας και πρέπει να τους τη δώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος ε, της ε, Επιτροπής θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο κύριο Τζεντιλόνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ πολύ κυρία Τινάλη που τοποθετήσατε ε, στην ημερήσια διάταξη αυτό το θέμα της ε, διεθνούς φορολόγησης επιχειρηματικών κερδών είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την Επιτροπή ΕΚΟΝ και την Επιτροπή ΤΑΞ και προφανώς για όλο το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ και για το παλιότερο έργο σας για αυτό το θέμα. Η Κομισιόν ε, αναζητά μια ευρωπαϊκή λύση. Θα πρέπει για παράδειγμα να συνεργαστούμε στο μέλλον στον εξυγχρονισμό των φορολογικών κανόνων για τα επιχειρηματικά κέρδη. Για παράδειγμα, οι φορολογικέ δραστηριότητε θα πρέπει να φορολογούνται ακόμη και χωρί φυσική παρουσία. Αυτό αφορά τον πυλώνα 1, τη μετατόπιση των φορολογικών δικαιωμάτων. Επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ε, και τους, ε, τις νέες μορφές ε, άδικου φορολογικού ανταγωνισμού που είναι ο πυλώνας 2. Οι λύσεις θα πρέπει να είναι παγκόσμιες, ε, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνουν τα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα, ιδιαίτερως αυτών των επιχειρήσεων που λειτουργούν χωρίς φυσική παρουσία σε συγκεκριμένες φορολογικές δικαιοδοσίες. Επίσης, θα πρέπει να ε, φρενάρουμε και να μειώσουμε τον, τον υπερβολικό φορολογικό ανταγωνισμό εργαζόμενοι σε διεθνές επίπεδο για μια παγκόσμια λύση, ταυτόχρονα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή έκβαση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Θέλω να σας καθησυχάσω και να δηλώσω ότι οι ιδιαιτερότητες της εσωτερικής αγοράς θα τύχουν σεβασμού σε οποιαδήποτε λύση προκύψει από διεθνείς διαπραγματεύσεις. Πάντα εργαζόμαστε προς όφελος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των ευρωπαίων φορολογουμένων. Γι' αυτό το λόγο στόχος μας είναι να πετύχουμε αυτούς τους στόχους χωρίς περαιτέρω επιπλοκές στους κανόνες που διέπουν τις επιχειρήσεις. Οι νέοι κανόνες θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι απλοί και ε, θα πρέπει να γίνει ε, μια αναδιανομή υπέρ των συμφερόντων των πολιτών μας. Θα πρέπει να δούμε αναλυτικά τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί για τους πρώτους δύο πυλώνες έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να πάρουν τις αποφάσεις τους ενημερωμένα. Τα πρώτα πορίσματα είναι θετικά. Ε, αναφέρουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βγει κερδισμένη από τον πυλώνα 1 και όλα τα κράτη-μέλη θα ε, βγουν ευνοημένα από τον πυλώνα 2. Η Κομισιόν έχει ζητήσει πλέον ε, τα, από τα κράτη-μέλη να υποβάλουν τα εθνικά του στοιχεία έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε πιο λεπτομερή την οικονομική μας ανάλυση. Ω συμπέρασμα, αν καταλήξουμε σε παγκόσμια συμφωνία για, και για του δύο πυλώνε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποφασίσει πώ θα εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία ε, διεθνώς ή αν η συμφωνία είναι μερική μέχρι το 2020, είναι απόλυτα σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τότε η Κομισιόν θα αναλάβει δράση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Και τώρα, εξ του ΕΛΚ, θα δώσω το λόγο στον κύριο Μάρκους Φέρμπερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά κύριε Επίτροπε για αυτή την ξεκάθαρη δέσμευσή σας που μόλις ε, διατυπώσατε. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό πολλά πράγματα τα οποία ε, ζητήσαμε από κοινού, διαπιστώσαμε από κοινού στην προηγούμενη θητεία θα πρέπει να λυθούν. Και η καλύτερη δυνατή λύση βεβαίως ε, ε, είναι να γίνει διασυνοριακά γιατί τα φορολογικά προβλήματα είναι διεθνή και θα πρέπει να τα προσεγγίσουμε σε αυτή τη διεθνή τους διάσταση. Ούτε ώστε οι χώρε μέλη να γίνουν ενεργά, αλλά και άλλα επίπεδα δικαιοδοσία, όπως είναι η ΕΠΑ, για παράδειγμα, που ιδιαίτερα στον τομέα της ψηφιοποίηση ε, δραματίζουν σημαντικό ρόλο. Θα πρέπει να απομακρυνθούμε από την ιδέα μιας ε, φυσικής ε, παρουσίας, ε, μιας επιχείρησης υπαρκτών μηχανημάτων και υπαρκτού φυσικού, εργατικού, φυσικής παρουσίας του εργατικού δυναμικού. Όλα αυτά δεν παίζουν πλέον κανένα ρόλο. Γι' αυτό θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά τα θέματα, πώς έχει ψηφιοποιηθεί δηλαδή η οικονομία. Αλλά θα πρέπει να καθαρίσω τα μετά του οίκου μας πρώτα. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ένας ε, ανταγωνισμός ε, εις βάρος των εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσεγγίσουμε ξεκάθαρα τα προβλήματα και καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι μόνο την Επίτροπο Ανταγωνισμού, αλλά και ε, καλό και εσάς ως νέο επίτροπο να δείτε αυτά τα φορολογικά θέματα γιατί θα πρέπει να ξηρανθούν οι δικές μας φορολογικές οάσεις πρωτίστως. Σας ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος των σοσιαλιστών θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Φερνάντες. Ευχαριστώ πολύ κύριε, κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Πριν από λίγη ώρα συζητούσαμε για την νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά δεν συζηλέγαμε ποια θα είναι αυτή ε, η πολιτική σε σχέση με άλλες κεντρικές τράπεζες. Λέγαμε τι πρέπει να κάνει ε, σχετικά με την είσοδο ή έξοδο ροής ε, κεφαλαίων και ποιο είναι το αποθεματικό. Δεν το συζητούσαμε όμως γιατί καταφέραμε να ασκήσουμε εν τέλει ευρωπαϊκή κυριαρχία όσον αφορά την νομισματική πολιτική. Κάτι που τα κράτη-έθνη δεν είχαν τη δεκαετία του 90 ε, όταν ε, ε, απέτυχε το νομισματικό πρόγραμμα της Ευρώπης και όταν δεν ήταν οι χώρες ικανές να ασκήσουν την νομισματική τους πολιτική. Τώρα έχουμε φορολογική πολιτική γιατί τώρα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο γιατί οι μεγάλες εταιρείε, οι ψηφιακέ πολλές εταιρείες ε, ε, ε, μετακινούνται από τις διάφορες νομικές δικαιοδοσίες και προσπαθούν να κινηθούν μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών έτσι ώστε να μην πληρώσουν φόρους και οι εθνικές αρχές ενώ τυπικά έχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τη δική τους φορολογική πολιτική δεν καταφέρνουν να το κάνουν και θα πρέπει λοιπόν την επιτυχία που είχαμε με την νομοθετική πολιτική πολιτική, να την εφαρμόσουμε και στην φορολογική πολιτική. Δεν θέλουμε κράτη-έθνη, θέλουμε ελάχιστες ε, ε, ε, φορολογητές βάσεις. Χρειαζόμαστε επίσης ένα κοινό πλαίσιο φορολόγησης όσον αφορά την κίνηση των κεφαλαίων. Χρειαζόμαστε ελάχιστα πρότυπα ελέγχων έτσι ώστε να υπάρχει η διασφάλιση ότι κάποιος ηγείται ε, των θεμάτων αυτών κάποιος ο οποίος ε, ε, θέλει να προωθήσει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να ενεργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να αναλάβει τα ενία της φορολογικής πολιτικής. Ευχαριστώ πολύ για την ομάδα Renew, ο κύριος Γκαρικάνο. Ευχαριστώ. Κύριε Τζεντιλόνι, σας πω μερικά νούμερα. Δεν θα τα πιστέψετε. Πέρσι η Apple στην Ισπανία πλήρωσε 4 εκατομμύρια ευρώ φόρο με 394 εκατομμύρια πράξεις. Το Facebook 864.000 864, ευρώ και το Netflix πλήρωσε 3.146 ευρώ φόρο. 3.000 φόρο. Με... με σε ένα κτίριο το οποίο, στο οποίο θα χωρούσαν 24 κατοικίε ε, έχει έδρα το Netflix στην Ισπανία. Μόνο με τα ενίκια θα πληρώνουν παραπάνω. Αυτά είναι παραδείγματα για το πώ οι μεγάλε πολυεθνικές εταιρείε αποφεύγουν να πληρώνουν φόρου. Πώ θα ζητήσουμε από του πολίτε μα και από τι μικρέ επιχειρήσει να πληρώνουν το δικό του φόρο αν επιτρέπουμε αυτοί που κερδίζουν τόσο πολλά να μην πληρώνουν. Πώς θα χρηματοδοτήσουμε το κράτος ευμερίας μας αν αυτοί που, που κερδίζουν τα πιο πολλά δεν συνεισφέρουν αναλογικά. Πώς θα υπερασπιστούμε την ελεύθερη αγορά αν οι κανόνες δεν είναι ίδιοι για όλους. είναι μία από τι μεγαλύτερε προκλήσει που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Οι πολίτε μα μας κοιτούν στα μάτια και ελπίζουν ότι θα βρούμε μία δίκαιη λύση. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε ότι η μαγκοσμιοποίηση και η ψηφιοποίηση άλλαξαν τον κόσμο. Όμω, όπως έλεγε ο κ. Φέρμπερ, συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις του 21ου αιώνα με μέτρα του 19ου. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Η φορολογία θα πρέπει να προσαρμοστεί στην καινούργια εποχή. Το ψήφισμα αναζητεί κανόνες έτσι ώστε η, ε, η ίσπραξη των φορών να συμβαδίζει με τη δημιουργία κερδών. Αυτή η πρωτοβουλία θα πρέπει να υιοθετηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Μία χώρα από μόνη τη δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να αντιμετωπίσει την φοροδιαφύγη και τη φοροαποφυγή μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων. Γι' αυτό λόγο θα πρέπει να συνεργαστούμε και η συνεργασία να ξεπεράσει τα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπω είπε η κυρία Τινάλη, το θέμα δεν είναι μόνο η φορολόγηση των ψηφιακών επιχειρήσεων, αλλά και πολλών άλλων πολυεθνικών. Οπότε, στόχος νούμερο ένα, παγκόσμια λύση στον ΩΣΑ. Είναι το κατάλληλο φόρουμ. Αλλά, όπως είπατε κι εσείς, αν ο ΩΣΑ δεν θα καταφέρει μέχρι το τέλος 2020 να καταλήξει σε συμφωνία, θα πρέπει να πάρουμε εμείς εδώ τα μέτρα μας. Και εμείς θα τα στηρίξουμε. Αν στον ΩΣΑ καταλήξει σε αποτυχία διαπραγμάτευση το ψήφισμα επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει μια ενιαία φωνή στι διαπραγματεύσει αυτέ. και είμαστε υπέρ τη φορολογική δικαιοσύνη. Το ψήφισμα καθιστά σαφέ ότι δεν θα δεχτούμε ούτε μικρέ επιχειρήσει ούτε οι αυτοπασχολούμενοι να πληρώνουν περισσότερου φόρου από ότι οι πολυεθνικέ επιχειρήσει. Θέλουμε μια ανοιχτή ελεύθερη αγορά, αλλά με κοινού κανόνε για όλου. Θα υπερασπιστούμε το κράτο ευημερία μα και τα έσοδά μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, εκ μέρους των Πρασίνων, ο κύριος Γκίγκολτ θα πάρει το λόγο για 3,5 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Εδώ και 20 χρόνια από τότε που ήμουν στο Πανεπιστήμιο μάχομαι υπέρ μιας φορολογικής δικαιοσύνης για ένα ελάχιστο φορολογικό συντελεστή και αύξηση της, της διαφάνειας ούτως ώστε αυτοί που χάνουν από την παγκοσμιοποίηση να μην ε, πληρώνουν περισσότερους ε, φόρους, αλλά να έχουμε ένα πιο δίκαιο φορολογικό πλαίσιο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θλίβει όταν ε, διαπιστώνω ότι παρά τις ε, προσπάθειες μιας ε, διεθνούς φορολογικής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο πέρσι και πρόπερσι για πρώτη φορά ο ουσιαστικός φορολογικός συντελεστής των επιχειρήσεων έπεσε κάτω από το 20% και ξέρουμε ότι αυτοί οι πολύ χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές δεν προέρχονται από το γεγονό ότι οι μικρές επιχειρήσεις δεν πληρώνουν ε, φόρους αλλά είναι οι μεγάλοι όμιλοι αυτοί οι πολυεθνικές επιχειρήσεις οι οποίες ε, φοροδιαφεύγουν και δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε τις καταστροφικές επιπτώσεις αυτής της φορολογικής ανισότητας αυτό ζημιώνει την ιδέα της ε, οικονομίας της ε, αγοράς ε, που έχει το νόημα ότι όλοι εντός της αγοράς δρούν κάτω από ίδιες προϋποθέσεις. Επίσης, ζημιώνει την ιδέα της εσωτερικής αγοράς. Για μια εσωτερική αγορά γιατί πρόκειται για μια ιστορική αγορά όπου ορισμένες επιχειρήσεις δεν φορολογούνται. Και με τον τρόπο αυτό το ζήτημα αυτό άπτεται της νομιμοποίησης, δημοκρατικής νομιμοποίησης της ε, δημοκρατικής ε, συνεργασίας μεταξύ των χωρών μελών. Εδώ και πολλές δεκαετίες συζητούμε για, για το θέμα αυτό, αλλά δεν καταφέρνουμε να το λύσουμε. Και αυτό, όπως σας είπα, συνδέεται με την νομιμότητα ε, του, ε, της, ε, του Συμβουλίου, της Επιτροπής αλλά και του ίδιου του Κοινοβουλίου έστω και αν το Κοινοβούλιο διαδρανώνει τη θέλησή του εδώ και χρόνια να λύσει αυτό το πρόβλημα. Ε, όσον αφορά και το τραπεζικό ε, τραπεζική χεμήθεια οι επιχειρήσεις ε, έχουν ε, εκατομμύρια ε, σκιώδεις, εικονικές θυγατρικές οι οποίες δεν φορολογούνται ποτέ. Αυτό που αποφασίσαμε στην Επιτροπή Juncker, την οδηγία κατά της φοροαποφυγής 1 και 2, το σύστημα BEPS, έχει τόσα ελλείμματα που δεν αξίζει καν το χαρτί πάνω στο οποίο είναι τυπωμένο. Οι αγορές ακινήτων είναι έτσι διαρθρωμένες ούτως ώστε ε, τα κέρδη να μεταφέρονται σε τρίτες χώρες. Γι' αυτό είναι κατεπήγον να έχουμε ελάχιστους κοινού φορολογικούς συντελεστές. Είναι θλιβερό το γεγονός ότι, ορισμέ, ότι οι χριστιανοδημοκράτες και κάποιοι φιλελεύθεροι ε, έχουν ε, πρόβλημα να προσχωρήσουν σε αυτή την ιδέα της θέσπισης ελάχιστων φορολογικών συντελεστών νομίζω ότι έχει έρθει ε, το, επίσης το πλήρωμα του χρόνου το Συμβούλιο να προχωρήσει σε μια φορολογική διαφάνεια. Ευχαριστώ πολύ για την ε, ομάδα ID. Δίνω το λόγο στον κύριο Μπέκ. Κυρία Πρόεδρε, ε, καταγγελίες για φορολογικό dumping και χαμηλές φορολογικές εισπράξεις δρούν καταλητικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να έχει μία φορολογική πολιτική με μία ενιαία φορολογική αρχή, ούτως ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη φορολογική ολοκλήρωση μέσω θέσπιση ενός ψηφιακού φόρου. Οι προθέσεις είναι ξεκάθαρες καταρχήν θα δημιουργήσουν νέες υπερεθνικές αρμοδιότητες. Τα εθνικά, οι εθνικές υπηρεσίες θα αποδυναμωθούν. Όλο και λιγότερες αποφάσεις θα λαμβάνονται κατά συνέπεια δημοκρατικά. Ε, παντοδύναμε θα είναι οι λεγόμενοι ανεξάρτητοι οργανισμοί, η ΕΚΤ, τα δικαστήρια. Άρα λοιπόν οι ανεύθυνοι οργανισμοί, ε, ε, ε, μετατρέποντας την οικονομία σε μεταναστευτική πολιτική ε, εις βάρος του, των πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικαλείται το άρθρο 113 για ομοφωνία και ταυτόχρονα προσπαθεί να το παρακάμψει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, επιβάλλει τους υψηλότερους φόρους της επιχειρήσης. Ωστόσο, ε, τα ε, κέρδη πληρώνονται υπέρ των παράνομων μεταναστών. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, συνετιστείτε. Οι πολίτες θέλουν περισσότερη δημοκρατία και κράτος δικαίου. Όχι περαιτέρω πληρωμές ε, υπέρ σεναρίων, φανταστικών σεναρίων ε, διάσωσης. Για την ECR δίνω το λόγο στον κύριο Ζόντσα για μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι. Κύριε Επιτροπέ. Ας ε, δεχτούμε ότι όλοι είμαστε υπέρ της ε, καταπολέμησης των επιθετικών φορολογικών πολιτικών ε, και σε αυτό είμαστε όλοι σύμμαχοι. Θα πρέπει όμως να βρούμε και μια να αναζητήσουμε και μια συμφωνία, μια συνένεση σε παγκόσμιο επίπεδο. Νομίζω ότι τέτοιου είδου ε, επιθετικέ πολιτικέ ε, έχουν επηρεάσει πολύ την οικονομία και θα, συνεχίσουν να την επηρεάζουν. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε μια απλή λύση που θα βασίζεται σε αυστηρέ αναλύσει. Δυστυχώ όμω το ψήφισμα δεν είναι λογικά συνεπέ. Δηλαδή, από τη μια μεριά χαιρόμαστε για την δημιουργία του δεύτερου πυλώνα αυτού που αποκαλείται δεύτερος πυλώνας. Φορολόγηση της δραστηριότητα εκεί στο που λαμβάνει χώρα. Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Στην πραγματικότητα η κατάσταση είναι διαφορετική γιατί αυτός ο κανόνας θα φορολογήσει εταιρείε που ε, μία θηγατρική τους έχει ε, πουλήσει αγαθά υπηρεσίες ε, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη πού έλαβε χώρα η δραστηριότητα. Πρέπει να τα αναλύσουμε καλύτερα και θα πρέπει να προβλέψουμε και εξαιρέσεις έτσι ώστε το κείμενο αυτό πραγματικά να δώσει θετικό αποτέλεσμα γιατί αλλιώς μπορεί να έχει παρενέργειες σε πολλές χώρες και να ευνοήσει μόνο μερικές. Θα πρέπει να αλλάξουν υπόψη τα συμφέροντα όλων. Ευχαριστώ. Ο λόγος τώρα στον, στην ΚΟΕ και στον κύριο Κουσμάου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό το κείμενο είναι μια προσπάθεια να ε, καταπολεμηθεί η φοροαποφυγή ε, των μεγάλων επιχειρήσεων, ε, η οποία δημιουργεί τεράστιες απώλειες φορολογικών εισόδων, εσόδων. Αυτά τα φορολογικά έσοδα οδηγούν σε αύξηση του φόρου για τον υπόλοιπο, την υπόλοιπη φορολογική βάση και χειροτέρευση των υπηρεσιών που προσφέρονται από το κράτος. Όμως υπάρχει και ένα θέμα ή δίκες και ίσης μεταχείρισης μεταξύ των κρατών μελών, γιατί ορισμένα κράτη αναπτύσσουν στρατηγικές για να αφαιρέσουν φορολογικά έσοδα από άλλα κράτη. Και αυτή τη στιγμή Βρισκόμαστε σε ένα όργανο που συζητάει το θέμα του δίκαιου, ισότιμου ανταγωνισμού κλπ. Και έχουμε μπροστά μα τεράστιε επιχειρήσει οι οποίε έχουν τη δυνατότητα να ξεφύγουν από τι φορολογικέ του υποχρεώσει. Αντίθετα με αυτό που συμβαίνει με μικρότερε επιχειρήσει ή με φορολογούμενου. Όταν μιλάμε για ελάχιστη φορολόγηση σε διεθνέ επίπεδο, θα πρέπει να λέμε αποτελεσματική φορολόγηση. Γιατί αλλιώς θα εξακολουθήσουμε να παίζουμε το ίδιο παιχνίδι με άλλους κανόνες. Ένα πράγμα έχει κατάσταση σαφές. Αυτοί που προτείνουν το συγκεκριμένο ψήφισμα υποστηρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει πρωτοβουλία σε αυτό το επίπεδο. Να μην δηλαδή καταλήξουμε ξανά στις ε, γνωστές ε, συνήθει δικαιολογίε, ότι ο αγώνας είναι δίκαιο, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και όλου του άλλου να συμφωνήσουν. Σα ευχαριστώ πολύ και ε, από τους μη εγγεγραμμένου, ο κύριος Λευτέρη Νικολάου Αλαβάνος που θα πάρει το λόγο. Ένα μισή λεπτό παρακαλώ. Τα περί δίκαιη φορολόγηση αποτελούν μέρος των σφοδρών αντιπαραθέσεων σχετικά με την επιβολή φόρων σε μονοπωλιακούς ομίλους τρίτων χωρών που ανταγωνίζονται ευρωενωσιακές επιχειρήσεις εμπορικοί πόλεμοι για τον έλεγχο τομέων της οικονομίας με μεγάλη κερδοφορία όπως η ψηφιακή οικονομία η ενέργεια οι λεγόμενες πράσινες επενδύσεις. το να μιλάτε σήμερα εδώ για δίκαιη φορολόγηση είναι ένα κακόγουστο αστείο αφού οι κρατικοί προϋπολογισμοί οι οποίοι ελέγχονται και επικυρώνονται από την κομισιόν συνιστούν μοιρασιά τη λίας των ομίλων σε βάρος του εισοδήματος των εργαζομένων έτσι στην ελλάδα με τον προπολογισμό τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, μισθωτοί και μικροί επαγγελματίε συνεισφέρουν στα φορολογικά έσοδα του κράτου κράτους 93% ενώ οι επιχειρήσεις 7%. Ταυτόχρονα μειώνεται η φορολογία των οικονομικών ομίλων από 28% σε 24% ενώ η φορολογία των μερισμάτων, των καθαρών κερδών δηλαδή των επιχειρηματιών, υποδιπλασιάζεται στο 5%. Την ώρα που συνεχίζεται η αφέμαξη των λαϊκών οικογενειών, επιβάλλονται κάθε λογής χαράτσια στις λαϊκές οικογένειες ενώ δίνονται ελαφρύνσεις στους βιομήχανους με τζάμπα ρεύμα που είναι πανάκριβο για το λαό με αφορολόγητο στους εφοπλιστές πετρέλαιο την ώρα που φορολογούνται οι φτωχοί αγρότες. αυτή είναι η νέα κανονικότητα που ευαγγελίζεται η τωρινή και υλοποιούσε η προηγούμενη κυβέρνηση. οι εργαζόμενοι τα λαϊκά στρώματα μαχητικά πρέπει να διεκδικήσουν ουσιαστική φορολόγηση των κερδών του κεφαλαίου κατάργηση των φοροαπαλλαγών αφορολόγητο όριο που να καλύπτει τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας κατάργηση των υψηλών πολύ άδικων έμεσων φόρων. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Γκιόρη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρόεδρε. Ναι, το γεγονός ότι και οι ψηφιακές επιχειρήσεις θα πρέπει να καταβάλουν φόρους. Δεν είναι δυνατόν το Google ε, και το Facebook ε, να μην ε, καταβάλουν τους φόρους. Θα πρέπει να βρεθούν διεθνείς λύσεις. Ο ΣΟΑ είναι μια δεδειγμένη πλατφόρμα εδώ. Ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο πυλώνες. Με το πρώτο πυλώνα συμφωνώ γιατί με τον τρόπο αυτό οι χώρες μέλη θα έχουν περισσότερα φορολογικά δικαιώματα. Δεύτερον, εκεί που θα πρέπει να θεσπιστεί ένας ελάχιστος φορολογικός συντελεστής. Ε, εδώ δεν συμφωνώ γιατί θεωρώ ότι δεν υπάρχει μια σχετική έρευνα εν σχέση με τις ε, επιπτώσεις ενός τέτοιου ε, συστήματος θέσπισης ελάχιστου φορολογικού συντελεστή και ενδεχομένως οι επιχειρήσεις θα μεταφέρουν τις έντρες τους σε άλλη χώρα. Ε, θα πάνε σε μια χώρα που θα έχουν τις ελάχιστες φορολογικές επιβαρύνσεις και με τον τρόπο αυτό θα υπονομεύσουμε την φορολογική μας ανταγωνιστικότητα και θα δημιουργηθούν νέες φορολογικές οάσεις. Ε, όταν ε, ε, ε, θα πρέπει καταρχήν να εκπονήσει κάποιες μελέτες σε σχέση με τις επιπτώσεις αυτού του συστήματος. Στο κείμενο αναφέρεται ότι η φορολογική πολιτική θα πρέπει να εναρμονιστεί. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα σχετικός προβληματισμός ε, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κάτι τέτοιο θα ζημίωνε την ευρωπαϊκή, τον ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί θα έφευγαν οι επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πολιτάγκ. Eh, eh, Ευχαριστώ πολύ κύριε ε, Πρόεδρε. Θα μιλήσω ε, Ολλανδικά αυτή τη φορά. Ε, γίγαντες ε, όπως η Netflix ή η Google ε, κερδίζουν εκατομμύρια και δεν πληρώνουν τίποτα, πληρώνουν ψίχουλα. Οι κυβερνήσεις και τα κόμματα είναι λογικό που θέλουν να επιβάλλουν ε, κάποιους ε, εθνικούς φορολογικούς συντελεστές και εθνικούς φόρους. Ωστόσο, ε, απειλούνται εν τέλει με εμπορικές κυρώσεις γιατί μπορεί αυτό να έχει επίπτωση και ακόμα και στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για την συζήτηση της μεταρρύθμισης. Χρειάζεται μεταρρύθμιση. Είναι απαρχαιωμένο το σύστημα ε, και οι χώρες ε, είναι διαρκώς υποχρεωμένες ε, να μειώνουν τα επίπεδα της φορολόγησης. Δεν είναι δυνατόν να υπομένουμε, να υποκύπτουμε συνέχεια στα όσα λένε οι Ηνωμένε Πολιτείε και προσπαθούν να επιβάλλουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Θα πρέπει οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει μεγάλες καταβάλει προσπάθειες. Η ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ε, θα πρέπει και εντός των συνόρων και εκτός των συνόρων να ακολουθούν την ίδια πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο ε, στον κύριο Πισλάρου. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Πρόεδρε, θα μιλήσω ρουμανικά. Κύριε Επίτροπε ε, Τζεντιλόνι, κυρία Πρόεδρε, κυρία ε, εισηγήτρια, είναι γεγονός ε, ότι η συζήτηση που έχουμε σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντική. Εγώ ε, όμως θα προσεγγίσω το θέμα με τρόπο διαφορετικό από ε, τους προλαλήσαντες συναδέλφους. Ε, ωστόσο, συμφωνώ ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υποστηρίξουμε το ψήφισμα. Στόχος μας δεν είναι να μεταχειριστούμε ή να θεωρήσουμε τις πολυεθνικές ως εχθρό του λαού, γιατί δημιουργείται μία εντύπωση σε Ευρωπαϊκή ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στις χώρες όσα γενικότερα ότι σημαντικά ποσά ε, χάνονται από την φορολόγηση λόγω της ε, πρακτικής ε, της μετακίνησης των κερδών από τη μία χώρα στην άλλη. Ε, βεβαίως σε πολλές χώρες ΩΣΑ, ε, αλλά κυρίως στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολίτες ακούν όλο και περισσότερο αυτό το αφήγημα. Αυτό που πρέπει να υπογραμμιστεί πάντως ε, είναι ότι πρόκειται για πρόβλημα δεοντολογίας. Ναι, αλλά υπάρχει και ένα πρόβλημα το οποίο σχετίζεται με τον ανταγωνισμό αλλά και με τον συντονισμό ανάμεσα στις χώρες μέλη. Οι χώρες, στην ουσ... οι, συγγνώμη, οι πολυεθνικές εταιρείες, επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ε, το πλαίσιο το οποίο έχουμε μεταξύ μας και το οποίο είναι ανεπαρκές και ακριβώς κινούνται εντός αυτού του πλαισίου. Ε, θα πρέπει να εναρμονιστούν τα φορολογικά συστήματα. Ε, ε, θα πρέπει επομένως να κινηθούμε με διτό τρόπο ένα δίκαιο ποσοστό φορολόγησης αφενός και ένα συντονισμένο πλαίσιο αφετέρου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει και μπορεί να δώσει το παράδειγμα. Δεν πρέπει να κηρύξουμε πόλεμο στις πολυεθνικές εταιρείε ε, ε, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα το οποίο θα δίνει την δυνατότητα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μην βρίσκονται σε δυσμενή ε, θέση και συγκριτικά να υφίστανται μεγαλύτερο κόστος και θα πρέπει οι σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών να είναι καλά περιγραμμένες. Να μην λησμονούμε τα όσα υπάρχουν ήδη στην πρόταση. Θέλουμε ένα σύστημα απλό, ένα σύστημα το οποίο να προβλέπει ε, τις ε, καταστάσεις και να μην δημιουργεί στρέβλωση του ανταγωνισμού. Ο κύριος Ερνέστ Ουρτασούν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, Καλώς ορίζουμε αυτή τη συζήτηση και το ψήφισμα που θα υιοθετηθεί αυτή τη εβδομάδα. Είναι σημαντικό να παίξουμε κέριο ρόλο στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το πώς θα φορολογείται η ε, πώς αφορολογούνται οι ψηφιοποιημένες ε, ψηφιακές επιχειρήσεις. Ε, αυτή η πρόταση όμως ξεπερνάει αυτό το στόχο και έχει ως στόχο να προσαρμοστεί το φορολογικό σύστημα στον 21ο αιώνα. Οι κανόνες μας αυτή τη στιγμή προέρχονται από τον 20ο αιώνα. Μεταφορές μεταξύ θηγατρικών αυτή τη στιγμή φορολογούνται σαν να πρόκειται για μεταφορές μεταξύ ανεξάρτητων εταιριών. Αυτό αποτελεί το σημείο εκκίνησης ε, ε, μια σειράς ε, τακτικών φορολογικής φοροδιαφυγής. Θα μπορούσαμε να βασιστούμε στην αρχή ότι κάθε επιχείρηση με τις θηγατρικές της θα φορολογείται ως μια ενιαία οντότητα. Ο ήδη ξεκίνησε ε, τις με μια πρώτη πρόταση η οποία μπλοκαρίστηκε και μπλοκαρίστηκε και η δεύτερη πρόταση του ΩΣΑ το 2016. Χρειαζόμαστε διεθνείς διαπραγματεύσεις ε, για να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα μέχρι το τέλος του 2020. Όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να βάλουν στην άκρη τις διαφορές τους και να μιλήσουμε με μία ενιαία φωνή. Και χρειαζόμαστε και φιλοδοξία, όχι τον ελάχιστο κοινό παρανομαστή. Για να εξασφαλίσουμε ότι ε, οι επιχειρήσεις θα φορολογούνται εκεί που έχουν την οικονομική τους δραστηριότητα εκεί που ε, κερδίζουν χρήματα, εκεί που έχουν πελάτες, εκεί που υπογράφουν συμβάσεις, εκεί που έχουν προσωπικό. Ε, οι, οι προσδοκίες των πολιτών είναι ψηλές. Αν δεν καταφέρουμε να τους ικανοποιήσουμε, ε, θα αποτύχουμε και θα καταστραφούν και τα φορολογικά μας συστήματα. Θα πρέπει να δράσουμε από κοινού για να επιτύχουν οι διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ. E, Κύριε Μακάρτη, ευχαριστώ πολύ. Όπως είπαν και άλλοι ομιλητές, υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία στην πρόταση του ΩΣΑ. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι ε, τα φορολογικά δικαιώματα ε, θα πρέπει να ε, θα πρέπει να κατοχυρωθούν ε, ωστόσο είναι αναγκαίο ε, να δούμε ότι η προσέγγιση του ΩΣΑ τελικά μπορεί να χαμηλώσει τα ποσοστά αποφυγής μόνο κατά 5%. Ε, είναι οι δύο πυλώνες αυτών των προτάσεων, εάν συμφωνηθούν στο μέλλον, ε, θα σημάνουν μια ουσιαστική μετατόπιση προς ένα πιο βιώσιμο και πιο δίκαιο σύστημα. Εγώ προειδοποιώ την ίδια μου κυβέρνηση ότι ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσει το ζήτημα της ε, φοροαποφυγής των ε, πολυεθνικών ομίλων, για παράδειγμα στη Silicon Valley χρειάζεται μια νέα στρατηγική. Είναι... Οι περισσότεροι θεωρούν ότι ένα τόσο άδικο σύστημα είναι δυστυχώς αναπόφευκτο. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Βέρα ε, Δελκαστίγιο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, οι ψηφιακές τεχνολογίες της σήμερα ε, πλέον δεν είναι απλώς, ε, ε, ε, στοιχείο της οικονομικής εικόνας, αλλά πρωταγωνιστές. Είτε πρόκειται για την μεταποιητική βιομηχανία, είτε πρόκειται για τη γεωργία, τον τουρισμό, την ενέργεια κλπ. Κατά την έννοια αυτή, μία, ένα φορολογικό ε, πλαίσιο σαν αυτό που έχουμε τώρα ε, βρίσκεται πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Ε, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες παράγουν οικονομική αξία. Αυτό είναι αλήθεια ωστόσο. Υπάρχουν και πολλές ε, εταιρείε οι οποίες ε, χρησιμοποιούν ε, τις άειλες, τα άειλα κέρδη τους ή το άειλο ενεργητικό. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε έναν ψηφιοποιημένο κόσμο και επομένως θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τον, την φορολόγηση. Βεβαίως πρώτα θα πρέπει να μεταρρυθμίσουμε και το νόμο του ανταγωνισμού, το πλαίσιο του ανταγωνισμού. Τούτη τη στιγμή μιλάμε φυσικά για τα φορολογικά. Ωστόσο θα πρέπει πρώτα να ξεκινήσουμε την ε, μεταρρύθμιση των αρχών που διέπουν την, ε, τον ανταγωνισμό. Ε, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και την φορολογική μεταρρύθμιση. Αυτό θα έχουμε τη δυνατότητα βέβαια και την ευκαιρία να το συζητήσουμε και αργότερα στα πλαίσια της θητείας αυτής. Μη και κάτι ουσιαστικό, δηλαδή αυτήν την όθηση που δίνει η ηγεσία και που θα πρέπει να έχουν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς επίσης και οι διαδοχικές προεδρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύρια Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όλες και όλοι ακούσαμε ε, να γίνεται λόγος ε, τα τελευταία χρόνια για πολλά ε, φορολογικά σκάνδαλα οι πολυεθνικές ε, στην ουσία ε, ξεγλιστράνε χρησιμοποιώντας ε, τα διαφορετικά φορολογικά μας συστήματα. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε πολλές διαφορές όσον αφορά τα φορολογικά πλαίσια μας. Άκουσα προηγουμένως έναν συνάδελφο που έλεγε ότι δεν θα πρέπει να βλέπουμε τις πολυεθνικές ως εχθρούς. Δεν λέμε κάτι τέτοιο, αντιθέτως λέμε ότι και οι πολυεθνικές θα πρέπει να συμμετέχουν ε, ε, στα κοινά ε, με τον αναλογούντα δίκαιο φόρο. Ένα δις κάθε χρόνο χάνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω αυτής της φόρο αποφυγής και της φορολογικής απάτης. Θα μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε με τα χρήματα αυτά την οικολογική μετάβαση που είναι απολύτως απαραίτητη. Βεβαίω βεβαίως ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, και ότι το 2,0 είναι απλώς κάτι απολύτως λογικό. Ε, λέει ότι θα πρέπει και σε παγκόσμιο επίπεδο να υπάρξει ένα ελάχιστο ποσοστό φορολόγησης και η φορολόγηση να, και, να πληρώνουν όλοι ένα δίκαιο ποσοστό. Αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Αγαπητοί συνάδελφοι, η φορά και το γεγονός ότι είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοιο φαινόμενο είναι σκανδαλώδης. Πάρα πολλοί άνθρωποι στην Ευρώπη ε, έχουν την ε, ευθύνη να ε, εισπράττουν ε, φόρους. Ε, η ευθύνη θα πρέπει να ανάληψη ευθύνη θα πρέπει να ισχύει για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Πολλές επιχειρήσεις δεν καταβάλουν σωστά τους φόρους. Γιατί όμως υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες φοροαποφυγής. Εναπόκειται σε εμάς του πολιτικούς να κλείσουμε αυτές τις ε, τρύπε και να επιβάλλουμε μια δίκαιη φορολογική πολιτική στις μεγάλες επιχειρήσεις. Ε, η Ευρώπη χάνει δισεκατομμύρια ευρώ ε, θα πρέπει η Γερμανική ε, Προεδρία του Συμβουλίου το 2021 να κάνει σημαντικά βήματα εδώ. Θα πρέπει να φέρουμε την Ευρώπη στο επίπεδο του 21ου αιώνα. Ε, χρειαζόμαστε σημαντικές ε, απαντήσεις σε μείζωνα ερετήματα ε, και σε σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Χρειαζόμαστε ένα ελάχιστο φορολογικό συντελεστή και στις με τον ΩΣΑ θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια συμφωνία μέχρι το τέλος του 2020. Εάν όχι θα πρέπει να κάνουμε μια πρόταση νομοθεσίας για μια δίκαιη φορολόγηση της ψηφιοποιημένης οικονομίας, για μια σωστή κατανομή των ευθυνών δαπανών, ούτω ώστε η Ευρώπη να αποκτήσει ένα πιο οικολογικό και κοινωνικό πρόσωπο. Γιατί μόνο έτσι θα επιτευχθεί η κοινωνική δικαιοσύνη μέσω τη φορολογική δικαιοσύνη. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Φερέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι πολυεθνικές εταιρείες ε, γλιτώνουν 500 ε, εισπράττουν 500 δισεκατομμύρια ευρώ ε, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ε, μέσω φόρων για να ελαφρυνθούν οι υπόλοιποι φορολογούμενοι και να βελτιωθούν οι υποδομές των χωρών μας. Οι φιλελεύθερες πολιτικές περί της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίου, της με, ελεύθερης μετακίνησης επιχειρήσεων έχουν οδηγήσει σε αυτό το φαινόμενο. Οι προτάσεις που έχουμε εγκρίνει ε, για ένα νέο σύστημα φορολογής των επιχειρήσεων ε, δεν έχουν επηρεάσει πολλές από αυτές τις πολυεθνικές. Διότι με τη χρήση φορολογικών ε, παραδείσων επιτρέπουν τον εαυτό τους να εξακολουθούν να διαφεύγουν και να φοροαποφεύγουν. Πολλά πρέπει να γίνουν για να καταπολεμηθεί το φαινόμενο. Αυτό και η φορολογική απάτη. Η μάχη δεν περνάει μόνο από την εναρμόνιση θα πρέπει να σεβαστούμε την κυριαρχία των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Ωραία. Ο λόγος στην κυρία Τάλερ. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η αγορά ποτέ δεν ε, περίμενε η διοίκηση να δημιουργήσει τις ε, ε, το κατάλληλο πλαίσιο για τις ε, δικές του εξελίξεις, δηλαδή τις εξελίξεις της αγοράς. Και το γεγονός αυτό οδηγεί σε κάποια νομικά κενά από τα οποία υποφελούνται οι πολυεθνικοί όμιλη και ταυτόχρονα μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες επομίζονται το φορολογικό βάρος, κάτι το οποίο είναι εντελώς άδικο. Εγώ η ίδια εδώ και 12 χρόνια είμαι επιχειρηματίες, γι' αυτό μπορώ να παρακολουθήσω, να αισθανθώ πολύ σωστά αυτή την κατάσταση. Ε, ε, ε η των ΟΣΑ είναι υπό εξέλιξη και θεωρώ ότι θα πρέπει να επισημάνουμε κάποια πράγματα. Θα πρέπει να απομακρυνθούμε από παροχημένες ε, αντιλήψεις ότι μόνο η φυσική παρουσία των επιχειρήσεων είναι ικανή προϋπόθεση φορολόγησης. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι η οικονομία μας θα ψηφιοποιείται όλο και περισσότερο. Γι' αυτό χαίρομαι για την πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου και πραγματικά θα υπερψηφίσω το ψήφισμα. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μάρεκ Πέλκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Λένε ότι δύο πράγματα είναι σίγουρα στον, στον κόσμο. Ο θάνατος και οι φόροι. Ε, βεβαίως... Ε, Ακούσαμε και όλες αυτές τις ιστορίες για τα Lux, Leaks και λοιπά. Ε, το BEPS δεν έχει κάνει και πολλά πράγματα ε, και ε, βεβαίως από τις προτάσεις που κάνει ο ΩΣΑ θα πληγούν το Facebook, Google και άλλα ψηφιοποιημένα και ιντερνετικά ε, μορφήματα, μορφώματα. Ε, θα πρέπει να δράσουμε πάντως από κοινού και μάλιστα σε διεθνές επίπεδο. Γι' αυτό θα πρέπει να ε, πείσουμε τις Ηνωμένε Πολιτείες ότι θα πρέπει να φορολογείται οποιαδήποτε αξία δημιουργείται. Βεβαίω και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πείσουμε και τους συνήθεις υπόπτους να λειτουργήσουν σωστά εάν ε, οι διαβουλεύσεις ε, σε εθνικό επίπεδο δεν ε, επιτύχουν μέχρι το τέλος του 2020, η κυρία Φόντερ Λάγεν έχει υποσχεθεί ότι θα πρέπει να μας υποσχεθεί ότι θα προχωρήσει μια ευρωπαϊκή λύση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ρέγνερ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ αξιότιμε κύριε πίτροπε. Εάν θέλουμε να δούμε τα πράγματα σωστά, τα ΠΕΠΣ θα μας φέρουν στον 21ο αιώνα. Και αυτό είναι σημαντικό. Η ε, φόρη είναι μια επένδυση στις ε, υποδομές. Οι επιχειρήσεις θέλουν να έχουν ε, κέρδη, αλλά θα πρέπει να εισφέρουμε το δικό τους μερίδιο στη φορολόγηση. Οι φόροι θα πρέπει να πληρώνονται εκεί που σημειώνονται κέρδη το Facebook, η Google κλπ. θα πρέπει να πληρώνουν κανονικά τους φόρους τους, γιατί τα χρήματα αυτά θα πρέπει να πάνε στα δημόσια ταμεία. Το Facebook δεν πληρώνει φόρους στην Αυστρία παρά τα τεράστια κέρδη. Ε, και ενώ άλλες επιχειρήσεις καταβάλουν ε, σωστά τους φόρους τους. Αυτό είναι εντελώς άδικο και είναι ξεκάθαρο για να λειτουργήσει το ΠΕΠΣ χρειαζόμαστε διαφάνεια. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι όμιλοι καταβάλουν φόρους και ποιοι όχι. Ε, ε, θα πρέπει να έχουμε ε, φορολογικούς καταλόγους. Η Αυστρία υπερψήφισε την άρση των υφιστάμενων ε, φραγμών ε, προκειμένου να υπάρξει μια μεγαλύτερη διαφάνεια. Και το ίδιο θα πρέπει να γίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέσπιση ελάχιστο φορολογικού συντελεστή 18% μόνο έτσι μπορούμε να καταπολεμήσουμε το, dumping, το φορολογικό dumping προς τα κάτω. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μαργαρίδα Μάρκες. Ένα λεπτό. Θα μιλήσω στα πορτογαλικά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ε, η συζητήση των ΩΣΑ είναι μια ευκαιρία να απαντήσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο σε αυτό το πρόβλημα της φορολόγησης ε, στην ψηφιακή εποχή. Ε, ό,τι αποφασιστεί θα αλλάξει τις φορολογικές αρχές της παγκόσμιας οικονομίας. Η συζήτηση προχωράει προς τη σωστή κατεύθυνση, παρόλο ότι πολύ αργά και καθυστερημένα. Ένας ελάχιστος φορολογικός ε, συντελεστής ε, που προτείνεται για κάθε μια φορολογική δικαιοδοσία ε, είναι μια πολύ καλή ιδέα. Εν τω μεταξύ, ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο θα προχωρήσει στις δικές του προτάσεις. Όμως η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι διαπραγματεύσεις για αυτούς τους δύο πυλώνες θα γίνουν παράλληλα. Τέλος, ελπίζουμε ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία κατά τη διάρκεια του 2020, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου. Αυτή η συμφωνία είναι απολύτω απαραίτητη για να εξασφαλίσουμε καλύτερη φορολογική δικαιοσύνη και κοινωνική δικαιοσύνη στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στο Catch the Eye. Δύο άτομα έχουν ζητήσει το λόγο. Οι φορολογικέ ε, πολιτικέ θα πρέπει να ευνοούν την πλειοψηφία των πολιτών. Και όλοι θα πρέπει να πληρώνουν φόρους με τους ίδιους κανόνες. Και οι φόροι θα πρέπει να πληρώνονται εκεί που δημιουργούνται τα έσοδα και τα κέρδη. Η φορολογία, οι φόροι επιτρέπουν τη χρηματοδότηση κρατικών πολιτικών. Οπότε ψηφίζω και με τα δύο χέρια υπέρ του ψηφίσματο που ζητάει οι επιχειρήσει να πληρώσουν φόρου εκεί που εισπράττουν ε, τα κέρδη του. Αυτό είναι σημαντικό για να αναπτυχθεί η Ευρώπη όπω πρέπει. Ευχαριστούμε πολύ. Δύο συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Τσίποχάτρου πρώτα. Okay. Uh, Mr. Kelleher. Uh, thank you. Well, I will be... Ευχαριστώ. είναι κάτι το οποίο με προβληματίζει από πολλέ απόψει, αλλά εγώ θα ήθελα να επισημάνω το εξή. Στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ό,τι αφορά την μονομερή τη ε, δράση, σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια ότι μπορούμε να φέρουμε την δίκαιη φορολόγηση και την παγκοσμιοποιημένη φορολόγηση χωρί να εμπλακεί στη συζήτηση ο υπόλοιπο κόσμο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί αυτό υπονομεύει την ανταγωνιστικότητά μα ω Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποθαρρύνει τι επενδύσει προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να είμαι σαφή, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, παλεύει να ανταγωνιστεί τον υπόλοιπο κόσμο και αγκομαχά σε ό,τι αφορά την παγκόσμια οικονομία. Έχουμε ε, μερικέ ε, πολυεθνικέ που ξεκίνησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τελικά κατάφεραν να μεγαλώσουν και να ευοδοθούν παγκοσμίω. Όμω η ιδέα ότι μπορούμε εμεί μόνοι μα, μονομερό, να ε, δράσουμε χωρί να εμπλέξουμε του εταίρου μα, είναι κάτι που υπονομεύει την ανταγωνιστικότητά μα και αποθαρρύνει τι πολυεθνικέ ε, να απασχολήσουν Ευρωπαίου πολίτε. Ευχαριστώ. Η συζήτηση για αυτό το θέμα τελειώνει με τον Επίτροπο, τον κύριο Τζεντιλόνι. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συζητήσαμε σήμερα το απόγευμα ένα θέμα που θα είναι κρίσιμο τα επόμενα χρόνια για την Ένωσή μας. Και βέβαια και για τη βιωσιμότητα της ενιαίας αγοράς και του κοινωνικού μας μοντέλου. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι η συζήτηση ήταν χρήσιμη. Θέλω απλώς να τονίσω Δύο σημεία. Πρώτον, η δική σας υποστήριξη, η υποστήριξη του Κοινοβουλίου θα είναι κρίσιμη τα επόμενα χρόνια. Απολύτως κρίσιμη. Αν θέλουμε να διασφαλίσουμε μια πραγματική μεταρρύθμιση. Δεύτερον, η Κομισιόν εργάζεται προσπαθώντας να πετύχει μια κοινή θέση στο τραπέζι του ΟΣΑ. Πρέπει να συνεργαστούμε με την Προεδρία, διότι επισήμως αυτοί γούνται τις συγκεκριμένες συζήτηση. Νομίζω ότι θα έχουμε πολύ καλή συνεργασία και με την Κροατική και μετά με την Γερμανική Προεδρία. Να είμαι ξεκάθαρος. Είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στην εξέβρεση μιας συνολικής παγκόσμιας λύσης. Δεν είναι κάτι που κάνουμε χωρίς πραγματική αφοσίωση. Παρά τις ε, δυσκολίες ε, αυτές, αυτή την εποχή, που υπάρχουν στις πολυμερείς διαπραγματεύσεις, ε, τις οποίες γνωρίζουμε και να αναγνωρίζουμε, ε, ε, παραμένουμε πλήρως αφοσιωμένοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε και εναλλακτικέ βέβαια. Όπως είπα προηγουμένως, αυτό που μου ανέθεσε ο πρόεδρος ήταν να εργαστώ επ' αυτή την, επ αυτής της παγκόσμιας λύσης, να βρω τα εργαλεία με μεγάλη αφοσίωση και αν είναι δυνατό να βρω και τον ευρωπαϊκό τρόπο που θα πετύχουμε κάτι τέτοιο. Για να βρούμε αυτόν τον τρόπο πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο. Κλείνει τώρα η συζήτηση. Ε, θα γίνει την Τετάρτη η ψηφοφορία. Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ε, όμως πριν πάμε στο επόμενο θέμα διακόπτουμε για λίγο την συνεδρίαση. Πείτε. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση της κυρίας Ρετζιμέντη η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ιορδανία, στο χασιμητικό βασίλειο της Ιορδανίας. Η κυρία Ρετζιμέντη ως εισηγήτρια έχει το λόγο. Καλησπέρα, Πρόεδρε, συνάδελφε, κύριε Επίτροπε. Το να παίρνω το λόγο στην Ολομέλεια ως εισηγήτρια για αυτό το σημαντικό φάκελο είναι μεγάλη μου τιμή. Είμαι πολύ ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα στην Επιτροπή ΙΝΤΑ και από την ομόφωνη ψηφορία της έκθεσης που παρουσίασα και συνέστησα το να χορηγηθεί μία τρίτη χρηματοοικονομική βοήθεια 500 εκατομμυρίων ευρώ στο χασμητικό βασίλειο της Ιορδανίας. Για να φτάσω σε αυτό το συμπέρασμα χρειάστηκε να αναλύσω με προσοχή την οικονομική και κοινωνική κατάσταση της Ιορδανίας και να σημειώσω τις αξιέπαινες προσπάθειες που κάνει η χώρα αυτή σε ό,τι αφορά την υποδοχή των προσφύγων και την καταπολέμηση της Ισλαμικής τρομοκρατίας. Αλλά ε, και στην διαχείριση των προηγούμενων δανείων που δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση από τις αξιολογήσεις που έγιναν ε, για την υλοποίηση των προηγούμενων προγραμμάτων μακροοικονομικής βοήθειας που δόθηκαν στην Ιορδανία προκύπτει ότι τα κονδύλια που δόθηκαν ε, υπό τη μορφή δανείων χαμηλότοκων μακροπρόθεσμα συνεισέφεραν στο να διατηρηθεί η μακροοικονομική σταθερότητα της χώρας και είχαν κυρίως ένα θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Τα προγράμματα υλοποιήθηκαν αποτελεσματικά και σε στενό συντονισμό με τις αρχές της Ιορδανίας ε, εν όψιον της ε, χαμηλής ανάπτυξης ε, και των μειούμενων επενδύσεων στις 11 Ιουλίου 2019 οι αρχές Ιορδανίας ζήτησαν περαιτέρω κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες ανάγκες της χώρας σε ό,τι αφορά την εξωτερική χρηματοδότηση και του ισοζυγίου που σχετίζεται με τις συνθήκε αστάθεια τη περιοχή, ε, μεταξύ των οποίων παρουσία στην Ιορδανία ενός ε, υψηλού αριθμού προσφύγων από τη Συρία. Στις 6 Σεπτεμβρίου 2019, η Επιτροπή υιοθέτησε πρόταση για ένα τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης ε, μέχρι τα 500 εκατομμύρια ευρώ θεωρώ ότι λαμβάνοντα υπόψη τι προσπάθειε τη Ιορδανία για την καταπολέμηση τη μεταναστευτική κρίση και την καταπολέμηση τη τρομοκρατία και διαπιστώνοντα την ανάπτυξη σε ό,τι αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημοκρατία, αυτό το δάνειο αποτελεί μια προσθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θα βοηθήσουμε μια χώρα τη γειτονία που έχει μεγάλη γεωπολιτική σημασία να διαχειριστεί κοινωνικά και κοινωνικά προβλήματα σημαντικά. Ε, η σύραξη της ε, Συρίας ε, είχε αρνητική οικονομική επίπτωση στην Ιορδανία λόγω της διακοπής του περιφερειακού εμπορίου, της μείωσης των εσόδων του τουρισμού και της επιδείνωσης της εμπιστοσύνης των επενδυτών και της μείωσης των ισρών κεφαλαίου στην περιοχή. Η πίεση που ασκήθηκε στις δημόσιες υπηρεσίες της Ιορδανίας, κυρίως σε ό,τι αφορά τον τομέα της υγείας, σε πρόσβαση στην εκπαίδευση και σε βασικά αγαθά, είναι δύσκολο να υποστηριχθεί από τη χώρα και πρέπει να αναγνωρίσουμε παρόλα αυτά την αξιέπαινη προσπάθεια στο να εξασφαλίσει ε, μια αξιοπρεπή υποδοχή στους πρόσφυγες και για τους οποίους, παρά τις πολυάριθμες δυσκολίες, εγγυάται σήμερα την πρόσβαση σε δημόσια υγειονομική περίθαλψη και στην αγορά εργασίας. Θεωρώ επίσης ότι είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη τις προσπάθειες της Ιορδανίας στην καταπολέμηση της Ισλαμικής τρομοκρατίας, προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Η Ιορδανία είναι στρατηγικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συνεργασία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της εμπορίας όπλων αλλά και της ανταλλαγής προσωπικών δεδομένων μεταξύ Ευρωπόλ και των αρμοδίων αρχών της Ιορδανίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Το βασίλειο της Ιορδανίας συνεχίζει ε, να σέβεται τις ε, δημοκρατικές αρχές, να προωθεί την ε, θρησκευτική ειρηνική συνύπαρξη και να υποστηρίζει την ανεξιθρησκεία ε, ε, και κάνει σημαντικά βήματα προς τα μπρος για την προστασία των ενηλίκων και των δικαιωμάτων των γυναικών. Επίσης, χάρη στην προοδευτική απελευθέρωση των αμοιβαίων αγορών, η παρουσία ενός σταθερού εξωτερικού εταίρου αποτελεί εγγύηση και για τις ε, επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, γιατί δίνονται περισσότερες ευκαιρίες για το εμπόριο, την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις στην Ιρδενία. Θα ήθελα να πω ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η οικονομική βοήθεια θα πρέπει να είναι στοχευμένη στο να ενθαρρύνει την ανάπτυξη των επιχειρηματικών επενδύσεων και των προγραμμάτων στη χώρα. Επίσης, είναι απαραίτητο να εγγυηθούμε με όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας ένα κατάλληλο έλεγχο των κονδυλίων, προκειμένου να υπάρχει μια διαφανής και ορθή χρήση τους. Θεωρώ επομένω ότι είναι απαραίτητο να δείξουμε με αυτή την ενίσχυση της υποστήριξη, την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωση σε μια χώρα όπως η Ιορδανία και εύχομαι ότι η βοήθεια θα μπορέσει να δοθεί σύντομα. Εύχομαι η αυριανή ψηφοφορία να επιτρέψει τη χορήγηση της ε, χρηματοοικονομικής βοήθειας στο Χασαμιτικό Βασίλειο τη Ιορδανία. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια να σας πω ότι μιλήσατε 1,5 λεπτό παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Ε, θα πρέπει μόνο 20 λεπτά, 20 δευτερόλεπτα λιγότερη να είναι η συζήτηση. Ο Επίτροπος έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια την κυρία Ρετζιμέντη και την Επιτροπή Ίντα για την ε, πολύ καλή αυτή έκθεση και για το πνεύμα συνεργασία. Ευχαριστώ και την Επιτροπή Προλογισμών και την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για τη στήριξή του. Πρέπει να υπενθυμίσουμε εδώ το ιστορικό της Ιορδανίας. Από το 2011 η οικονομία έχει πληγεί σημαντικά από τις ε, περιφερειακές ταραχές, ιδίως ό,τι αφορά το γειτονικό Ιράκ και τη Συρία, που έχει οδηγήσει σε απρόσμενες και απροσδόκητες, ε, απροσδόκητους οικονομικούς κλειδονισμούς. Παρότι υπάρχουν και διθρωτικές αδυναμίες ε, και έλλειψη ανταγωνιστικότητα που υπήρχαν και πριν το 2011. Αυτή λοιπόν η αναταραχή έχει πλήξει την ανάπτυξη και έχει ε, δυσκολέψει πολύ τα δημοσιοοικονομικά. Και ο πόλεμος στη Συρία έχει επηρεάσει πολύ την Ιορδανία γιατί οδήγησε σε εισρωή 1,3 εκατομμυρίων ε, Σύρων στη χώρα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αυξάνει την πίεση στα δημοσιονομικά της Ιορδανίας, στις δημόσιες υπηρεσίες και στις υποδομές. Σε αυτές τις δύσκολες ε, συνθήκες η Ιορδανία έχει καταφέρει μέχρι τώρα να διατηρήσει τη μακροοικονομική της σταθερότητα χάρη σε μια κατάλληλη ε, ανταπόκριση και διεθνή στήριξη. Τούτων λεχθέντων και κατόπιν αιτήματο των Ιορδανικών Αρχών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε στι 6 Σεπτεμβρίου μια πρόταση για νέο πρόγραμμα μακροοικονομική αρρωγή προ την Ιορδανία ύψου 500 εκατομμυρίων ευρώ ε, εν είδη δανείου. Ε, βάσει των δύο προηγούμενων προγραμμάτων, που έχουν υλοποιηθεί επιτυχώς. Η νέα αυτή η οικονομική αρρωγή θα βοηθήσει την Ιορδανία να ε, βελτιώσει την οικονομική της κατάσταση χάρη στους ελκυστικούς όρους του δανείου και να προωθήσει τις διαθετικές μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για την ε, ανάπτυξη και την αντοχή της οικονομίας της. Όλα αυτά εντάσσονται σε μια ευρύτερη ε, προσπάθεια για στήριξη προς την Ιορδανία. Φυσικά, εδώ υπάρχει και αιρεσιμότητα, βασίζεται σε ένα σύνολο μέτρων που θα συμφωνηθούν σε ένα μνημόνιο κατανόησης και σίγουρα θα υπόκειται η χώρα και σε αναθεωρήσεις και αξιολογήσεις του προγράμματος. Το πρόγραμμα αποτελεί μία σαφή ερμηνεία και ένδειξη της ε, δέσμευση τη Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξει την Ιορδανία σε μια περιοχή που συνεχώς παρουσιάζει ε, ταραχές ή προβλήματα και μεταβλητότητα. Αυτό θα δει, αποστείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, τηρεί τις δεσμεύσεις της και εξακολουθεί να βρίσκεται στο πλευρό της Ιορδανίας και σε, στο πλευρό όσων ζουν σε αυτή τη χώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον ε, Επίτροπο. Ξεκινάει η συζήτηση εκ μέρους ε, των πολιτικών ομάδων. Πρώτος έχει το λόγο ο κύριος Ντέιβιτ Μακάλιστερ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, κύριε Επίτροπε, Επιτρέψτε μου λίγες ε, παρατηρήσεις από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για αυτό το θέμα. Ακούσαμε την εισηγήτρια και τον Επίτροπο να λέει πως η Ορδανία είναι ενώπιον τεράστιων προκλήσεων, μειώνεται η ρυθμή ανάπτυξης, αυξάνεται η ανεργία και ειδικά στους νέους. Ήδη ε, υπάρχουν πολλά πράγματα που οδήγησαν σε αυτό. Είναι η γειτονική χώρα ε, Συρία, όπως και το Ιράν, ε, που πλήττονται και αυτές όπως και η Ορδανία από το είναι σε και το εμπόριο των όπλων. 1,3 εκατομμύρια επίσης Σύριοι έχουν προσφύγει στην Ιορδανία. Είναι τεράστια λοιπόν η επιβάρυνση στον προπολογισμό της χώρας. Είναι ε, παρόλα αυτά υποδειγματική η αντίδραση της χώρας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει αυτή τη μακροοικονομική χρηματική υποστήριξη των 500 εκατομμυρίων ευρώ όπως διαπιστώσαμε επιτόπου στην Ιορδανία και όπως είπε και ο Επίτροπος Τζεντιλόνι το Κοινοβούλιο πρέπει να ακολουθήσει την πρόταση της Κομισιόν για να μπορέσει ο εταίρος μας, ο σύμμαχός μας η Ορδανία, να ανταποκριθεί σε αυτές τις ε, προκλήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κώστας Μαυρίδης έχει το λόγο. Δεν είναι εδώ. Επόμενος ομιλητής ε, ε, <clears throat> ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, εξ ονόματος της ομάδας ε, Renew, θα ήθελα να υποστηρίξω τη χορήγηση αυτής της τρίτης μακροοικονομικής ενίσχυσης στην Ιορδανία. Θεωρούμε ότι θα μπορούσε να συνεισφέρει στο να υποστηρίξει τη χώρα αυτή στις προσπάθειές της για να καταπολεμήσει την αστάθεια που δημιουργείται από την Συριακή Κυβέρνηση στην περιοχή. Υπενθυμίζουμε επίση ε, ότι υποστηρίζουμε ένθερμα την πολιτική γειτονία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, που είναι επίση ε, σημαντική για τη σταθερότητα τη Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Όμω, Παρόλο που υποστηρίζουμε επί της ουσίας το έτοιμο αυτό, λυπόμαστε που βρίσκεται στα χέρια μια εισηγήτριας που προέρχεται από ε, ένα κόμμα της ακροδεξιάς, ταυτότητα και δημοκρατία. Εμείς στην ομάδα Renew ε, θέλουμε να δηλώσουμε αποφασισμένοι Ευρωπαίοι δεν ισχυρά σε αυτό το ημικύκλιο ότι απορρίπτουμε τις ευρωσκεπτιστικέ ιδέες που είναι καταστροφικές ε, και διαχέονται από την ακροδεξιά. Ε, θέλουμε να πούμε ότι αυτή η πολιτική οικογένεια χαρακτηρίζεται από έλλειψη συνοχής, ε, γιατί από τη μία υποστηρίζει τον Μπασαρελεσάτη και από την άλλη δέχεται να βοηθήσει τα κύρια θύματά του. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει ο, ο κύριος ε, Τιερή Μαριανή. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου αρχικά να χαιρετήσω την ποιότητα του έργου της κυρίας Ρετζιμέντη που παρουσίασε αυτή την έκθεση. Πολύ σωστά αναφέρει πόσο αποδιοργάνωσε την Ιορδανική κοινωνία η κρίση στη Συρία. Ε, μια κοινωνία που ήδη αντιμετώπιζε σημαντικές προκλήσεις ε, με πληθυσμό που προέρχεται από την Παλαιστίνη, με ισχυρή παρουσία των αδελφών μουσουλμάνων είναι μία από τις ε, πιο βασικές και ισχυρέ δυνάμεις οικονομικά μιλώντας στην ευρύτερη περιοχή. Έχει διατηρήσει το νομισμά της, έχει αυξήσει τουριστική δραστηριότητα. Η Λουίς ε, Ρετζιμέντη αναφέρει ε, και την ανάπτυξη που υπήρχε μέχρι τώρα. και η Ιορδανία αντιμετώπισε πολύ σωστά τους χριστιανούς της Ιορδανίας. Πρέπει λοιπόν να επωφεληθεί μιας διεθνούς ε, συνδρομής ε, η Ορδανία ε, για να βρουν έναν τόπο να ξαναχτίσουν τις ζωές τους όσοι προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και από τον ISIS. Η χώρα αυτή έχει απομειστεί τις επιπτώσεις μιας διεθνούς κρίσης και ένα πολέμου για τον οποίο δεν ευθύνεται. Πώς μπορούμε να ε, εξηγήσουμε ότι δεν θα υπάρξει καμία υλοποίηση κανενό ε, προγράμματο κατάσταση σύρων προσφύγων. Έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε μια στρατηγική πολιτική που είναι απαραίτητη και εμεί είμαστε φυσικά ευνοϊκά διακείμενοι προ την ε, έκθεση αυτή. Ευχαριστούμε. Στα πλαίσια της διαδικασίας ΚΑΤΣΙΔΙΑΗ έχουμε Ε, μία, ένα αίτημα για να μιλήσει ένας ομιλητής. Ο κύριος Τουντοράκη, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Είμαι ο κύριο ο κύριος Τσουχαντάρου. Ε, πήγε στο νοσοκομείο σπευμένος. Ε, θεωρούμε ότι η ζωή δεν θα πρέπει να εξαρτάται από πολιτικά θέματα, θα πρέπει να είναι ένα δικαίωμα ανεξάρτητα από το πολιτικό χρώμα ε, και μπορώ να σας πω ότι οι πολίτες στην Ιορδανία χρειάζονται αυτό το δάνειο για να μπορέσουν να επιβιώσουν, για να έχουν πρόσβαση στη υγειονομική περίθαλψη και εμείς ε, θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί πρόκειται για έναν εταίρο που πραγματικά σέβεται τις ευρωπαϊκές αξίες. Εγώ θα ψηφίσω και με τα δύο χέρια υπέρ της πρότασης αυτής. Ευχαριστούμε, Επίτροπος έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα απλώς να υπογραμμίσω το γεγονός ότι το Συμβούλιο έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι θα εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εφόσον το αυτό εγκρίνει την θέση του στην πρώτη ανάγνωση άμεσα και η διαδικασία μπορέσει να είναι έτοιμη σε λιγότερο από τέσσερις μήνες από τη στιγμή που η Κομισιόν κατέθεσε την πρόταση. Νομίζω ότι αυτή η ταχεία λήψη αποφάσεων ε, μέσα σε μια τέτοια κρίση δίνει ε, τη δυνατότητα να είναι ε, επίκαιρη η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή που χρειάζεται απόλυτα η Ορδανία. Να ευχαριστήσω λοιπόν την εισηγήτρια και το Κοινοβούλιο για την αφοσίωσή τους. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία η εισηγήτρια, κυρία Ρεζιμέντη. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι για τις παρεμβάσεις σας και ιδίω ε, αφορά το συνάδελφο γιατρό γιατί και εγώ είμαι γιατρός. Ε, είναι πολύ σημαντικός αυτός ο φάκελος ε, και πρέπει να αναλυθεί πέρα από αυτά που μας χωρίζουν τις πολιτικές ομάδες και ε, χαίρομαι που στην Επιτροπή ΙΝΤΕ είχαμε ομόφωνη ψηφοφορία. Θέλω να υπογραμμίσω ότι η αναγκαιότητα μιας θετικής ψηφοφορίας στο φάκελο αυτό θα πρέπει να υποστηριχτεί απόλυτα το Κοινοβούλιο και να εκφραστεί κατά συνείδηση. Επίσης θα πρέπει να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα των κρατών μας. Γι' αυτό εύχομαι να έχουμε υπερψήφιση του φακέλου αυτού. Αξίζει αυτόνομα να αξιολογηθεί αφήνοντας κατά μέρους κάποιες προκαταλήψεις και δυναμικές ε, ομάδων ε, που συχνά πλήττουν ε, τη δική μου ομάδα και μάλιστα αβάσιμα. Ευχαριστώ. Με την τελευταία αυτή παρέμβαση κλείνει η συζήτηση για αυτό το θέμα. Αύριο θα γίνει η ψηφοφορία. Φτάνουμε λοιπόν στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, της αγορεύσης διάρκειας ενός λεπτού. Κυρία Μπόσκορ έχει το λόγο πρώτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το τελευταία χρόνια στην Ουκρανία έχουν ε, τεθεί μεγάλοι περιορισμοί στα γλωσσικά δικαιώματα των μειονοτήτων. Είναι ο, ο νόμος για την εκπαίδευση και το άρθρο 7, το οποίο έπρεπε να αναθεωρηθεί σύμφωνα με την σύσταση της Επιτροπής της Βενετίας, ε, που ε, δεν έχει αναθεωρηθεί που ε, στην ουσία ε, δημιουργούν το πρόβλημα. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διάταξη στο νόμο η οποία πρέπει να καταργηθεί γιατί ενέχει διακρίσεις. Οι νομοθέτες λοιπόν στην Ουκρανία θα έπρεπε να θεσπίζουν νόμους ε, για τις μειονότητες ε, με την εμπλοκή των μειονοτήτων. Αυτό έχει γίνει και στο παρελθόν. Θα πρέπει λοιπόν να αναβληθεί η χρήση αυτού του νόμου μέχρι να γίνει η έγκριση του νέου νόμου. Ελπίζω η Ουκρανία να κατανοήσει ότι πρέπει να γίνονται σεβαστές οι διεθνείς συνθήκες και τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο για το γεγονός ότι έμεινε εδώ ε, για τόσο χρόνο και παρακολούθησε την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κύριος ε, Τσιουχοντάρου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε θα ήθελα να πω ότι έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το σύστημα Σέγγεν. Το σύστημα Σέγγεν ε, μας βοηθά στη διαχείριση των συνόρων και η Ρωμανία πληρεί τα κριτήρια αυτά. Θα ήθελα να ζητήσω να ακολουθηθούν χωρίς χρονοτριβή ε, οι συστάσεις του Κοινοβουλίου. Να ενταχθεί λοιπόν η Ρουμανία στη Σέγγεν. Το είχε πει και ο κύριος Μπούζεκ και ξέρετε πότε το είχε πει ότι έπρεπε να μπει στις 8 Ιουνίου του 2011. Σχεδόν 10 χρόνια έχουν περάσει και γι' αυτό εγώ θα πρέπει να επιστρέψω στην πρατηρίδα μου και να πω στους Ρουμάνους ότι σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μια ακόμη φορά ζήτησα από το Συμβούλιο και την Κομισιόν να ξαναμπούμε Σέγγεν. Πληρούμε όλα τα κριτήρια και ελπίζουμε αυτό να γίνει το γρηγορότερο, γιατί και οι Ρουμάνοι έχουν δικαίωμα να είναι σε αυτόν τον ευρωπαϊκό χώρο, καθώ εμεί τιμούμε και σεβόμαστε τι ευρωπαϊκέ αξίε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπένιαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στις 15 Νοεμβρίου Υπήρξαν και μαστηρίες κατά του τριπλασιασμού των ποινών του φυσικού αερίου στο Ιράν και διαδόθηκαν ταχύτατα. Το καθεστώς ε, προτίμησε την καταστολή και εμπόδισε, παγόρευσε τις ε, κινητοποιήσεις στις 17 Νοέμβρη για να σταματήσει την επέκταση των φαινομένων. Ε, σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Αμνηστίας, 300 άτομα και πάνω έχουν χάσει τη ζωή τους και υπάρχουν εκτιμήσεις από άλλους οργανισμούς που ανεβάζουν το φόρο αίματος στους 1.500. Και μάλιστα υπάρχουν στοιχεία ότι υπάρχουν ε, γυναίκες και παιδιά ανάμεσα στα θύματα. Χιλιάδες έχουν ε, συλληφθεί. Καλούμε την διεθνή κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταδικάσει αυτή την καταστολή και να ζητήσει την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων. Γιατί πρόκειται και για μια κατάφορη ε, παραβίαση των δικαιωμάτων όσων έχουν συλληφθεί. Πρέπει και το Ιράν να δεχθεί την ε, ελευθερία έκφρασης ε, και πολιτικής δράσης. Ευχαριστώ. Κύριο Σέμιστρο Νίκο. Yeah. Ε, e Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε βαθιά κρίση, το ίδιο και εγώ. Έχω παρακολουθήσει αυτή την παράσταση τους τελευταίους μήνες και δεν διασκεδάζω. Δεν φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη δέσμευση και γενικά δεν υπάρχει καλό περιεχόμενο. Να σας ε, δώσω άμεσο feedback. Καταρχάς, ε, το σενάριο δεν βγάζει νόημα. Το ένα επεισόδιο έλεγε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπέρ της ειρήνης και μετά ε, δεν σταματάμε παρά όταν φτιάξουμε στρατό. Επίσης, οι διάφοροι ήρωες. Ε, ε, δεν τους γνωρίζω. Επίσης, χάνεται το μήνυμα. Θα έπρεπε να πάρουμε μαθήματα από τη Eurovision. Θα πρέπει να δίνουμε προσοχή στον κόσμο για να αρχίσει να χορεύει. Επίσης, αν τα πράγματα δεν ε, βελτιωθούν, θα σταματήσουν να έρχονται οι θεατές. Πρέπει στους θεατές μας να δείξουμε κάτι ε, καλό. Αυτό είναι το show του Νίκο Ζέμστροκτ. Είμαι ο Νίκο Ζέμστροκτ από τους Πράσινους. Ευχαριστώ. Να σας πω να, ότι θα πρέπει να βγάζετε το καπέλο σας όταν είστε εδώ μέσα στο μέλλον. Αυτό δεν ε, συνάδει με τους κανόνες ε, του Κοινοβουλίου. Η κυρία Περμπακάς έχει το λόγο τώρα. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι επιστρέφει ένα σκάνδαλο που έπληξε την υγεία εκατομμυρίων Ευρωπαίων ε, με την υπόθεση κλορτεκών. Το άρθρο 168 της Συνθήκης της Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, υποστηρίζει ότι πρέπει να προστατεύουμε την ανθρώπινη υγεία. Εμεί ζητάμε ως βουλευτέ από το Ευρωπαϊκή Εδάφη να δοθεί μια βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί οι συμπατριώτε μου στις αντίλες έχουν ε, υποστεί άμεσες ε, ή παρά πλευρε συνέπειε. Η παραπλευρε συνεπειε η χρηση του κλορντερκών είναι υπεύθυνη για πολυάριθμα πλευρήματα υγεία ε, και ήταν γνωστά οι συνέπειε αυτέ στη γαλλική κυβέρνηση που όμω συνέχισε να διατηρεί τη χρήση του ε, από το 68 στο 1973. Η υγεία κάθε Ευρωπαίου θα πρέπει να είναι ένας κοινό στόχος ε, και γι' αυτό ε, θα πρέπει να δώσουμε αποζημίωση στα θύματα. Ευχαριστώ κύριο Στέρτς. Yeah, buenas, Καλησπέρα σας ε, και ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Τζόνσον και τον Βρετανικό λαό για την ε, καταπληκτική εκλογή τους νίκη με το συντηρητικό κόμμα ε, το οποίο είχαμε την ε, τιμή εδώ να συμμετέχουμε με κοινού στην ομάδα ECR. Λυπάμαι που θα αποχωρήσουν γιατί πιστεύω ότι χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο τους Βρετανούς για τη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως τους συγχαίρω επειδή συνεχίζουν να υπερασπίζουν αυτό που θα θεωρούν ότι είναι δίκαιο και δεν εκφοβίζονται. Οι βρετανικές εκλογές για μας είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνουν μια εξέταση της συνείδησή τους, κάτι που δεν έκανα στις 23 Ιουνίου 2016. Τότε ε, ξεκίνησε μια περίοδος, έπρεπε να ξεκινήσει μια περίοδος προβληματισμού για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως αντίθετα ε, απέρριψε την απόφαση των Βρετανών. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη μεγάλη ευκαιρία να αποφύγει να ακολουθήσουν το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες που αισθάνονται όλο και χειρότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κόβεται το μικρόφωνο του μιλητή. Ε, πρέπει να δούμε ότι επιστρέφει πιο αυστηρή Με συγχωρείτε, αλλά κόβετε το μικρόφωνο του μιλητή. Οι διερμηνείς δεν ακούνε. Ε, είναι θέμα δικαιοσύνη να μείνετε πιστοί στο χρόνο σα. Επόμενη η κυρία Κόνετσνα. Πρόεδρε, Επίτροπε. Η βιομηχανία Χάλιβα επανελειμμένω έχει μιλήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Λέγοντα ότι υπάρχει κρίση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αντιστραφεί αυτή η τάση, όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Οι εταιρείε ε, κόβουν την παραγωγή, απολύουν ε, εργαζομένους και εξετάζουν και το ενδεχόμενο να κλείσουν. Η Αρσελόρ Μιτάλ σταμάτησε την παραγωγή στην Κρακοβία και έτσι είχαμε 1.300 απολύσεις. Η Chatham Steel ε, ανακοίνωσε μέτρα που θα κοστίσουν 3.000 ε, θέσεις εργασίας. Σε άλλη εταιρεία 2.500 απολύσεις στη Σλοβακία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι προωθεί την οικολογική χαλιβουργία, όμως ταυτόχρονα δημιουργούν ποσοστώσεις για ε, το κακό εντό αγωγικών ατσάλι από τρίτε χώρε. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθήσει, λοιπόν. Ευχαριστώ, κύριο Τσβέρ. Κύριε Πρόεδρε, ένα θέμα που αναφέρθηκε με μεγάλη ανησυχία από τους ευρωβουλευτές τις τελευταίες εβδομάδες είναι η ε, πολύ κακή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν μετά τις ε, ε, διαμαρτυρίες που ξεκίνησαν στις 15 Νοεμβρίου και έχουν περάσει σε τουλάχιστον 200 πόλεις. Υπάρχουν δολοφονίες, σκοτομοί και παρόλο που λέει το, η, κυβέρνηση ότι έχουν μειωθεί ο αριθμός. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους και πολλοί που έχουν συλληφθεί. Ε, πάνω από 500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τουλάχιστον ε, οι περισσότεροι από αυτούς ήταν γυναίκες και μικρά παιδιά. Κοιτάξτε τη νύχτα. Αυτή η εικόνα δείχνει ε, το κορίτσι αυτό 14 ετών. Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη να στείλουν μια ε, αποστολή εξέβρεσης δεδομένων στην περιοχή το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καρθία Ντελπλάνκο έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Εκτιμάται ότι 400.000 δεκάτομα ζουν στο δρόμο στην Ευρώπη και μάλιστα δεν είναι κάτι εφήμερο. Θεωρείται ότι στη χώρα μου περίπου το 50% βρίσκεται πάνω από τρία χρόνια σε αυτήν την κατάσταση. Το είναι κανεί άστεγο ε, σκοτώνει. Είναι πάρα πολύ ευπαθεί οι άνθρωποι αυτοί και μάλιστα πλήττει και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ηθαγένεια ε, στην Ευρώπη. Το βλέπουμε ε, μάλιστα ε, θέλετε και στις ίδιες τις πόρτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Αυτό θα πρέπει να μας κάνει να νιώθουμε ντροπή. Έχουμε την υποχρέωση να αντιδράσουμε απέναντι σε αυτήν την κατάσταση, όχι μόνο επειδή το λέει το θεματολόγιο του 2030 ή ο κοινωνικός πυλώνας, αλλά γιατί έχουμε εργαλεία στη διάθεσή μας. Χώρες όπως η Φιλανδία μας δίνει δείχνουν ότι έχουμε πιο αποτελεσματικού τρόπους να δράσουμε. Μπορούμε να δράσουμε απευθεία ε, και να στείλουμε συστάσεις ε, στα κράτη-μέλη που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Μπορούμε και πρέπει να δράσουμε. Thank you, Frau Ευχαριστώ, κυρία Μπρόφι Τζέιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ίσως αυτή να είναι η τελευταία μου ευκαιρία να μιλήσω εδώ εκ μερου της ε, Βορειοδυτικής Αγγλίας. Είμαι η σωστή. Δεν είδα το όνομά μου. Μπορώ να ξαναξεκινήσω. Ναι, μπορείτε να ξαναξεκινήσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ίσως να είναι η τελευταία μου ευκαιρία να μιλήσω εκ μέρους ε, της ε, Νοτιοδυτική Αγγλίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση που στάθηκε στο πλευρό μας όταν όλοι οι άλλοι μας είχαν εγκαταλείψει. Μας δώσατε ένα δίχτυ ασφαλείας όταν δεν μας το έδωσε κανείς άλλος και τη δυνατότητα και την εξουσία να διαμορφώσουμε τα δικαιώματά μας, μας συνδέσατε με τον κόσμο και μας διευρύνατε τους ορίζοντες. Μας δώσατε νοσοκόμες, γιατρούς, μας δώσατε καθαρό αέρα και θέσατε, μας θέσατε στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων. Και το πιο σημαντικό από όλα, όταν δεν είχαμε καμία ευκαιρία στην περιοχή μας, πιστέψατε σε μας. Είμαστε ευγνώμονες, ξέρουμε το καλό που κάνετε. Οπότε αυτό δεν είναι το τέλος. Ε, εμείς ε, θέλουμε να ζούμε σε μια ανοιχτή χώρα, ανεκτική, που θα συνεργάζεται με τους γειτονές της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ραγίζει η καρδιά μου που φεύγουμε από όλα αυτά. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Φρανσίσκο Γκερέιρο έχει το λόγο. Πρόεδρε, στις 10 Δεκεμβρίου η Ζαμπέλ Λορένσο, ακτιβιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκδιώθηκε από τα κατελημένα εδάφη της Δυτικής Σαχάρας από τις Μαροκινές Αρχές. Η Ζαμπέλ ε, είναι Πορτογαλίδα υπήκος ε, και πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις για να είναι στη χώρα. Είχε όλα τα απαραίτητα έγγραφα, διαβατήριο και είχε και εισιτήριο επιστροφή για τις Πάλμας. Ε, αυτό που ήθελε να κάνει είναι να γνωρίσει την κατάσταση των πολιτικών ε, κρατουμένων. Η Λαζαμπέλ Λορένσο θεωρήθηκε ω ε, persona non grata και ε, θεωρήθηκε ότι παρεβαίνει στην εθνική κυριαρχία του Μαρόκου. Της κατάσχεσαν το κινητό και δεν τις επέτρεψαν να κάνει καμία κλίση. Συνεχίζεται δηλαδή η καταστολή του Μαρόκου και στη Δυτική Σαχάρα θα πρέπει να τελειώσει αυτή η κατάσταση και θα πρέπει να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα αυτή. Ευχαριστούμε. Κυρία Κριστίνα Άντερσον έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Τα Χριστούγεννα είναι πρωτών πυλών, η πιο ωραία γιορτή του χρόνου. Γι' αυτό δράτω με τις ευκαιρίες σας να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και υγεία, ευτυχία ε, στο, για το νέο έτος. Αλλά φέτος ε, οι ευχές μου πηγαίνουν κυρίως στους Βρετανούς. Σας ευχαριστώ που μας δείξατε πώς βγαίνουμε από αυτή την ευρωπαϊκή και γραφειοκρατική τυραννία. Και ορίστε, σας εύχομαι ευτυχισμένο Brexit, σας εύχομαι ευτυχισμένο Brexit. Επιτέλους θα είστε ελεύθεροι. Χειροκροτώ τους Βρετανούς. Thank you. Ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος ε, Κάνετ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, το ερώτημα στην ουσία είναι, μπορούμε να έχουμε μια δίκαιη μετάβαση εάν δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Σήμερα υπάρχουν ε, πόλεις στη Βουλγαρία που δεν έχουν ε, νερό. Πάνω από 130.000 ε, πολίτες πρέπει να κάνουν Χριστούγεννα χωρίς πόσιμο νερό. Και μάλιστα φαίνεται ότι το πόσιμο νερό που είναι δικαίωμα κάθε Ευρωπαίου πολίτη στην ουσία χρησιμοποιείται για βιομηχανικούς σκοπούς. Είναι μια κατάφορη αδικία και πολιτική διαφθορά. Ταυτόχρονα έχουμε έναν γενικό εισαγγελέα που ποτέ δεν έφερε αντίθεση και αντίρρηση στα ανώτερα επίπεδα της εξουσίας. Και τώρα βλέπουμε ότι ο ίδιος θα λάβει τη θέση του ε, Υπουργού Καταπολέμησης Διαφθοράς στη Βουλγαρία. Υπάρχουν περιβαλλοντικά προγράμματα εκατομμυρίων, αλλά δεν νομίζω ότι η Βουλγαρική Εισαγγελία θα ε, εγγυηθεί την σωστή δαπάνησή τους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, στη Μούρσια, στην Ισπανία, ε, στην ε, ε, έχουμε μία λιμνοθάλασσα που, όπου στα μέσα Οκτωβρίου ε, εξαφανίστηκαν 3.000 ε, ψάρια. Μάλλον εμφανίστηκαν 3.000 τόνοι ψάρια νεκρά. και είδαμε ότι τελικά δεν ήταν φυσικά τα αίτια, αλλά είναι η εντατική γεωργία, κερδοσκοπία των ε, κυβερνήσεων τα τελευταία 40 χρόνια και τώρα θα πρέπει να ελέγξουμε ε, τα λίματα ε, στη Λιμνοθάλασσα. Ζητώ λοιπόν υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να παρέχει περισσότερες λύσεις που βασίζονται στη φύση για να ερευνηθεί αυτή η συγκεκριμένη υπόθεση και να δοθεί βοήθεια στους αλείς στην περιοχή της Μπούσια στην Ισπανία. Ευχαριστώ. Ε, κύριος Κέλεχερ. Όταν φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι υπόλοιπε ε, χώρες δεν θα έχουν πανεπιστήμια ε, στα καλύτερα 30 του κόσμου. Θα πρέπει λοιπόν μέσα από τον ορίζοντα για την Ευρώπη να ε, διασφαλίσουμε ότι το Συμβούλιο, η Κομισιόν ε, το... και τα κράτη-μέλη επενδύουν στην καινοτομία, στην έρευνα και στην μετάβαση σε μια οικονομία για την οποία μιλάμε συνεχώ στην οικονομία χωρί εκπομπέ αερίου. Αν δεν έχουμε λοιπόν τα πανεπιστήμια, πώ θα ερευνήσουμε προ αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει στην Ευρωζώνη και στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε τέτοιες γνώσεις. Πρέπει να ενισχύσουμε τις επενδύσεις, να ενθαρρύνουμε την γνώση μέσα από τον ορίζοντα και να βρούμε τον τρόπο μέσω των ε, πανεπιστημίων να επενδύουμε ε, σε κολέγια στις διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Αυτό είναι και μέσα στα πλαίσια ε, Τη μελλοντική μα στρατηγική, να σταματήσουμε με το Σύμφωνο σταθερότητα και να πάμε στα πανεπιστήμια. Ευχαριστώ κύριος Κώστας Παπαδάκης, έχει το λόγο. Νόμενα ευχολόγια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καθόλου δεν ανακόπτουν την επιθετικότητα της Τουρκίας, τις παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων γειτονικών κρατών, όπως δείχνει και το αυθαίρετο τουρκολιβικό σύμφωνο αντίθετα το διεξαγόμενο παζάρι για το προσφυγικό η πώληση όπλων της γερμανίας και άλλων κρατών στην τουρκία οι διαβεβαιώσεις περί στρατηγικού εταίρου της ευρωπαϊκής ένωσης την αποθρασύνουν. με δεδομένη την ανάλογη στάση των ηνωμένων πολιτειών του νάτο και του οηε σε ρόλο πόντιου πιλάτου είναι εκτός πραγματικότητας και επικίνδυνος ο καλλιεργούμενος εφησυχασμός από την κυβέρνηση της νέας δημοκρατίας και το σύριζα πολύ δε περισσότερο το κυβερνητικό κλίμα εφορίας οι ευρωατλαντικές μεθοδεύσεις για συνδιαχείριση σε αιγαίο και ανατολική μεσόγειο θα οξύνουν τις αντιθέσεις και θα περιπλέξουν περισσότερο την κατάσταση. τα λαϊκά συμφέροντα είναι σε αντίθεση με αυτά των ομίλων. η απάντηση είναι η ένταση της λαϊκής πάλης κατά των ξένων βάσεων των αστικών τάξεων και των υπερελιστικών ενώσεων για να ζήσουν οι λαοί ειρηνικά με τη δική τους εξουσία με σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα. Η κυρία Σναλεγκλάβακ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να κάνω μια ε, σύντομη επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και στο ρόλο της στη διαμόρφωση της Ευρώπης. Θα συνεχίσω στα ακροατικά. Κύριε η συμφωνία αυτή θα είναι κλειδί για το μέλλον της Ευρώπης και του κόσμου. Βλέπουμε αλλαγές στον κόσμο, βλέπουμε πυρκαγιές, ε, την αύξηση της στάθμης της θάλασσας. Ε, ολόκληρα νησιά φαίνεται ότι θα εξασφανιστούν στο Σπλίτε, στην Κροατία. Έχουμε τα υψηλότερα επίπεδα στη στάθμη της θάλασσας από ό,τι ποτέ. Βρισκόμαστε λοιπόν αντιμέτωποι με μεγάλες ε, πυρκαγιές, ε, δασικές πυρκαγιές ε, και πλημμύρες. Συνεχώς βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα το τελευταίο διάστημα. Η Κροατία έχει πάνω από χίλια νησιά τα οποία έχουν αποφασίσει να μην χρησιμοποιούν ε, πλαστικά ε, ε, στο χώρο τους, στα σπίτια τους. Αυτό είναι για να ενισχυθεί η οικονομική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος. Όπως είπε και ο Μπάνκι Μουν, είμαστε η μόνη γενιά που θα μπορέσει να κάνει βήματα υπέρ του περιβάλλοντος. Αλλιώς θα υπάρξει πρόβλημα. Οι επόμενες γενιές δεν θα μας συγχωρήσουν ποτέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. στο Παναμά την περασμένη εβδομάδα είχαμε την πρώτη ε, ευρω... Λατινοαμερικάνικη Κοινοβουλευτική Συνέλευση και είχα και την τύχη να μπορέσω να συμπροεδρεύσω στη συνεδρίαση αυτή η οποία είναι τόσο ε, σημαντική τώρα που η περιοχή φαίνεται να βιώνει σημαντικές ταραχές εμείς οι Ευρωπαίοι θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι υποστηρίζουμε τις διμερείς ε, σχέσεις ότι ε, έχουμε μια στρατηγική σχέση που θέλουμε να συνεχίσουμε και τα επόμενα πέντε χρόνια για να δώσουμε και συνταγές να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της περιοχής. Ποιες είναι οι συνταγές, ε, πολέμηση της ανισότητας και θεσμικό πλαίσιο. Πρέπει να έχουμε ισχυρούς ε, θεσμούς που να ακούν τα αιτήματα των πολιτών και ταυτόχρονα η κοινωνική συνοχή να αποτελεί το θεμέλιο της δημοκρατίας μας. Ταυτόχρονα οι βουλευτές και των δύο περιφερειών έστειλαν ένα μήνυμα ισχυρό. Θέλουμε να ξανέχουμε συνόδου κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΛΑΚ και μεταξύ πρωθυπουργών και προέδρων και των δύο περιφερειών. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Πέτερ Πόλακ. Έχει το λόγο. αν ο Χίτλερ είχε κερδίσει τον πόλεμο, δεν θα ήμουν σήμερα εδώ σε αυτό το σώμα. Σήμερα υπάρχουν βουλευτές εδώ που τον θαυμάζουν, όπως και αυτή την θεωρία του για την ανατερότητα. Όμως ε, δεν κοιτούν ε, τι γίνεται και τι κάνουμε, αλλά το δικό τους το μυαλό. Ε, υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στον Παγκόσμιο Πόλεμο στη Σλοβαγία σήμερα ε, υπήρχαν άνθρωποι και βγήκαν στο δρόμο με ε, στολές ε, και δεν τρέπονται να βάζουν το σταυρό του Χριστού και ταυτόχρονα να είναι υπέρ του μίσους. Όμως ο Θεός δεν έχει καμία σχέση με το, μύθο, με το μίσος οι ακρεότητες, ο εξτρεμισμός ε, ανθούν μεταξύ των νέων κυρίως. Πρέπει να μην μείνουμε σιωπηροί μπροστά στην άνοδο του φασισμού. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο φασισμός δεν θα τους ε, αναλώσει, ότι δεν θα είμαστε τα επόμενα θύματα. Ο Βίκας Πινιέρο έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ, Επίτροπε. Πολλές φορές πρέπει να έρθουμε σε αυτή την ολομέλεια για να καταγγείλουμε τη στάση και τις καταχρηστικές πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις από μια low-cost εταιρεία, τη Ryanair. Στην περίπτωση αυτή, είχαμε ε, το εξή γεγονός ε, εμπόδισαν ε, να πετάξει μία νεαρή η οποία έπρεπε να μετακινείται σε μία ηλεκτρική, σε ένα ηλεκτρικό καροτσάκι. Η Ryanair θεωρήσε ότι δεν είχε δικαίωμα να πετάξει, ότι δεν είχε δικαίωμα να πάει με το αναπηρικό της καροτσάκι και την άφησε ουσιαστικά στο έδαφος ε, γιατί ε, δεν μπορούσε να κινηθεί η κυρία αυτή χωρίς ε, το καροτσάκι. Πόσα λοιπόν ακόμη θα πρέπει να συμβούν, πόσο ακόμη θα πρέπει να παραβιάζει η Ryanair το Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο και πόσο θα πρέπει ουσιαστικά να παραβιάζει τα δικαιώματα των επιβατών της για να πάρουμε κάποια μέτρα. Σας παρακαλώ, παρακαλώ να ενδιαφερθείτε για να είναι αυτή η τελευταία περίπτωση. Ευχαριστώ, κυρία Σουζάνα Σικάρτη. Σε όλη την Ευρώπη έχουμε έχουμε το Nutri-Score, μία ετικέτα που ε, ουσιαστικά αξιολογεί ως υγιή προϊόντα αυτά που έχουν λίγη ζάχαρη και λιπαρά και την παρμεζάνα, τη δική μας το προσούτο ε, ή το έξτρα περθένο ελαιόλαδο τα θεωρεί μη υγιεινά προϊόντα. Όμως ε, είναι ένα σύστημα αυτό που μπερδεύει τον καταναλωτή, προσπαθεί να τον καθοδηγήσει και να τον προσανατολίσει σε προϊόντα που τελικά στο σύνολό τους δεν είναι υγιεινά. Οι γιαγιάδες μας ε, χρειαζόταν, ε, χρειάζονταν αυτό το νουτρισκόρι, ή μια ετικέτα με διάφορα χρώματα για να ξέρουν ε, πόσο ελαιόλαδο θα βάλουν στη σούπα. Ήξεραν την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά της μεσογειακής δίαιτας και όλα τα προϊόντα που συνιστούν τη δίαιτα αυτή που είναι made in Italy. Εμείς η μόνη ετικέτα που δεν περισπιζόμαστε πάντα είναι το made in Italy. Σε αντίθεση με του εργατικού και του φιλελευθέρου, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να ε, στρουθοκαμιλίζει σε ό,τι αφορά τι εκλογέ. Γιατί το αποτέλεσμα δεν έχει να κάνει με του ανόητου Βρετανού ψηφοφόρου ή τα μέσα ενημέρωση ή του ε, φασίστε, ε, του αρνητέ κλιματική αλλαγή. Ούτε ο Τραμπ φταίει, ούτε η εξωγήινη σε κάθε βήμα η Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξε να δώσει λιγότερα αντί να δώσει περισσότερα. Το είδαμε σε, σε όλες τις προηγούμενες πρωθυπουργίες. Ε, επέλεξε να κάνει τα πρώτα πιο δύσκολα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα μόνιμο μέλος ε, του Συμβουλίου Ασφαλείας, ένα ιδρυτικό μέλος ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης φεύγει οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πάρουν λιγότερα, ε, η φορολογία θα αυξηθεί, τα πράγματα θα είναι χειρότερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλ, μάλλον το Ηνωμένο Βασίλειο, θέλει να έχει μια πολύ καλή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να προσφέρει λιγότερα. Πρέπει λοιπόν να μάθετε το μάθημά σα από τον Brexit, ότι τα έθνη μα πετυχαίνουν περισσότερα όταν ε, υιοθετούν την ε, θεωρία τη ελεύθερη αγορά. Αν το κάνετε αυτό, τότε και οι Βετανοί θα στηρίξουν μια πιο πράσινη, ασφαλή, πιο πλούσια και ευτυχισμένη Ευρώπη. Να πω, συνάδελφε, ότι η διαδικασία εξόδου έχει τρία μέρη. Υπάρχουν ε, οι μεταβατικές ε, ρυθμίσεις ε, και οι διαπραγματεύσεις για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε αυτό τον τομέα. Και τώρα έρχομαι στην κυρία Ιρένα Γιώβεβα. Αυτή η κρίση στην καρδιά της Ευρώπης πραγματικά δεν ξέρετε γιατί πράγμα μιλάω ακριβώ, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα, πολλές επονίδη στις καταστάσεις ε, ε, που λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα ο Βούτζεκ. Ε, είχαμε στη Βοσνία Ερσεγοβίνη με ένα καταβλισμό προσφύγων και ήταν μια ντροπή. Έκλεισε αυτό γιατί ήταν πήγον όμως αυτό δεν έφερε σε τέλος και σε πέρας την κρίση των προσφύγων. Όχι, χρειαζόμαστε συμφωνία. Μια κοινή συμφωνία για μια κοινή πολιτική μετανάστευσης και ασύλου, η οποία θα επιλύσει πλήρως ε, τα ζητήματα στις χώρες προέλευσης. Γιατί, γιατί αν δεν έχουμε τέτοια συμφωνία, εμείς θα είμαστε τελικά το μεγαλύτερο όνειρο στην καρδιά της Ευρώπης. Ο κύριος Τόμισλαφ Σόκολ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο καρκίνο σήμερα είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα σε ό,τι αφορά τη γνωμική περίθαλψη και στην Ευρώπη και παγκοσμίω. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο, σχεδόν 2 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη ζωή του εξαιτία του καρκίνου και το 40% αυτών των θανάτων θα μπορούσαν να έχουν αποφευθεί αν είχαν εφαρμοστεί τα κατάλληλα μέτρα. Από την άλλη, ξέρουμε ότι η περίθαλψη ε, έγκυται σε αρμοδιότητα των κρατών μελών βάσει του άρθρου 168 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για την Ευρωπαϊκή Ένωση για την μη ανάληψη δράση ό,τι αφορά τον καρκίνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μία σειρά εργαλεία στη διάθεσή τη και οικονομικά και νομοθετικά ε, για την καταπολέμηση του καρκίνου, για συνοριακές υπηρεσίε υγειονομικής περίθαλψης, το πρόγραμμα ορίζων, ε, πολιτική συνοχής που επιτρέπει ε, επενδύσεις σε υποδομές στον τομέα της υγείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει τα εργαλεία στη διάθεσή τη για να καταπολεμήσει τον καρκίνο. Υπάρχει πολιτική βούληση τη Κομισιόν και του Κοινοβουλίου και πιστεύω ότι πραγματικά θα πρέπει να επενδύσουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε τα κατάλληλα αποτελέσματα. Α δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα γραφειοκρατικό τέρα, αλλά μπορεί πραγματικά να βοηθήσει του ε, πολίτε. Και τέλος, Ευχαριστώ. Ο μηχανισμός συνεργασίας εφαρμόστηκε το 2006 πριν η Ρουμανία και η Βουλγαρία να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο σκοπό αυτού του μηχανισμού είχε σχεδιαστεί ω ένα σύστημα ανάλυσης και ελέγχου του συστήματος δικαιοσύνης Ρουμανία Βουλγαρίας προκειμένου οι δύο αυτέ χώρες όταν θα έχουν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εθετήσουν τέτοια πρότυπα δημοκρατίας και κράτους δικαίου με τις υπόλοιπε ευρωπαϊκές χώρες. Όμως στην περίπτωση της Ρουμανίας βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια αυτό ο μηχανισμό συνεργασία και ελέγχου ε, μεταμορφώθηκε σε πολιτικό μηχανισμό, ενώ ήταν τεχνικός. Και αυτή η έκθεση περιλαμβάνει μια σειρά λαθών και δημιουργήσε και μια αρνητική αντίδραση από τους δικαστές της ε, Ρουμανίας. Έχουμε ποιοτικά, ποσοτικά λάθη να υπάρχουν στην έκθεση αυτή. Η τελευταία έκθεση, σχέση με τη Ρουμανία, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, αρνείται ε, κάποια πράγματα που προβλέπονται από το Σύνταγμα της Ρουμανίας. Καλό την Κομισιόν να αξιολογήσει εκ νέου τον τρόπο που γίνεται η αξιολόγηση του δικαστικού συστήματος της Ρουμανίας και να ξαναγράψει την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Τελείωσε και αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Αύριο το πρωί, Τρίτη, στις 9 η ώρα το πρωί θα συνεχιστεί η συνεδρίαση. Θα δείτε και στο ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις αντίστοιχες πληροφορίες. Ε, με αυτό κλείνουμε τη σημερινή συνεδρίαση.